Possiamo allora cominciare i nostri e Ας ξεκινήσουμε την ε, συνεδρίασή μας. Ο συνήθως να θυμίσω ότι η συνεδρίαση θα μεταδοθεί μέσω διαδικτύου και θα βιντεοσκοπηθεί. Είναι μια ανακοίνωση που πρέπει να την ε, κάνω πάντοτε, αλλά σήμερα έχει και ουσιαστική αξία, γιατί βλέπω λίγους βουλευτές μας εδώ στην αίθουσα. Όμως, οι εμπειρογνώμονες δεν θα πρέπει να αποθαρρυνθούν και άλλοι μπορεί να προσέλθουν Για βεβαίως όσοι απουσιάζουν θα μπορούσαν να ακούσουν ή να δουν αυτά που θα μας παρουσιάσετε, γιατί όλα δεν σκοπούνται ήθελα να κάνω και μια ανακοίνωση προς τους συναδέλφους που είναι εδώ παρόντες. Ένα ζήτημα που έθεσαν χθε οι συνάδελφοι Νταφ και Γκουαλτιέρη. Υποστήριξαν ότι δεν ίσχυε η τελική ψηφοφορία για το θέμα της τσεχικής δημοκρατίας. Επί της ουσίας, ήδη χθε το βράδυ έγιναν κάποιες παρατηρήσεις ορθές και επειδή υπήρχαν διαδικαστικές ε, αμφιβολίες Μα απασχόλησε το κατά πόσο έπρεπε το θέμα αυτό να τεθεί μετά την λήξη τη ψηφοφορία, προ το τέλο τη συνεδρίαση, ή να έπρεπε να τεθεί αμέσω μετά την ψηφοφορία. Οι υπεύθυνοι τη Ολομελία μου είπαν ότι παρόλο που το θέμα δεν τέθηκε εγκαίρω, και νομίζω και εγώ, όπω μου είπα και εκείνη, ότι μπορούμε να ακολουθήσουμε ένα δρόμο που θα μπορούσαμε να το χρησιμοποιήσουμε και ως προηγούμενο και για τη δική μας και για άλλες επιτροπές. Επειδή η αλήθεια είναι διαφορετική, η πραγματικότητα δηλαδή ήταν εσφαλμένη, μπορούμε να μεταβάλουμε την απόφασή μας. Πρέπει νομίζω να κηρύξω και θα γραφτεί και στα πρακτικά ότι η τελική ψηφοφορία ακυρώνεται. Δεν ισχύει. Θα πρέπει να την επαναλάβουμε. Μόνο την τελική ψηφοφορία. Η ψηφοφορία αυτή θα πρέπει να γίνει στην επόμενη συνεδρίαση, όπου θα προβλεφθούν ε, ψηφοφορίες. Καλώς εγέρθηκε λοιπόν το θέμα, γιατί ήταν πρωτοφανές να ψηφίσουμε με ηλεκτρονικό σύστημα, όπου οι ψήφοι δεν αντιστοιχούν σε ονόματα. Και λόγω των ε, συναδέλφων που δεν είχαν τις κάρτες μαζί τους και ψήφισαν σηκώνοντα το χέρι, τελικά παραποιήθηκε το αποτέλεσμα. Έγινε λάθος ε, με το συνολικό αποτέλεσμα. Δεν ξέρουμε λοιπόν ε, πώς ψήφισε ο καθένας χωριστά, επειδή η ψηφοφορία ήταν ηλεκτρονική, οπότε καλό είναι να ακυρωθεί και να ξαναψηφίσουμε. Περνάμε τώρα και στο βασικό μας θέμα για σήμερα τίτλο «Μέθοδος άμεσης συμμετοχή των πολιτών στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρότυπο για μια πιο δημοκρατική Ευρώπη». Το θέμα είναι σημαντικό, διότι εδώ και πολύ καιρό μιλάμε για το δημοκρατικό έλλειμμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση ένα ζήτημα στο οποίο προσπάθησε να προτείνει λύσεις η όλη διαδικασία της συνθήκης της Λισαβόνας. Ωστόσο ακόμη η πορεία μας δεν έχει εξασφαλίσει την πλήρη κάλυψη των πολιτών από δημοκρατικής σκοπιάς. Η δημοκρατία και το έλλειμμά της στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι κατά πρώτον διαρθρωτικού χαρακτήρα. Πρέπει να βελτιώσουμε στο δυνατόν περισσότερο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων και τον τρόπο που προβάλλονται προς τον λαό. Υπάρχει βέβαια και μια συναισθηματική ψυχολογική διάσταση εδώ είναι σημαντικό ο ευρωπαϊκός λαός να αισθάνεται λαός και μάλιστα ευρωπαϊκός. Αλλιώ απομακρύνεται από την Ευρώπη. Υπάρχουν κάποιοι μηχανισμοί που οφείλουμε να μελετήσουμε. Ακόμα και από την άποψη των μέσων που χρησιμοποιούμε, διότι Το τι θέλει θέλουν οι πολίτε τη Ευρώπη μπορεί να μην φαίνεται μεγάλη σημασία αρχικά, αλλά έχει σημασία για τη συνείδηση που διαμορφώνεται στο νου για το πώ ε, μπορούν να αισθάνονται πολίτε τη Ευρώπη. Η συμμετοχική δημοκρατία λοιπόν καθιερώνεται από τη συνθήκη της Λισαβόνας με τις ε, πρωτοβουλίες των πολιτών. Οι εγγυήσει λοιπόν που δίδονται είναι ήδη ένα πρώτο Η Επιτροπή αυτή έχει μελετήσει δύο κανονισμούς, κυρίως τον 211 για την υλοποίηση και επιμακρών έχει εξετάσει το θέμα αυτό. Σε αυτή τη φάση οι πρωτοβουλίε των πολιτών, νομίζω, όπω καταγράφονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, έχουν φτάσει τι 10 και για αυτές Ήδη έχει κινηθεί η διαδικασία λήψης αποφάσεων. Υπάρχουν βεβαίως κάποιες δυσκολίες, όπως η χρήση του ηλεκτρονικού συστήματος, όπου απαιτούνται και ιδιαίτερες εγγύησεις για τη συλλογή υπογραφών και εγγύησεις ασφάλειας Αυτή ήταν μια σύντομη εισαγωγή στο θέμα. Προφανώς δεν είναι μόνο οι πρωτοβουλίες των πολιτών αυτές που θα αυξήσουν την ε, αίσθηση της δημοκρατίας στην Ευρώπη. Πρέπει να είμαστε εφάνταστοι εδώ, να επινοήσουμε και άλλα συστήματα και να το συζητήσουμε. Δεν μπορούμε να συγκρίνουμε τη συμμετοχική δημοκρατία μιας μικρής κοινότητας, τη συμμετοχή δημοκρατία, μιας μικρής κοινότητας, σκέφτομαι την αρχαία Ελλάδα, την αρχαία αγορά, όπου όλοι οι πολίτε συζητούσαν και ψήφιζαν, δεν μπορούμε να συγκρίνουμε ένα τέτοιο σύστημα με την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπου έχουμε σχεδόν μισό δι ε, πολιτών που αποτελούν ένα κοινό λαό. Χρειάζεται λοιπόν εδώ ιδιαίτερη φαντασία. Όπως λέει και το Γερμανικό Συνταγματικό Δικαστήριο, πρέπει να δούμε πώς θα διαμορφωθεί ο Ευρωπαϊκός Δήμος ο ευρωπαϊκός λαός. Δεν θέλουμε να είναι απλώς ένα άθροισμα πολιτών, αλλά ένας λαός με κοινή συνείδηση. Γι' αυτό λοιπόν σήμερα θα ακούσουμε τους ειδικού μας, τον κύριο Γέργες, τον κύριο Κάουφμαν, τον καθηγητά Σίλερ, τον καθηγητή Κίρς Γκέσνερ, τον ε, κύριο Λίμπερτ, τον κύριο Γκρός και την κυρία Μπράουν Μπίντερ για καθέναν από τους εμπειρογνώμονες έχουμε και ένα τίτλο παρουσίασης. Μπορούμε κάθε φορά να ακούμε δύο λοιπόν από τους ειδικού μας. Θα τους αποδίδουμε 11 λεπτά για την παρουσίαση αυτή και μετά από τις δύο παρουσιάσεις μπορούμε να κάνουμε διάλογο με, την, ε, με τα μέλη της Επιτροπής. Εδώ να χαιρετήσω θερμά και να ευχαριστήσω για την παρουσία του τον κύριο Χέφνερ Εκείνος ε, σχεδίασε την ε, συνάντηση αυτή και συνεισέφερε τα μάλα στην επεξεργασία του κανονισμού 211 που προανέφερα. Νομίζω καλό θα ήταν να τον ακούσουμε και εκείνον. Κύριε Χέφνερ. Ja, herzlichen Dank. Ευχαριστώ. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Καζίνη και να καλωσορίσω και εγώ τους ειδικού μας, τους συμμετέχοντες, τους προσκεκλημένους στην ακρόαση. Θεωρώ πως ε, είναι ιδιαίτερη η στιγμή αν και βεβαίως θα θέλαμε κάπως ε, μεγαλύτερη συμμετοχή των βουλευτών αλλά να εξηγήσω στους καλεσμένους μας πως είναι πολύ πολύ άσχολη η σημερινή μέρα. Υπάρχουν πολλές συνεδριάσεις που διεξάγονται παράλληλα και κάποιοι συνάδελφοι άρα δεν μπορούν να έρθουν. Εμείς θέλουμε να ασχοληθούμε με το θέμα της συμμετοχής των πολιτών, της δημοκρατίας και της άμεσης δημοκρατίας στα κράτη-μέλη και στο επίπεδο της Ένωσης. Εγώ έχω την εντύπωση πως το θέμα αυτό γίνεται κάθε μέρα πιο σημαντικό σε μια υπερεθνική κοινότητα κρατών όπου είναι κάτι το ενδιάμεσο μεταξύ Ομοσπονδίας και Ομοσπονδιακού κράτους το ζήτημα είναι πώς θα υπάρξει μια δημοκρατική νομοποίηση μέσα των πολιτών. Εάν δεν το καταφέρουμε αυτό, τότε οι πολίτες θα έχουν την εντύπωση πως τα δικαιώματα της κυριαρχίας ε, που πηγαίνουν πάνω από το σύνηθες επίπεδο του κράτους ε, πηγαίνει χέρι-χέρι με την απώλεια δικαιωμάτων. Οπότε ε, ο εξευρωπαϊσμός της λήψης αποφάσεων θα σημάνει και το τέλος της δημοκρατίας και της συμμετοχής των πολιτών. Αυτό δεν επιτρέπεται. Θέλουμε μια δημοκρατική ένωση, όπως αναφέρεται και στην χάρτα των θεμελιωδών δικαιωμάτων και στις συνθήκες, αλλά νομίζω πως δεν έχουμε ακόμα επαρκείς απαντήσεις στο ερώτημα του πώς ορίζουμε τη δημοκρατία πέρα από το εθνικό κράτος. Και αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο είναι αποφασιστικό για το μέλλον της Ευρώπης. Εγώ είμαι πεπισμένος πως η Ευρώπη μόνο τότε θα επιτύχει όταν κερδίσουμε δηλαδή και τα μυαλά και τις καρδιές των ανθρώπων όταν θα είναι μια Ευρώπη δημοκρατική όταν οι πολίτες θα έχουν την εντύπωση πως μπορούν να εμπλακούν άμεσα στην ευρωπαϊκή πολιτική, στη λήψη αποφάσεων και πως μετράει ο λόγος τους και πώς μπορούν να επηρεάσουν τις αποφάσεις. Εάν συμβεί το αντίθετο, εάν υπάρχει εντύπωση πως πηγαίνουμε προς μία τεχνοκρατική μορφή λήψης αποφάσεων και είναι μόνο θεατές οι πολίτες και δεν ξέρουν πώς μπορούν να εμπλακούν, τότε θα απομακρυνθούν από την Ευρώπη και αυτό βεβαίως πρέπει να το εμποδίσουμε, αλλά είπα πως το θέμα αυτό αφορά και κάτι πέρα από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Για το πώς δηλαδή θα μπορέσουμε να οργανώσουμε τη δημοκρατία πέρα από το κράτος έθνος. Πώς όλα αυτά τα όργανα, τα θεσμικά, τα υπερεθνικά, τα διεθνή τα οποία εξ ανάγκης ε, αποκτούν όλο και περισσότερες αρμοδιότητες, πώς θα μπορέσουμε να διασφαλίσουμε πώς θα υπάρχει μια επιρροή των πολιτών σε αυτά. Αυτό είναι λοιπόν το μεγάλο ζήτημα και ταυτόχρονα παρατηρούμε στην Ευρώπη συγκλονιστικές εξελίξεις. Εάν δούμε τις τελευταίες δύο δεκαετίες τις εξελίξεις ε, στην λήψη αποφάσεων διαπιστώνουμε πως στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στα κράτη-μέλη σε επίπεδο Δήμου, Περιφέρειας, κράτους μέλους υπάρχει μια τεράστια διάδοση νέων μορφών λήψης αποφάσεων και συμμετοχής του λαού. Οπότε και ο κόσμος ζητάει περισσότερη συμμετοχή και έχουμε νέες μορφές συμμετοχής. Και με τη μορφή της διαβούλευσης, αλλά και πολύ περισσότερες νέες διαδικασίες ε, άμεσης δημοκρατίας. Αν σκεφτώ παραδείγματος χάρη ε, τα μεγάλα παραδείγματα στη Γερμανία, από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο μέχρι το 1990 είχαμε λίγες αποφάσεις οι οποίες ε, λήφθησαν σε τοπικό ή περιφερειακό επίπεδο από τους πολίτες. Και στα 21 χρόνια από το 1990 μέχρι το 2011 υπήρχαν χιλιάδες τέτοιες αποφάσεις οι οποίες ε, λήφθησαν με αυτόν τον τρόπο. Οπότε χρησιμοποιήθηκαν πολύ περισσότερο αυτές οι δυνατότητες αποφάσεων και αυτά τα οποία έλεγε ο κόσμος, ε, αυτά τα οποία υπήρχαν ως φόβοι ε, απέναντι σε αυτές τις μορφές συμμετοχής ότι θα ήταν παράλογες οι αποφάσεις, ότι δεν υπάρχει λογική συζήτηση, πώς θα επικρατήσει ο λαϊκισμός ή παραδείγματος χάρη όταν αφορούσαν τα οικονομικά υπήρχε ξεκάθαρη η ανησυχία πως ε, δεν θα μπορούσαν να κρίνουν σωστά για τους φόρους, τα έξοδα και ότι θα χρεοκοπούσε το κράτος. Γιατί θα σκέφτονταν μόνο τις δαπάνες και όχι ότι πρέπει να έχει έσοδα το κράτος. Αλλά κάναμε εμπειρικές έρευνες και αποδεικνύουν ακριβώς το αντίθετο. Εκεί όπου συμμετέχουν οι πολίτες στις αποφάσεις ε, για τους φόρους, ε, εκεί πέρα, λοιπόν, ακριβώς, διαπιστώνουμε πως οι πολίτες χρησιμοποιούν πιο αποτελεσματικά, πιο υπεύθυνα το χρήμα. Οι χώρες αυτές είναι πολύ λιγότερο χρεωμένες από άλλες όπου δεν συμμετέχει ο λαός στη λήψη αποφάσεων. Οπότε η συμμετοχή των πολιτών δεν βοηθάει μόνο στο να εκμηρωθεί η σχετική επιθυμία και να υπάρξει και στήριξη κτλ. Αλλά σε πολλούς τομείς μας δίνει και νέες ιδέες και με δυνατότητες δηλαδή συζητιούνται τα πράγματα δημοσίως και μπορεί ο κόσμος να συμμετέχει αυτή είναι μια διαφορά της συμμετοχικής δημοκρατίας σε σχέση με την αντιπροσωπευτική δημοκρατία που δεν θέμε να αμφισβητήσουμε αλλά αποτελεί τη βάση της δουλειάς μας στο Κοινοβούλιο. Αλλά στην αντιπροσωπευτική δημοκρατία ανακατεύονται πάρα πολλά ζητήματα ταυτόχρονα και βεβαίως είναι και το ζήτημα των προσώπων. Ενώ στη συμμετοχική δημοκρατία, στην άμεση δημοκρατία, υπάρχει πάντα ένα συγκεκριμένο ερώτημα για το οποίο αναζητούνται λύσεις. Και όπως είπα, οι εμπειρικές έρευνες, η πείρα δείχνει πως δεν υπάρχει μόνο ενίσχυση της νομοποίησης, αλλά και ουσιαστικά καλύτερες αποφάσεις. Σήμερα λοιπόν έχουμε προσκαλέσει ειδικού Jahrzehnten beschäftigen und που ασχολούνται με το θέμα αυτό δεκαετίες και θέλουμε να μάθουμε από αυτούς ποια μέσα, ποιες διαδικασίες υπάρχουν, ποιες εμπειρίες υπάρχουν, θετικές και αρνητικές. Θέλουμε να μάθουμε τι σημαίνει αυτό για την Ευρωπαϊκή Ένωση, τι μέσα και διαδικασίες θα μπορούσαν να υπάρχουν στο επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή ποιους, ποιες νέες διαδικασίες θα μπορούσαμε να αναπτύξουμε έτσι ώστε να έχουμε από τώρα μεγαλύτερη συμμετοχή των πολιτών. Αυτό αναμένουμε από τους ειδικού και θα ακούσουμε τώρα σε δύο γύρους των δύο μιλητών τους ειδικού μας και μετά θα έχουμε βεβαίως και χρόνο για ερωτήσεις και βέβαια θα έχουμε και πολύ περισσότερο χρόνο το απόγευμα γι' αυτό θα ακούσουμε εκεί πέρα τρεις ομιλητές για να υπάρχει πάλι αρκετός χρόνος για να μιλήσουν αλλά και να απαντήσουν ερωτήσεις από τα μέλη της Επιτροπής και τους λοιπούς. Ο Πρόεδρος. Η... Είπε να ξεκινήσουμε αμέσως και εγώ λέω να δώσουμε αμέσως τον λόγο στον καθηγητή Κριστιαν Γεωργής από το Πανεπιστήμιο της Βρέμης. Έχετε το λόγο. Vielen Dank, Herr Hefner. Grazie, Presidente, per l'invito. Ευχαριστώ κύριε Χέφνερ και σας ευχαριστώ και εσάς κύριε Καζίνη για την πρόσκληση. Είναι μεγάλη τιμή για μένα. Αλλά θα μιλήσω στην ε, γλώσσα την πιο, αν θέλετε, απλή και ξεκάθαρη τα αγγλικά. Για να βοηθήσω την επικοινωνία. Ελπίζοντας ότι η άμεση συμμετοχή του ακροατηρίου θα είναι πιο δυνατή με τα αγγλικά και ελπίζω και να μιλώ αρκετά καλά τα αγγλικά ώστε να το πετύχω αυτό. Πάνω απ' όλα και υπό τις, παρόντες, υπό τις παρούσες συνθήκες είναι ε, πάρα πολύ σημαντικό για την Ευρωπαϊκή Ένωση να μιλήσουμε εδώ για το πώς θα μπορέσουμε να ενδυναμώσουμε την ε, συμμετοχή δημοκρατία σε όλα τα επίπεδα. Και η δική μου παρέμβαση σίγουρα ε, θα είναι μάλλον αρκετά ε, θεωρητική διότι μας είπαν ε, ότι θα πρέπει να έρθουμε εδώ και να σας δώσουμε κάποιες εξηγήσεις και πρακτικές λύσεις. Αλλά αληθεύει επίσης το ότι βρισκόμαστε σε μια εποχή που γίνεται ένας πολύ σημαντικός διάλογος για το μέλλον της δημοκρατίας στην Ευρώπη και υπάρχουν και κάποιες διελκυστίνδε μεταξύ αφενός ε, τη τεχνοκρατικής διαχείρισης της κρίσης ε, και από την άλλη πλευρά ε, το αίτημα, η διεκδίκηση για περισσότερη δημοκρατία. Αυτό θα είναι και το επίκεντρο τη δική μου μικρής παρέμβαση. Θα ξεκινήσω με μία εξέταση της βιβλιογραφίας όπως κάθε καλός δικηγόρος και έπειτα θα περάσω σε κάποιες πρόσφατες προτάσεις οι οποίε τέθηκαν για την επινόηση μια νέα μορφής δημοκρατίας. Η μία πρώτα στη διατύπωση μία πρώτα στη διατύπωση μια ομάδα συλλαδέλφων στη Φλωρεντία, ενώ την άλλη ε, ο πολίς Γιούργεν Χάμπερμας, μεταξύ άλλων. Αφού σα πω όλα αυτά, στη συνέχεια θα σα μεταφέρω τι δικέ μου απόψει και τα δικά μου οράματα για την περισσότερη δημοκρατία στην Ευρώπη. Πρώτα απ' όλα, τι λέει η συνθήκη για την, δημοκρατική, για την συμμετοχική δημοκρατία. Πιστεύω ότι τα γνωρίζετε όλοι πολύ καλά, διότι την έννοια αυτή ε, πρώτα απ' όλα την εμπνεύστηκε η Ευρωπαϊκή Συνέλευση και η συνθήκη τη Λισαβόνα πρόσθεση, μάλλον διατήρησε την έννοια αυτή τη συμμετοχικής δημοκρατία που δεν έρχεται σε αντίφαση ως έννοια με την αντιπροσωπευτική δημοκρατία, αλλά τη συμπληρώνει. Πρόκειται παρόλα αυτά για ένα ουσιώδες, θεμελιώδες ζήτημα και όπως ε, όλα τα σημαντικά ζητήματα της ευρωπαϊκής πολιτικής σχολίασε και το Συνταγματικό Δικαστήριο της Γερμανίας, φαντάζομαι γνωρίζετε, αλλά σε μια απόφασή του για την ε, συνθήκη της Λισαβόνας στο Συνταγματικό Δικαστήριο λέει ότι δεν υπάρχει όργανο λήψης πολιτικών αποφάσεων ε, το οποίο προέρχεται μετά από εκλογές. Η νέα αρχή τη συμμετοχή δημοκρατία και οι μηχανισμοί τη δεν επαρκούν κατά το Συνταγματικό Δικαστήριο τη Γερμανία για να αντισταθμίσουν την έλλειψη τη αντιπροσωπευτική δημοκρατία. Γνωρίζουμε ότι το γερμανικό δικαστήριο συνήθως ε, ε, λειτουργεί με επιχειρήματα ναι ή όχι ή ναι αλλά ε, την ίδια ακριβώς στρατηγική χρησιμοποιεί και η απόφαση για την ε, Λισαβόνα λέει ότι ναι, μεν η διαβουλευτική συμμετοχή των πολιτών και των ε, κοινωνικών του οργανώσεων ε, στην ε, πολιτική διακυβέρνηση δεν μπορεί να αντικαταστήσει την νομιμοποιητική σχέση που βασίζεται στι εκλογέ και άλλε προφορίε. Ωστόσο, αυτά τα στοιχεία τη συμμετοχική δημοκρατία μπορούν να συμπληρώσουν την νομιμοποίηση τη Ευρωπαϊκή Δημόσια Αρχή και η αποκεντρωμένη συμμετοχή μπορεί να καταστήσει πιο αποτελεσματική αυτή την πρωταρχική, αντιπροσωπευτική και δημοκρατική σύνδεση της νομιμοποίησης. Υπάρχουν κάποιες... Ε, ε, Υπάρχουν αυτές οι δύο έννοιες λοιπόν της αντιπροσωπευτικής και της συμμετοχική δημοκρατίας ε, που δεν είναι δύο διαφορετικές εναλλακτικέ, ούτε είναι και αντιφατικές έννοιες. Δεν θέλω να επισέλθω σε θεωρατική συζήτηση ε, θέλω να στραφώ στις δύο υποδείξεις, στις δύο προτάσεις που σας προανέφερα για την ενίσχυση της δημοκρατίας στην Ένωση, τις οποίες πρόσφατα κατέθεσαν ε, διακεκριμένοι συνάδελφοι στο τραπέζι. Οι δύο αυτές από φαινομενικά απέχουν πόρο μεταξύ τους, αλλά ε, στην πραγματικότητα ουσιαστικά έχουν ως υπόβαθρο και οι δύο την αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης ε, και ανταποκρίνονται αυτής της εντάσεις που υπάρχουν μεταξύ της δημοκρατικής ε, δέσμευσης αφενός και της διαχείρισης κρίσης αφετέρου. Ποια είναι η βασική ιδέα. Πρώτα απ' όλα, εκδημοκρατισμός μέσω κοινοβουλευτικής συμμετοχής για την εκλογή του Προέδρου συγκεκριμένα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Και αυτό βέβαια αφορά άμεσα αυτό το θεσμικό όργανο. Πρώτα απ' όλα ο Μιγέλ Ποϊάρης Μαδούρο που ήταν ε, ε, εισηγητής δικαστής ε, στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και επίσης από τον Ματία Κούμ. Ο Μπαρόζο έχει οθετήσει την ιδέα αυτή και την έχει περασπιστεί. Δύο στοιχεία της όλης συλλογιστικής θα ήθελα να σας μεταφέρω. Πρώτα απ' όλα, Υπάρχουν, κάποιες δομικοί, κάποιοι δομικοί περιορισμοί για την αυτόνομη δημοκρατική λήψη αποφάσεων. Έχουμε λήψη αποφάσεων σε πολλού τομεί. Ατομική ενέργεια, φορολογική, δημοσιονομική πολιτική και όλα αυτά επηρεάζουν, έχουν εξωτερικές επιπτώσεις ε, αν λαμβάνονται σε ένα κράτο μέλο και στα άλλα κράτη-μέλη. Αποφάσει που λαμβάνονται σε ένα κράτο μέλο όμω, δεν λαμβάνουν υπόψη ούτε και υποτίθεται θα έπρεπε να λαμβάνει υπόψη τα συμφέροντα των ε, γειτονικών χωρών. Είναι ένα επιχείρημα λογικό, ε, αλλά αυτό που δεν είναι τόσο εύκολα κατανοηθεί είναι, και έτσι λένε η Μαδούρο και Κουμ, ότι υπάρχουν τελικά αυτές οι εξωτερικές επιπτάσεις, άρα θα πρέπει να υπάρχει μια εξωτερική υπερεθνική αρχή για την αντιστάθμιση αυτών των επιπτώσεων. Αυτή η υπερεθνική αρχή λοιπόν που βλέπουμε να αναδύεται σήμερα ε, και που έχει να κάνει με τη διαχείριση της κρίσης. Ε, πώς γίνεται αυτή η διαχείριση της κρίσης από τα κράτη-μέλη της κυβερνήσεις. Δεν υπάρχει όμως νομιμοποίηση, γιατί δεν υπάρχει αντιπροσώπευση, δεν υπάρχει έκφραση της κοινοβουλευτική δημοκρατίας. Άρα έρχονται οι δύο αυτοί συνάδελφοι, κάνουν ένα επόμενο βήμα προς τα εμπρός και λένε πώς μπορούμε να δημιουργήσουμε μια δομή αντιμετώπισης της κρίσης σε υπερεθνικό επίπεδο που να είναι πιο δημοκρατική. Έτσι λοιπόν έρχεται η αρχή και η ιδέα της άμεσης εκλογής του πρόεδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αυτές οι άμεσες εκλογές θέλουν οι δύο αυτοί συνάδελφοι να οργανώνονται, οι άμεσες εκλογές να διοργανώνονται από δύο ομάδες, δύο κόμματα θέλετε που θα ε, παρουσιάζουν υποψηφίους ε, στην ευρωπαϊκή κοινή γνώμη. Θα παρουσιάσουν τα προγράμματά τους ε, και έτσι θα έχουμε αυτή τη μεγαλύτερη, πιο δημοκρατική διαδικασία. Και έτσι θα προχωρήσει περισσότερο ο εκδημοκρατισμό τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Εγώ έχω προσωπικά κάποιε αμφιβολίε. Κυρίω γιατί δεν μπορώ να καταλάβω πώ αυτό ο ανακλεγή πρόεδρο ε, μπορεί να ενταχθεί σε αυτέ τι δομέ. τις φυστάμενες και πώς αυτός ο νέος πρόεδρος θα μπορούσε να έχει την εξουσία και την αρμοδιότητα ώστε πραγματικά να αποφασίζει για κρίσιμα ζητήματα που μπορεί να στοιχίζουν πολλά χρήματα για κάποιους ε, από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ άλλοι ζητούν αλληλεγγύη ε, καταλαβαίνετε όλα αυτά που ε, τα βιώνουμε και σήμερα, όλες αυτές τις αντιπαραθέσεις. Πιστεύουμε ε, πραγματικά ότι μπορούν να επιληθούν όλα, αυτά ε, με την άμεση εκλογή του Πρόεδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Δεν είμαι τόσο πεπισμένος. Δεύτερη τώρα πρόταση. Πρόταση του Γιούργεν Χάμπερ μας. Ίσως να την ακούσατε ή να τη διαβάσατε στην Frankfurter Allgemeine. Εκεί λοιπόν υπέβαλε ε, αν θέλετε, ένα μανιφέστο. Κάθε εβδομάδα γράφει και από ένα το συγκεκριμένο ήταν ιδιαίτερα ισχυρό υπό την έννοια ότι ασκεί κριτική ο Χάμπερ μας στην πολιτική διαδικασία που παρατηρούμε σήμερα. Ενώ την άλλη πλευρά υπογραμμίζει πόσο σημαντική έχει γίνει η Ευρώπη. Κατά την άποψη του Χάμπερ μας λοιπόν η Ευρώπη είναι η μόνη ευκαιρία που έχουν οι Ευρωπαίοι για να αντιμετωπίσουν τα προβλήματά τους. Τι προτείνει λοιπόν ο Χάμπερ μας. Πρώτα απ' όλα παρουσιάζει μια ιδέα την Ευρώπη που είναι κοντά ε, στις αγωγές παρατηρήσεις που ακούσαμε, δηλαδή ότι η Ευρώπη δεν είναι ούτε ομοσπονδία ούτε και απλή ε, ένωση κρατών. Έχει οικοδομηθεί ουσιαστικά από ή απαρτίζεται από πολίτες που ανήκουν στο εθνικό ε, πολίτευμα, στην εθνική πολιτεία, αλλά είναι και Ευρωπαίοι πολίτες από την άλλη πλευρά. Αυτή η σχέση λοιπόν εθνικού-ευρωπαϊκού Ο Χάμπερ μα δεν λέει ότι θα πρέπει να υπάρξει μια Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία. Μπορεί να συνδυαστεί το εθνικό και το ευρωπαϊκό επίπεδο με διαφορετικού τρόπου. Πιστεύω ότι πρέπει, παραδείγματο χάρη, να υπάρξει ίσω μια νέα συνέλευση, μια νέα convention και ίσω και δημοψηφίσματα για να ενισχυθεί η συμμετοχή των Ευρωπαίων. Ήταν βέβαια πάντοτε κάπως ανεδαφικός, κάπως ουτοπικός, αλλά αυτό είναι και το μεγάλο του προσόν. Αυτή λοιπόν είναι η πρόταση του Χάμπερ μας. Δεν ξέρω πώς μπορεί να υλοποιηθεί όσο σοβεί αυτή η κρίση. Και δεν μπορώ επίσης να καταλάβω πώς αυτές οι διάφορες πρωτοβουλίες και πολιτικές ε, αρθρώσεις των πολιτικών δήμων θα μπορούσαν να ε, οδηγήσουν σε επιχειρησιακές λειτουργικές προτάσεις. Ο στόχο δεν είναι να δημιουργηθεί ε, μια, ένα νέο πολιτικό πρόγραμμα, αλλά είναι, αν θέλετε, η ε, μεγαλύτερη συμμετοχή στα κοινά, ε, στα πολιτικά δρόμενα των Ευρωπαίων πολιτών. Έχουμε να συζητήσουμε βέβαια τα υπέρ και τα κατά. Το θέμα είναι τι θα γίνει με τη μεταφορά εξουσίας και αρμοδιοτήτων από το ευρωπαϊκό στο εθνικό, από το εθνικό στο, ευρω, στο ευρωπαϊκό επίπεδο. Υπάρχουν πρακτικές δυσκολίες Εμένα πάντως με ενθουσιάζει η ιδέα η ευρωπαϊκή όλη αυτή διαδικασία να πάρει νέα ορμή, νέα όθηση με δημοψηφίσματα από άλλους λαούς, όχι μόνο από τους Δανούς ή από τους ε, Ολλανδούς, για παράδειγμα, να γίνει ευρύτερη όλη αυτή η διαδικασία και να οδηγήσει τελικά σε μια ανευρωπαϊκή συνέλευση. Βέβαια δεν μπορεί να γίνουν αύριο αυτά όλα τα πράγματα, αλλά τι κάνουμε μέχρι αύριο τι κάνουμε στο μεταξύ. Και εδώ έρχομαι και εγώ λοιπόν για να σας δώσω κάποιες δικές μου υποδείξεις και αυτές πολύπλοκες είναι, αλλά τουλάχιστον ε, να δείτε κι εσείς ε, ποιες είναι οι δικές μου ιδέες, πώς θα ήθελα εγώ να οικοδομηθεί αν οικοδομηθεί και συλληφθεί ενοιολογικά η νέα αυτή Ευρωπαϊκή Ένωση. Συνταγματική συνθήκη ενότητα πολυμορφία. Δηλαδή, μπορούμε να δημιουργήσουμε μια ευρωπαϊκή πολιτεία όχι με την ομοιογένεια. Γιατί έχουμε όλα αυτά τα θέματα ρυθμιστική πολιτική κτλ. Α, όχι λοιπόν με την ομοιογενειοποίηση, ε, αλλά με άλλου τρόπου, του οποίου θα σα περιγράψω. Συνεργασία και συμμετοχή των πολιτών. Θα προσπαθήσω να σας δώσω δύο θεωρητικές αρχές, δύο αξιώματα να περιγράψω και μετά θα σας ε, μεταφέρω κάποιες πρόχειρες σκέψεις για το πώς αυτά μπορούν να ελοπιθούν στην πράξη. Όπως προτείνουν Μαντούρο και Κουμ, πιστεύω ότι το ευρωπαϊκό δίκαιο έχει ε, νομιμοποίηση γιατί ουσιαστικά αναπληρώνει τις ανεπάρκειες των εθνικών δημοκρατιών. Η βασική υπόθεση είναι ότι έχουμε καταφέρει ε, να δημιουργήσουμε κάποιες αλληλεξαρτήσεις στην Ευρώπη, όπου τα εθνικά κράτη δεν μπορούν πλέον να επιλύσουν αυτόνομα τα προβλήματά τους. Διότι οι αποφάσεις που λαμβάνουν επηρεάζουν τους γείτονές τους και δεν είναι νομιμοποιημένες αυτές οι επιπτώσεις από αυτού που επηρεάζονται από τι αποφάσει αποφάσεις αυτές. Άρα υπάρχει ένα πρόβλημα εδώ νομιμοποίηση και θα πρέπει το κενό, το έλλειμμα που δημιουργείται να το καλύψει το ευρωπαϊκό δίκαιο. Το ευρωπαϊκό δίκαιο έχει αναπτύξει κάποιες τεχνικές για να επιβάλλει καθήκοντα και υποχρεώσει στα κράτη-μέλη, ώστε να λαμβάνουν υπόψη τις ανησυχίε των διαφόρων ε, άλλων κρατών, όπως υπόθεση Κασίστη Ντιζό και άλλες υποθέσεις του δικαστηρίου. Τώρα όμως ε, έχουμε μία επιτακτική ανάγκη, διότι δεν μπορούν επικοδομητικά σε εθνικό επίπεδο να επιληθούν τα προβλήματα τουλάχιστον αποτελεσματικά και επαρκώς. Δεν υπάρχει επίσης η δυνατότητα ε, να δημιουργηθεί και ένα πολιτικά αντιπροσωπευτικό σώμα σε ευρωπαϊκό επίπεδο που θα μπορούσε να το πράξει. Επομένως, χρειάζεται, και αυτή είναι η θέση μου, μία συνταγματοποιημένη, μία θεσμοθετημένη, αν θέλετε, συνεργασία. of the Europe. Πρέπει λοιπόν να δώσουμε δυνατότητα στους πολίτες να συμμετέχουν περισσότερο. πρέπει να έχουμε υπόψη μα ότι υπάρχει πολυμορφία στην Ευρώπη και υπάρχει σχετική αυτονομία επίση των κρατών μέλων. Άρα θα συνεχίσουν να προκύπτουν σημεία τριβή και τομεί διαφωνία. Δεν υπάρχει λοιπόν μέχρι στιγμή μια αρχή η οποία να έχει την αποκλειστική και έσχατη απότατη εξουσία για να λάβει μια τελική απόφαση. Στα σχόλιά μου για την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία, την Πρωτοβουλία των Ευρωπαίων Πολιτών, θεωρώ ότι είναι αξιοθαύμαστη αυτή η πρωτοβουλία, διότι ακριβώς ε, επιτρέπει τη διοργάνωση πολιτικών διαδικασιών μεταξύ αυτών των ευρωπαϊκών πολιτιών και συγχρόνως δημιουργεί διαδικασίες λήψης αποφάσεων βάσει διαδικασιών και συζητήσεων. Δεν έχουμε βέβαια τις εγγυήσεις ότι αυτές οι συζητήσεις θα καταλήξουν σε ένα συμπέρασμα το οποίο θα είναι αποδεκτό από όλους. Αλλά αυτή η λήψη αποφάσεων θα οδηγήσει σε αποφάσεις οι οποίες θα λαμβάνουν υπόψη, πιστεύουμε, ε, τα μελήματα όλων των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, και θα εξορροπούν ε, τις ανησυχίες των διαφόρων κρατών μελών. Ένα βασικό παράδειγμα είναι η ατομική ενέργεια. Το έχω μελετήσει δεν θέλω να επισέλθω βέβαια σε λεπτομέρειε γιατί είναι ιδιαίτερα λεπτό το ζήτημα. Είναι όμω ένα παράδειγμα. Παρ' όλα αυτά μα δείχνει πώ η ε, διαδικασία εθνική λήψη αποφάσεων επηρεάζει τι γειτονικέ χώρε. Ενώ από την άλλη πλευρά δεν υπάρχει Ευρωπαϊκή Αρχή η οποία αναλαμβάνει τελική απόφαση. Παρ' όλα αυτά πρέπει να βρεθεί, να οργανωθεί μια τέτοια πολιτική διαδικασία για να μπορέσουμε να συμβιώσουμε με κάποιο τρόπο ε, υπό προοπτικές και σκοπιές στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Βέβαια το πιο πιεστικό ίσως παράδειγμα είναι η οικονομική κρίση που αντιμετωπίζουμε σήμερα. Τεράστιοι κίνδυνοι. Η διαχείριση της κρίσης σε ευρωπαϊκό επίπεδο δεν ξέρουμε αν θα σώσει το ευρώ ή όχι. Αυτό που μπορούμε όμως να δούμε ήδη από τώρα είναι ότι υπάρχει αυτή η τάση διοργάνωσης της διαχείρισης της κρίσης μέσω μιας ενός μηχανισμού ε, υπερεθνικού ε, για τη διαχείριση της κρίσης. Αυτό απειλεί όμως τη δημοκρατία και το λέει και ο Χάμπερ μας στο μανιφέστο του. Εγώ είμαι Γερμανός δικηγόρος, άρα ε, δεν μπορώ παρά να αναφέρω για μια ακόμη φορά την απόφαση προηγούμενης εβδομάδας του Γερμανικού Σταγματικού Δικαστηρίου Όλοι ε, ανακουφίστηκαν, ε, η Ευρωπαϊκή Κοινωνία, η ε, Γερμανία και η κυβέρνηση και ούτω καθεξής. Βέβαια δεν παρεμβαίνει στην διαχείριση της κρίσης. Προσπαθεί να διατηρήσει και τις νοστομικές εξουσίες της Bundestag η απόφαση του δικαστηρίου σε ένα σημαντικό τμήμα της απόφασής του, το Συνταγματικό Δικαστήριο λέει ότι με την έγκριση της βοήθειας για τη σταθεροποίηση Bundestag ασκεί την επιρροή που ζητά το Σύνταγμα και συμμετέχει στις αποφάσεις σε ό,τι αφορά την ερεσιμότητα του ποσού και την διάρκεια της παροχής της βοήθειας. Καθορίζει δηλαδή τους βασικότερους όρους για την εκταμείευση κεφαλαίου. Ως Γερμανός πολίτης τα χρήματα τα οποία διαχειρίζεται η Bundestag, εγώ πραγματικά νιώθω ανακουφισμένο. Διότι λαμβάνονται υπόψη τα δημοκρατικά μου δικαιώματα. Ω πολίτη τη Ένωση, που είναι το άλλο μου μισό βέβαια, δεν είμαι και απόλυτα σίγουρο τι γίνεται με τη δημοκρατία για την υπόλοιπη Ένωση. Γιατί η δημοσιονομική αυτονομία δεν εννοείται ω ε, κοινή ευρωπαϊκή συνταγματική κληρονομιά. Γιατί δεν μπορεί να ζητήσει η γερμανική Bundestag από τα άλλα κρατημέλη, από άλλου πολιτικού φορεί τη Ένωση, να τηρήσουν κάποια αιτήματα λιτότητας που προέρχονται από τη Γερμανία από αλλού. Δημοσιονομική ε, κρίση λύνεται μόνο με τη λιτότητα. Δεν ξέρουμε. Σε μια προηγούμενη παράγραφο, το Σταματικό Δικαστήριο βέβαια διανοίγει μια πιο επικοδομητική προοπτική απομακρύνεται από το eternity clause τη βασικής νομοθεσίας και λέει ότι αυτή η ρήτρα δεν έχει ως στόχο να προστατεύσει μόνο συγκεκριμένα στοιχεία του γερμανικού συντάγματος, αλλά έχει ως στόχο να προστατεύσει ουσιαστικά τις δημοκρατικές διαδικασίες και τη δημοκρατική λήψη αποφάσεων και να παραμείνουν ανοιχτές οι δημοκρατικές διαδικασίες στην Ευρώπη. Αυτή είναι μια πολύ πιο επικοδομητική ιδέα που είναι πολύ πιο κοντά στα ιδανικά τα οποία εμπνέουν την πρωτοβουλία των πολιτών. Αυτό το είδου το επιχείρημα φαίνεται να προτείνει ότι η επίλυση των συγκρούσεων μεταξύ τη άσκηση των δημοσιονομικών εξουσιών δεν μπορεί να λυθεί με ε, την υπαγόρευση ε, αρχών και οδηγιών από μια υπερεθνική αρχή, αλλά μόνο με τη διοργάνωση πολιτικών διαδικασιών. Βέβαια, δεν έχω απάντηση ε, με αυτή τη σύντομη ομιλία που εκφώνησα για το πώ μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τη δημοσιονομική κρίση. Αυτό που μπορώ όμω να υπεγραμμίσω για μια ακόμη φορά είναι ποια είναι η απειλή σήμερα για τη δημοκρατία. Δηλαδή, στην Ευρώπη σήμερα η απειλή είναι ότι λαμβάνονται αφενός οι αποφάσεις Λαμβάνονται αποφάσει, δεν τι λαμβάνουμε εμεί. Λαμβάνονται από ένα τεχνοκρατικό σύστημα, από ένα τεχνοκρατικό μηχανισμό που προσπαθεί να επιβάλλει πειθαρχία στην Ένωση. Που δεν νομιμοποιείται δημοκρατικά σε καμία περίπτωση όμω. Και αυτή η ιδέα, άλλε ιδέες για το συνδυασμό της λιτότητα με κάποιου όρου. είναι και αυτό άκρο αντιδημοκρατικό. Εγώ λοιπόν τι λέω μόνο. Αν δεχθούμε ότι η Ευρώπη είναι κοινωνικο-οικονομικά πλουραλιστική, αλλά παρόλα αυτά πρέπει να λαμβάνει συνεργατικά και συλλογικά αποφάσεις, θα χρειαστεί η διαδικασία λήψη αποφάσεων να θεσμοθετηθεί και να συνταγματοποιηθεί, λαμβάνοντας υπόψη και τι ανησυχίε των κρατών μελών, αλλά σεβόμενοι και τι ανησυχίε των πολιτών που επηρεάζονται από αυτές τις αποφάσεις. Και εκεί πραγματικά εγώ βλέπω πολλούς τρόπους για να ξεκινήσουν όλες αυτές οι διαδικασίες και να ανοίξουν ε, στη συμμετοχή. Ε, να σταματήσω εγώ καλύτερα, γιατί νομίζω ότι εξάντλησα το χρόνο μου και ήμουν και αρκετά θεωρητικός και αόριστος, αλλά τι να κάνουμε. Yes, thank you very much, uh, Professor I would like... Σας ευχαριστούμε, καθηγητά Γιώργες. Να ζητήσω τώρα από τον κύριο Κάφμαν να έρθει και εκείνος, αν θέλει, στο Προεδρείο. Είναι πρόεδρος της πρωτοβουλίας ε, του Ιδρύματος Μαλλών ε, της Ευρώπης για τις πρωτοβουλίες και τα δημοψηφίσματα. Επίσης είναι υπεύθυνο εκλογικής περιφέρειας στη Σουηδία και ταυτόχρονα είναι και ερευνητής αλλά και ακτιβιστής. Thank you very much. Uh, thank you very much. Σας ευχαριστώ Γκερχάρτ, ευχαριστώ κύριε Κασίνη, ευχαριστώ ολόκληρη την Επιτροπή που οργανώνει αυτήν την ιδιαίτερη επίκαιρη ακρόαση. δεν είναι απλώς επίκαιρη, διότι είναι οξύτατη η κρίση σε ό,τι αφορά την νομιμοποίηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των θεσμικών της οργάνων, αλλά βρισκόμαστε στην καμπή μιας ολόκληρης πορείας εξέλιξης, μιας αλλαγής προς τον εκδημοκρατισμό της Ευρωπαϊκής Δημοκρατίας. Θέλω λοιπόν το θέμα αυτό να το βλέπω όσο το δυνατόν ευρύτερα. Γι' αυτό ξεκίνησα με ένα παγκόσμιο χάρτη. Βλέπουμε εκεί ότι η Ευρώπη είναι στο παγκόσμιο προσκήνιο. Ακόμη θεωρείται παράδειγμα από όλο τον υπόλοιπο κόσμο ως ε, παράδειγμα της ε, διακρατικής, της υπερεθνικής δημοκρατίας για πολλά χρόνια, για δεκαετίες, οργανώνονται τέτοιες ε, ε, Θυμάμαι το 92 στο Στρασβούργο, λόγου χάρη, όπου είχα παρουσιαστεί για να μιλήσω για μια διακρατική δημοκρατία. Και τότε ένας συνάδελφος από τις κάτω με γελιοποίησε και μου είπε ότι αυτά είναι ανοησίες. Η υπερεθνική δημοκρατία είναι κάτι το ανέφικτο. Σήμερα βεβαίως το συζητούμε πλέον και μάλιστα πολύ περισσότερο. Αυτά που συμβαίνουν τώρα δεν σημαίνουν ότι πρέπει να εγκαθιδρύσουμε την υπερεθνική δημοκρατία. Προσπαθούμε, απόπειρε κάνουμε. Προσπαθούμε να εξεύρουμε ποιοι είναι οι καλύτεροι τρόποι να υλοποιηθεί αυτό. Αν κοιτάξετε σήμερα το αρχείο τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τι Πρωτοβουλίε των Ευρωπαίων Πολιτών, που είναι πολύ καλό φτιαγμένο, θα δείτε ότι υπάρχουν ήδη 10 τέτοιε πρωτοβουλίε. Έχουν ήδη καταγραφεί. Την περασμένη εβδομάδα δημοσιεύτηκαν και μπορείτε ηλεκτρονικώς να υπογράψετε μια από αυτές τις πρωτοβουλίες, να την υποστηρίξετε. Αυτό είναι πολύ πιο σημαντικό από ό,τι πολλοί μπορεί να σκεφτούμε. Είναι η πρώτη φορά στα χρονικά που μια τέτοια πρωτοβουλία μπορεί να υπογραφεί ηλεκτρονικώς. Όχι μόνο στην Ελβετία, στην Ιταλία, στις ΗΠΑ. Σήμερα υπάρχουν δυνατότητες ηλεκτρονικής υπογραφής. Ακόμη και αν είναι λοιπόν δύσκολος ο δρόμος, εάν υπάρχουν πολλά εμπόδια, θα μπορούμε να δοκιμάσουμε. Και ήδη έχουμε μπει στη σωστή πορεία. Έχουμε εκκινήσει την όλη διαδικασία. Ζούμε τις πρώτες εμπειρίες της ε, υπερεθνικής δημοκρατίας και έχουμε ορίσει και κάποιες βασικές αρχές. Είναι σημαντικό να έχουμε λοιπόν μια αντίληψη της ε, ε, δημοκρατίας αυτής που έχει θεμελιωθεί και στις συνθήκες της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως τη Λισαβόνα, τα άρθρα 10 και 11. Κατανοούμε ότι η σύγχρονη δημοκρατία θα πρέπει να βασίζεται και στην συμμετοχή των πολιτών. Επιπλέον, έχουμε ορίσει και συμφωνήσει και συγκεκριμένες διαδικασίες. Οι πρωτοβουλίες των Ευρωπαίων πολιτών είναι διαδικασία, τύπος διαδικασίας που εγκρίθηκε από με ευρύτατη μάλλον πλειοψηφία στο Ευρωκοινοβούλιο. Έχει συμφωνηθεί μάλιστα από όλα τα κράτη-μέλη. Εδώ λοιπόν δεν μιλούμε μόνο για αρχή, αλλά μιλούμε και για διαδικασίες. Στην πράξη θέλουμε βεβαίω να δούμε τώρα τι μπορεί να γίνει και η όλη διαδικασία, η όλη έρευνα είναι συναρπαστική. Αυτό ξεπερνά τα όρια μιας απλής συζήτησης για το είδος συμμετοχής και την άμεση δημοκρατία. Έχουμε φτάσει πια σε ένα σημείο όπου δεν συζητιέται αν θα πρέπει να υπάρχει περισσότερη συμμετοχή ή συμμετοχική δημοκρατία, αλλά πώς θα διοργανωθεί, πώς μπορεί να τεθεί σε εφαρμογή. Μια σύγχρονη δημοκρατία θα πρέπει να βασίζεται σε αυτές τις αρχές που είναι η συμμετοχή και η άμεση δημοκρατία και αυτά είναι τα κύρια χαρακτηριστικά τη σύγχρονη της σύγχρονης ε, αντιπροσωπευτικής δημοκρατίας. Θα πρέπει να βασιστούμε σε, τρεις, ε, σε τρία καθοριστικά στοιχεία. Την, ε, το κράτο δικαίου, την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, αυτό το συμφωνούμε όλοι, το εγκρίνουμε όλοι, και την ιδέα ότι η σύγχρονη συμμετοχική δημοκρατία θα έχει και κάποιες ε, διαδικασίες εξουσιοδότησης δεν είναι δυνατόν όλοι οι άνθρωποι να ε, συνέρχονται σε συνέλευση για να ε, λαμβάνουν αποφάσεις. Πρέπει να υπάρχει και η αρχή της εξουσιοδότησης μέσω των ευρωεκλογών. Αυτό φαίνεται πολλές φορές να έχει οδηγήσει σε παρανοήσεις, παρόλο που υπάρχει ευρεία συνένεση. Ε, φαίνεται σαν να υπάρχει αντίφαση μεταξύ της συμμετοχικής δημοκρατίας και της εξουσιοδότησης. Αυτό είναι σφαλμένο αποδεικνύεται ότι πουδήποτε υπάρχει αυτή η μορφή συμμετοχής στην δημοκρατία, αυτό συμβαδίζει πάντοτε με την προστασία του κράτου δικαίου και την εκπροσώπηση, την εξουσιοδότηση δηλαδή. Είναι δύσκολο βεβαίως να θεμελιωθεί ένα τέτοιο σύστημα, διότι κάποιες φορές ε, αμφισβητεί κάποια μονοπόλια εξουσιών που ήδη λειτουργούν και πρέπει και εκείνοι να καταλάβουν ότι του συμφέρει να μοιραστούν λίγοι από την εξουσία που διαθέτουν και έχουν συγκεντρώσει για να ενισχύσουν τη δημοκρατία. Είναι πολύ ενδιαφέρον να σκεφτούμε ότι το πλαίσιο που δημιουργείται για την διακρατική δημοκρατία πρέπει να θεμελιωθεί πέραν των πρωτοβουλειών των πολιτών, των πολιτών και της ε, ε συνθήκης της Λισαβόνας να γίνει και σε επίπεδο εθνικών κρατών. Ήδη από το 1973 είχαμε 53 δημοψηφίσματα σε ευρωπαϊκά κράτη. Ήδη εδώ και δεκαετίε δημορφώθηκε η έννοια του Ευρωπαίου πολίτη και της ευρωπαϊκής ιθαγένειας. Θα έχουμε και τα γενέθλια, την επέτειο της γένεσης της έννοιας αυτής σύντομα. Έχουμε πλέον τη διαδικασία των Ευρωπαίων πολιτών. Υπάρχουν όμως ε, σοβαρές προκλήσεις εδώ για να υπάρξουν εδώ αποτελέσματα ε, χειροπιαστά. Ήμουν στην Ιρλανδία το Μάιο για να δω πώς θα πάνε οι εκλογές και είδα ότι πολλοί Ιρλανδοί, ιδίω ε, όσοι έχουν την εξουσία, δεν χαίρονται που πρέπει να ψηφίζουν κάθε φορά για ευρωπαϊκά δικαιώματα. Αυτό βασίζεται στην ιδέα ότι πρέπει οι πολίτε να μην είναι μέσα στα πράγματα, να μην γνωρίζουν πώ λαμβάνονται οι αποφάσει. Αυτό συμβαίνει και με τη διαδικασία των Ευρωπαίων πολιτών. Οι περισσότεροι πολίτε στην Ευρώπη δεν γνωρίζουν τα δικαιώματά του, δεν γνωρίζουν τι δέκα πρωτοβουλίε ήδη υπάρχουν και δημοσιεύονται και μπορούν να τι υπογράψουν. Δεν ξέρουν πώ να υπογράψουν δεν ξέρουν ότι τα κράτη-μέλη και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μπορούν να προτείνουν νέα νομοθεσία προ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Είναι λοιπόν θέμα ενημέρωση. Επίση, μια άλλη σοβαρή πρόκληση είναι το ποιοι άνθρωποι θα ενημερώνουν του πολίτε, ποιοι θα απαντούν στα ερωτήματά του. Οι άνθρωποι αυτοί, όσοι εμπλέκονται στην όλη διαδικασία, καθημερινά δέχονται πολλά ερωτήματα από όλη την Ευρώπη. Πώ θα γίνει αυτό, Πώ μπορεί να ξεκινήσουν οι πρωτοβουλίε των Ευρωπαίων πολιτών, Πώ υλοποιείται, Δεν υπάρχει υπάρχει δημόσια χρηματοδότηση για να ε, έχουμε εκπαίδευση για τους πολίτες, μια επίσημη διαδικασία υπεύθυνη ενημέρωση ανά την Ευρώπη δηλαδή. Υπάρχουν για την ώρα κάποιε δειλέ απόπειρε, αλλά όχι αρκετοί πόροι. Επίση, άλλη σοβαρή πρόκληση είναι η στήριξη όσων θέλουν να ασκήσουν τα δικαιώματά του. Κάποιε φορέ ε, συνηθίζω να λέω ότι αγωνιζόμαστε για να δούμε πώ μπορούμε να αλλάξουμε τι υποδομέ μα, την να μεταβάλουμε τη διάρθρωση των δημοκρατικών μα δικαιωμάτων. Όμω ήδη τα δημοκρατικά δικαιώματα που έχουν δεν ασκούνται πλήρω. Δεν τα αξιοποιούμε καθημερινά στην πράξη όπω θα μπορούσαμε. Αυτό βεβαίω που θα μπορούσαμε να κάνουμε είναι να έχουμε υποδομέ ε, που να επιτρέπουν στους Ευρωπαίους πολίτε να λάβουν γνώση όλων αυτών των στοιχείων και να γίνουν πραγματικά Ευρωπαίοι πολίτε. Έχουμε τόσο ωραία κτίρια με ωραίε αίθουσε όπω το Ευρωκοινοβούλιο, που είναι καθοριστικό παράγοντα τη οικοδόμηση τέτοιων υποδομών, αλλά δεν τα γνωρίζουν οι Ευρωπαίοι πολίτε. Οι Ευρωπαίοι πολίτε δεν το νιώθουν σαν δικό του ε, θεσμικό όργανο. Αυτό είναι πραγματική πρόκληση. Δεν είναι μόνο λοιπόν εφικτό να δημιουργηθεί μια τέτοια παιδεία, μια τέτοια νοοτροπία σε όλη την Ευρώπη, σε ευρωπαϊκό επίπεδο δηλαδή, να καλλιεργηθεί, αλλά δεν μπορεί μόνο να ενεργοποιούνται εδώ και όσοι εργάζονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Χρειάζεται και τοπική και περιφερειακή συνιστόσα. Σε περιφερειακή και τοπική συνιστόσα, ε, όπως ε, με τη διακρατική, θα πρέπει να επενδύσουμε. Μερικά βασικά χαρακτηριστικά αυτών των υποδομών θα μπορούσαν να είναι τα εξή. Να έχουμε χώρους χώρου όπου μπορούν οι πολίτε όχι μόνο να συναντώνται αλλά και να ενημερώνονται. Να μπορούν να πάνε εκεί και να ζητήσουν πληροφορίε όχι μόνο μέσω του διαδικτύου, αλλά σε κέντρα δημοκρατίας ανά την Ευρώπη. Σε τέτοιους χώρους, όπως ήδη σε πολλές περιπτώσεις σήμερα διαθέτουμε, θα μπορούσαμε να έχουμε αυτούς που θα ονομάζαμε πλοηγητές, πλοηγούς μάλλον, ε, υπευθύνους που θα ενημερώνουν για τέτοια θέματα. Να τους λένε το πρόβλημά μου είναι αυτό. Και εκείνοι να απαντούν. Είναι ευρωπαϊκή διάσταση, μήπω είναι τοπικό, μήπω είναι κρατικό. Αυτού του είδου η πλογή, ή σύνοδοι, θα πρέπει να ε, εκπαιδευτούν. Και επίση πρέπει να υπάρχει και η ηλεκτρονική μορφή αυτής της εκπαίδευσης να υπάρχουν αιτήσει που να μπορεί κανείς από ένα smartphone να τη στείλει. Να τη στείλει. Εφόσον γνωρίζει κανείς ήδη τα δικαιώματά του, μπορεί να βρεθεί σε κάποιον τόπο να δει μια πόλη όπου έχουν λόγο και οι πολίτες. Πρέπει λοιπόν να υπάρξει πολύ καλύτερη ενημέρωση με πολύ καλύτερες πλατφόρμες και πρέπει να είναι πιο τεκμηριωμένη η συζήτηση για τα δικαιώματα συμμετοχής. Χρειάζονται λοιπόν όλα αυτά τα καθοριστικά στοιχεία. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι οι απόπειρε, οι προσπάθειε είναι πολλαπλέ σήμερα στην Ευρώπη για να υλοποιηθούν όλα αυτά. Ακόμη όμω είναι στα πρώτα του βήματα στο Φαλόν στη Σουηδία προσπαθήσαμε να δημιουργήσουμε μια, όπως ονομάστηκε, δημοκρατική πόλη. Να δημιουργήσουμε κέντρα δημοκρατίας στις δημόσιες βιβλιοθήκες, όχι μόνο για να δανειζόνται δηλαδή βιβλία οι πολίτε στι βιβλιοθήκες αλλά να λειτουργούν και ως κέντρα δημοκρατικής ενημέρωσης για δημόσιες συζητήσει. Υπήρχαν ε, πλοηγοί αυτοί που ονόμασα πλοηγού προηγουμένω, συνοδοί οι οποίοι μπορούσαν να προσφέρουν καθοδήγηση, συμβουλέ, ενημέρωση στου πολίτε, να ε, μάθουν ποια είναι τα δικαιώματά του και πώ μπορεί να τα ασκήσει καλύτερα. Σε πολλέ ευρωπαϊκέ χώρε σήμερα θεωρείται ότι η συμμετοχή πρέπει να υποστηριχθεί, αλλά αυτό συνήθω γίνεται με την έκδοση εγχειριδίων. Εγχειρίδια με θέμα την άσκηση των δικαιωμάτων. Αυτά πάλι στέκονται στην περίπτωση των ήδη εκπαιδευμένων, ήδη ε, ε, ενημερωμένων πολιτών. Και πολλές φορές είναι δύσκολη και η πρόσβαση σε αυτά τα εγχειρίδια. Το κλειδί για όλα αυτά είναι η πρωτοβουλία των Ευρωπαίων πολιτών. Αυτή η διαδικασία. Όχι ότι είναι η μαγική λύση για όλα τα θέματα. Όμως μπορεί να είναι πραγματικά ε, το μαγικό ραβδί που θα συνδυάσει τις διαδικασίες, τα βασικά χαρακτηριστικά την διάσταση αυτή της συμμετοχής που θα είναι πρωτόγνωρη για όλο τον κόσμο. Η άμεση δημοκρατία και η συμμετοχή δεν είναι μόνο ένας τρόπος να αντιστέκεται κανείς και να λέει όχι. Είναι ένας τρόπος να αναπτύσσει κοινέ ιδέες, να επιτρέπει το διάλογο μεταξύ των πολιτών, αλλά και μεταξύ πολιτών και θεσμικών οργάνων. Αυτή η διαδικασία, αυτή η λειτουργία επιτρέπει και πολλά άλλα να, να λάβουν χώρα επιτρέπει τη χρήση των εργαλείων αλλά και πολλά άλλα πράγματα. Αυτή λοιπόν η τόσο σφαιρική διαδικασία, η τόσο σφαιρική υποδομή πρέπει να θεωρηθεί μια πολύ σοβαρή καινοτομία για την Ευρώπη και να αντιμετωπιστεί σαν πρόκληση. Εάν δεν λειτουργήσει, δεν θα αναπτυχθεί η Ευρώπη. Ο κ. Μπαρόζα πρόσφατα είπε ότι ακόμα και εκείνο το παραδέχτηκε, η Ευρώπη χρειάζεται περισσότερη δημοκρατία στην πραγματικότητα. Δεν σημαίνει αυτό ότι θα υπάρξουν ε, πολλαπλέ και ανεξέλεγκτε συνέπειε, όχι. Αλλά το συμπέρασμά μου είναι ότι βρισκόμαστε πραγματικά στα πλαίσια μια συμμετοχική επανάσταση, όχι μόνο στην Ευρώπη, αλλά παγκοσμίω και σήμερα. Οι δημοκρατικέ υποδομέ είναι πολύ περιορισμένε σε ορισμένα θεσμικά όργανα τα οποία έχουν πολύ ισχυρά θεμέλια. Έπειτα, έχω να παρατηρήσω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι πραγματικά μοναδική. Ε, ένα μοναδικό πλαίσιο που να επιτρέπει τον εκδημοκρατισμό των δημοκρατικών μα καθεστώτων. Αυτό επανειλημμένω ακούγεται, διότι λέμε πολύ συχνά ότι υπάρχει έλλειμμα δημοκρατία στην Ευρώπη έλλειμμα της Ευρω... δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά τα δικαιώματα έχουν ένα μοναδικό πλαίσιο παγκοσμίω, ένα πλαίσιο προστασία. Εδώ θα πρέπει να γίνει μια σοβαρή προσπάθεια για την κατανομή τη εξουσία. Εξουσία και συμμετοχή. Το να μιλάμε σήμερα για τη συμμετοχή και την ε, άσκηση δικαιωμάτων συμμετοχή, όλα αυτά σημαίνουν ότι ο στόχο δεν είναι να σχεδιάζουμε εμεί αυτό που θέλουμε, αλλά οι πολίτε να μπορούν να υλοποιήσουν αυτά που έχουν φανταστεί. Πρέπει να χρησιμοποιούμε λοιπόν όλε τι ευκαιρίε. Μπορούμε να τα πάμε πολύ καλύτερα, διότι σήμερα οι πολίτε σε όλο τον κόσμο αρχίζουν να έχουν τι πρώτε εμπειρίε τη δημοκρατία. Αρχίζουν να συμμετέχουν σε εκλογέ, όπω μια κυρία στη Λιβύη, που για πρώτη φορά μπόρεσε να βάλει την ψήφο της στην κάλπη δεν ήξερε τι θα βγει ω αποτέλεσμα, δεν ήξερε τι θα γίνει στο μέλλον. Ήταν πολύ χαρούμενοι που συμμετείχε. Πρέπει αυτό να το λάβουμε υπόψη σήμερα. Οι Ευρωπαίοι και οι Ευρωπαίε θέλουν να συμμετέχουν, οφείλουν να συμμετέχουν. Θέλουμε όμω να δημιουργήσουμε και ένα κατάλληλο πλαίσιο για όλα αυτά. Σα ευχαριστώ. Eh, και τώρα, διάλογο έρωτα απαντήσεις. Πρώτος ζήτησε το λόγο ο κύριος Ταρκόφσκι. Παρακαλώ. Ο κύριος Γκερέρο. Όχι, Ταρκόφσκι. Well, Πρώτα απ' όλα, καλώς ορίσατε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Χαιρόμαστε που μπορεί να γίνει αυτή η συζήτηση εδώ πέρα. Θα ήθελα να σα ρωτήσω για κάτι. Νομίζω Φρίτσαφ είχε κάνει μια διάκριση ε, μεταξύ νομοποίησης ε, αποτελεσμάτων και εισφορών και αν θεωρείτε πως ε, εξακολουθεί να υπάρχει γιατί το πρόβλημα το οποίο έχουμε τώρα όσον αφορά την νομοποιηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι πως αποτεχάνουμε όσον αφορά τα αποτελέσματα γιατί οι πολίτες Μπορεί να μην ήξεραν πολλά για τη δημοκρατία, ο μέσος πολίτης δεν σκέφτεται τις διαφορετικές αυτές έννοιες, αλλά τουλάχιστον υπήρχαν αποτελέσματα και η νομοποίηση των αποτελεσμάτων υπήρχε. Και το πρόβλημα είναι πώς αποτυγχάνουμε ε, ως αυτό. Και ακόμα και άνθρωποι οι οποίοι δεν είναι ειδικοί δεν ε, αντιλαμβάνονται πως δεν έχει ε, αποτελέσματα. Αυτή η υπερεθνική δομή. Και βεβαίως δεν ήρθαν πιο κοντά στου πολίτε ε, τόσα χρόνια, γιατί αποδεικνύεται πως αυτά τα οποία κάναμε εντό της Ευρωπαϊκή Ένωση, παρά το ότι εμεί ξέραμε πως ήταν απαραίτητα, δεν έπιαναν και δεν γοήτευαν την φαντασία του κόσμου και βέβαια δεν κάναμε τίποτα για την οικονομική διακυβέρνηση που είναι τα βασικά προβλήματα. Και βεβαίω το ζήτημα είναι ακριβώς ε, εάν θεωρείται πώ είναι σημαντική αυτή η νομοποίηση των αποτελεσμάτων ή αν κατά μία υπάρχουν αυτές οι ελλείψεις. Το Γερμανικό Ομοσπονδιακό Δικαστήριο, ειδικά όσον αφορά την απόφαση τη ε, Λισαβόνα είπε πως δεν είχε τέλεια νομιμοποίηση το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Α, βεβαίω ασχολήθηκε μόνο με τις έδρες, χωρίς να δει την ευρύτερη εικόνα. Γιατί είναι δύσκολο να μιλήσουμε για τις έδρες εδώ μέσα, για την κατανομή των εδρών. Γιατί επανέρχεται αυτή η συζήτηση, γιατί πρέπει να αποφασίσουμε σχετικά ε, τη στιγμή που θα ενταχθεί η Κροατία. Γιατί για χρόνια αυτό γινόταν παράλληλα με τις ψήφους στο Συμβούλιο. Και αυτή ήταν η ισορροπία η οποία έδινε κάποια δημοκρατική λύση. Αν κοιτάξουμε μόνο το ένα κομμάτι της εξίσωσης, βέβαια υπάρχουν προβλήματα. Και υπάρχουν βεβαίως διαφορετικές ιδέες, όχι όσον αφορά την ομοποίηση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αλλά το να γίνει, να, να φανεί περισσότερο στους πολίτες για να δουν πώς λειτουργεί η υπερεθνική δημοκρατία και αυτά μπορεί να γίνουν χωρίς αλλαγή της ε, συνθήκης. Το πρόβλημα που έχουμε είναι πως όταν γίνονται ευρωεκλογές τα θέματα είναι μόνο εθνικά. Κανένας δεν ενδιαφέρεται για το τι συμβαίνει μετά. Και τα εθνικά μας κόμματα στα οποία όλοι ανήκουμε δεν ε, ασχολούνται με ευρωπαϊκά ζητήματα. Και κυκλοφορούν βεβαίως ε, διάφορες ιδέες και κυκλοφορούσαν. τους χάρη. Δεν έχουμε συγκεκριμένο πρόγραμμα Ευρωπαϊκού Κόμματος. Ε, βεβαίως, επί τη ευκαιρία επεξεργαζόμαστε το καταστατικό των Ευρωπαϊκών Κομμάτων και ε, Βεβαίω πρέπει να πηγαίνουμε στι εκλογέ με ξεκάθαρη πλατφόρμα, δηλαδή τα κόμματα του ΕΛΚ να λένε αυτό είναι το πρόγραμμά μα. αυτή είναι η συνταγή δική μας για τα προβλήματα. Αυτός είναι ο υποψήφιός μας για πρόεδρος της Κομισιόν και αν ψηφίζετε μας, αυτά θα βρείτε μπροστά σα. Και αν έχουμε εμεί την πλειοψηφία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ε, προ τα εκεί θα πάει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί βεβαίω ε, αυτό θα είναι ο πρόεδρο τη Κομισιόν, η πλειοψηφία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Βεβαίω θα υπήρχαν και υπερεθνικέ λίστε που είναι δημοφιλεί μόνο εδώ μέσα, αλλά όχι στην Ολομέλεια βεβαίω, ε, καθώ θέλαμε να εκλέξουμε ένα μικρό αριθμό βουλευτών σε υπερεθνική λίστα. Το ερώτημα είναι εάν οι απόψεις Αυτέ θα μπορούσαν να δημιουργήσουν ένα ευρωπαϊκό δημόσιο χώρο. Δεν μιλάω για ευρωπαϊκό δήμο βεβαίω. Δεν ξέρω εάν το επιθυμούμε και αυτό. These questions can be debated and then when citizens see it that that... Και βεβαίω, ε, έτσι θα ε, υπάρξει μία κάποια νομιμοποίηση. Βεβαίως ε, Το ζήτημα είναι το να επιλύονται πραγματικά τα προβλήματα. Οπότε, ποια είναι η θέση η δικιά μου. Δεν γίνεται επανάσταση, δεν θα αλλάξουν οι συνθήκες, δεν θα αλλάξει η αντίληψη του κόσμου μέσα σε λίγα χρόνια. Αλλά τουλάχιστον εάν αλλάξει το κέντρο της συζήτησης και ε, πάει στο στυλ αυτούς τους ανθρώπους θέλω, ψηφίζω αυτό το πρόγραμμα, Εντάξει, μπορεί να μην ξέρω τα πάντα για τα ευρωπαϊκά, αλλά τουλάχιστον έχω αυτές τι συγκεκριμένες απόψεις και θέλω να λυθούν τα προβλήματα και άρα νομοποίηση των αποτελεσμάτων. Θέλετε να απαντήσετε στην κάθε μία ερώτηση ή στο τέλος των διαφόρων παρεμβάσεων. Αμέσως. Ωραία. Yeah. Uh, um, I'm very happy about this intervention because it allows... Χάρηκα για αυτή την παρέμβαση γιατί μου επιτρέπει να ξεκαθαρίσω κάποια πράγματα. Ναι, υπάρχουν άμεσες ε, σχέσεις ε, μεταξύ αυτών των οποίων λέτε και αυτά τα οποία είπε. Κοιτάξτε, αναφέρατε βεβαίως σε έναν άνθρωπο ο οποίος είναι απεσιόδοξος γιατί το μόνο το οποίο λέ, θεωρεί πως μπορούμε να επιτύχουμε στην, ε, με την Ευρώπη είναι να πούμε πως η Ευρώπη έχει αποτελέσματα. Η κρίση σήμερα για ΣΑΡΠ, Μαγιών και λοιπούς είναι πως η κρίση αυτή έχει τεράστια σημασία γιατί δεν φέρνουμε αποτελέσματα. Και ενισχύοντας την τεχνοκρατική πτυχή της Ένωσης, πάλι δεν θα επιτύχουμε αυτό το οποίο θέλουμε. Στην κατάσταση αυτή, η λειτουργία ε, ενός φόρουμ όπως το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ε, καθίσατε ακόμη πιο σημαντική. Όχι ότι το Κοινοβούλιο μπορεί να πει ότι τώρα θα λάβουμε την απόφαση για το τι θα γίνει για την Ελλάδα, ε, τι θα γίνει με τη γερμανική ηγεμονία, αλλά να δοθεί μια φωνή στις διαφορετικές αυτές προοπτικές και να αντιληφθούν οι άνθρωποι στην Ευρωπαϊκή Ένωση Ε, να αντιληφθεί άνθρωπο πως συζητιούνται αυτά τα ζητήματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και να πιστούν να επικοινωνήσουν με ένα διαφορετικό τρόπο. Το φοβερό σήμερα είναι η αντίληψη των ανθρώπων μεταξύ άλλων. Και από ό,τι κατάλαβα, η δική σας πρωτοβουλία είναι να εξηγήσετε πως το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι ένας χώρος πολιτικοποίησης στην Ευρώπη χωρίς να δημιουργεί βεβαίως έναν Δήμο που θα μας επέτρεπε να ε, αποφασίσουμε το ότι είναι σωστό για την Ένωση παντού, αλλά για να βρει μια τομή μεταξύ των πιο περιφερειακών ανησυχιών και της κοινή δέσμευση ε, της Ευρώπης σε ζητήματα δημοκρατικών αποφάσεων και κάποιες ε, αναδιανομής. Και Κάφμαν θέλετε να πείτε και εσείς κάποια πράγματα. Ναι, βεβαίως. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να μιλάμε για την νομοποίηση των αποτελεσμάτων και όταν μιλάμε για δημοκρατία, η διαφορά μεταξύ δημοκρατίας και μη δημοκρατίας βεβαίως δεν αφορά την νομοποίηση των αποτελεσμάτων αλλά την νομοποίηση των ε, συνεισφορών. Γιατί και η χειρότερη δημοκρατία μπορεί να πει έχω αποτελέσματα, άρα νομοποιούμε. Οπότε θα πρέπει να α, να σκεφτούμε παραδείγματο χάρη το, την πιθανότητα να λέμε πω ναι, εντάξει, οι άνθρωποι είναι ικανοποιημένοι, υπάρχουν αποτελέσματα και δεν μα ενδιαφέρει πράγματι η νομοποίηση της, ε, των συνεισφορών. Και βεβαίως, εφόσον είναι ατελείς οι δημοκρατίες μας, εγώ δεν θα έλεγα πως εφόσον η Ευρώπη έχει αποτελέσματα δεν χρειάζεται να συζητήσουμε άλλο αυτή την πτυχή του ζητήματος. Ευχαριστώ. Ο κύριος Μπρόνς. Αν είχα μία λίρα ή και ένα ε, ευρώ για κάθε φορά που άκουσα τη λέξη δημοκρατία σήμερα θα ήμουν πολύ ευτυχής. Αλλά βεβαίως έχω. Είναι τα έξοδα παραστάσεως που μου δίνουν. Εν πάση περιπτώσει. Υπάρχει καμιά φορά αντίστροφη σχέση μεταξύ της χρήσης της λέξη δημοκρατία και της πραγματικότητας, αρκεί να κοιτάξουμε τις επίσημες ονομασίες χωρών ε, ανά τον κόσμο. Όσος λέγονται δημοκρατίες ε, και λαϊκές δημοκρατίες συνήθως είναι οτιδήποτε άλλο εκτός από αυτό. Βεβαίως, για να είμαστε δίκαιοι, κάποια ε, θεσμικά όργανα έχουν πράγματι αποτελέσματα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση όμως θέλει δημοκρατική νομιμοποίηση για αυτά τα οποία έχει ήδη αποφασίσει. Οπότε οι δομές και οι διαδικασίες επινοούνται με τον ε, στόχο τον εκπεφρασμένο πως οι δημοκρατικές διαδικασίες είναι σωστές. Μάλιστα έχουν επινοηθεί για κάποιες λέξεις. Ακούσαμε κάποιες για δημοκρατικές αποφάσεις οι οποίες δεν είναι οι σωστές. Ε, ακούμε παραδείγματος χάρη τη λέξη λαϊκισμός η οποία χρησιμοποιείται λάθος. Ο λαϊκισμός ε, αναφέρθηκε και ξεκινήσε στην Αμερική ε, και θεωρεί το, το να απευθύνεται κανείς στους ανθρώπους ε, αδιακρίτως κλάσης. τάξης, με συγχωρείτε. μια άλλη λέξη που ακούστηκε ήταν το παράλογο και αυτό πάλι αφορούσε τη λάθος δημοκρατική απόφαση. Βεβαίως όταν γίνεται ένα δημοψήφισμα και η απάντηση είναι η λάθος η απάντηση είναι έτοιμη. Α, θα ξανακάνουμε δημοψήφισμα. Και στην ε, περίπτωση στην οποία έχουμε δύο φορές λάθος απάντηση, φαντάζομαι δεν θα κολλήσουμε τρίτο και τέταρτο δημοψήφισμα. Είχαμε δεύτερο δημοψήφισμα στην Δανία για το Μάστριχτ, δύο στην Ιρλανδία για τη Λισαβόνα και δύο για το Δημοσιονομικό Σύμφωνο. Βεβαίως, όταν απορρίφθηκε η συνταγματική συνθήκη στη Γαλλία και στην Ολλανδία, δεν έγιναν εκεί πέρα δεύτερα δημοψηφίσματα, απέσυραν τη συνθήκη. Την έβαλαν σε ένα άλλο πακέτο, παρά το ότι εδώ μέσα το παραδέχτηκαν κάποιοι πως μόνο αυτό έγινε, η συσκευασία άλλαξε και δεν έγιναν μετά καθόλου δημοψηφίσματα. Ωραία δημοκρατία. Βεβαίως, μπορεί να ανατραπεί και με άλλους τρόπους η λάθος απόφαση. Εάν ε, ξοδευτούν πάρα πολλά λεφτά υπέρ του νέου, όπως το Ηνωμένο Βασίλειο το 1975 ή τώρα πρόσφατα στην Κροατία, όπου επέρονταν για το πόσα λεφτά ξόδευαν για την πληροφόρηση του κοινού. Πληροφόρηση εννοούμε προπαγάνδα βεβαίως. Όταν μιλάμε για τις πρωτοβουλίες πολιτών, έτσι, για την περίπτωση κατά την οποία ε, λάβουν λάθος Πρωτοβουλίε οι πολίτες. Πρώτα απ' όλα περιορίζουμε τις ερωτήσεις, λέμε πω δεν πρέπει να είναι υπουσιώδεις. Αλλά αυτό ποιο το κρίνει. Μετά πρέπει να τηρεί τις ευρωπαϊκές αξίες. Ε, άρα αυτομάτως κόβονται κάποιες προβληματικές και ο κύριος Σεύκοβιτ προσέθεσε και ένα τρίτο κριτήριο. Είπε πως πρέπει να είναι προς το συμφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης και πάλι κάτι το υποκειμενικό. Αλλά βέβαια θα μιλάμε για τη μέθοδο, για το 1 εκατομμύριο υπογραφές σε διάφορες χώρες. Κατ' ουσίαν μόνο μεγάλες οργανώσεις μπορούν να φτάσουν αυτό τον αριθμό. Κόμματα, συνδικάτα, επιχειρήσεις. Η ιδέα πως ο απλός κόσμος, ένα εκατομμύριο απλοί άνθρωποι σε διαφορετικές χώρες, αυθορμήτω θα αναλάβουν μια πρωτοβουλία, είναι επικίνδυνη ψευδέστηση. Οπότε, αυτό το οποίο θέλει η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι συμμετοχή των ανθρώπων, αλλά με τους δικούς της όρους. Δηλαδή να συμμετέχουν υπακούοντας. Και μάλιστα δεν είναι κάτι το αυθόρμητο από κάτω προς τα πάνω, αλλά από πάνω προς τα κάτω. Ένας δημοκρατικός συγκεντρωτισμός. Και πολλοί βεβαίως λένε πως ε, είναι πολλοί οι άνθρωποι και ε, οι ψήφοι και άρα είναι δημοκρατία. Μα είναι μύθος ότι οι δεσποτείε δεν θέλουν να ψηφίζει ο κόσμος. Μάλιστα, τους υποχρεώνουν κιόλα. Το... Θέλετε να απαντήσετε ή να ακούσουμε και άλλου. Περιμένετε, θα περιμένετε, ακούσουμε και άλλες παρεμβάσει. Ωραία. Ο κύριος Γκερέρο έχει ζητήσει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θέλω να ευχαριστήσω τους εισηγητές και τον κύριο Χέφνερ για τη διοργάνωση της ακρόασης αυτής. Άκουσα την απάντηση που έδωσε ο κύριος Κάφμαν στον κύριο Τρασκόφσκι σε ποιο βαθμό η δημοκρατία είναι μια συνεχής και ατελής διαδικασία που δέχεται πάντοτε βελτίωση. Και θυμήθηκα και ένα βιβλίο του Τζον Ντάν που λέει ότι η δημοκρατία είναι ένα ταξίδι που δεν τελειώνει. Unfinished journey. Έρχομαι στην αρχική σας παρέμβαση. Είπατε ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει μεγαλύτερη επιθυμία για δημοκρατική συμμετοχή περισσότερη, χωρίς όμως να υπάρχουν και οι απαιτούμενες δομές, ώστε να ικανοποιηθεί το αίτημα των πολιτών για περισσότερη συμμετοχή. Είδαμε ότι πράγματι εκφράστηκε η επιθυμία αυτών των πολιτών να συμμετέχει πιο ενεργά στην πολιτική σε τρεις στιγμές συγκεκριμένα τη δεκαετία του 60 Να και λίγο νερό. Όπου μετά από μία περίοδο που η δημοκρατία ε, εννοείται ως κάτι χρηστικό απέναντι στο πολιταρχικό μοντέλο, το οποίο ο Τσέρτσιλ είχε ε, ονομάσει ως το μη χειρονβέλτιστον σύστημα. Υπάρχει λοιπόν στις Ηνωμένε Πολιτείες και στην Ευρώπη και σε πολλές ε, αναπτυγμένες χώρες εκείνη την εποχή επιθυμία να συμμετέχουν πιο ενεργά στην πολιτική. Αυτό χαρακτηρίζει το δεύτερο ήμιση κυρίως στις δεκαετίες του 60. Δεύτερη φάση τώρα πάλι φιλοδοξιά μεγαλύτερη ε, δημοκρατικής συμμετοχής που ορίζεται ως ποιότητα της δημοκρατίας είναι μετά την κατάρρευση του τείχου του Βερολίνου όταν δεν υπάρχει πλέον ε, το αντίπαλον δέο που αμφισβητεί τη φιλελεύθερη πλουραλιστική δημοκρατία. Τότε λοιπόν θέλουμε να εμπλουτίσουμε τη δημοκρατία με πιο ενεργό συμμετοχή των πολιτών. Και εκείνη την εποχή επίσης βιώνουμε την κόποση, αν θέλετε, ε, της αντιπροσωπευτικής δημοκρατίας. Έτσι θα μπορούσαμε να τη χαρακτηρίσουμε. Εγώ προέρχομαι από την Ισπανία. Θα σας θυμίσω ότι στην Ισπανία τα δύο τελευταία χρόνια είχαμε πολύ, αυτό το πολύ ισχυρό κίνημα ε, το, της 11ης ε, Μαρτίου, ανθρώπων, της 15ης Μαρτίου, ανθρώπων που νιώθουν απομακρυσμένοι και αποξενωμένοι και από την αντιπροσωπευτική δημοκρατία. Και η πρόκλησή μας είναι να συνδυάσουμε την αντιπροσωπευτική δημοκρατία, την ανάθεση καθηκόντων, ε, εκχώρηση αρμοδιοτήτων, και να το συνδυάζουν, παραλαμβάνω, με το οικοδόμα της αντιπροσωπευτικής δημοκρατίας που όπως είπε ο Σαρτόρη έχει παραμείνει όρθιο αυτό το οικοδόμα για δύο αιώνες, να το συνδυάζουν παραλαμβάνω με την ισχυρή δημοκρατία, με την συμμετοχική δημοκρατία Όπω όπως ε, και εσείς γνωρίζετε πολύ καλά. Είναι ε, και τίτλος του βιβλίου του Μπάρμπερ... Strong Democracy. Ισχυρή δημοκρατία, συμμετοχή λοιπόν δεκαετίας 90 ε, εκείνης εποχής. Πρέπει λοιπόν αυτή την επιθυμία των πολιτών να προχωρήσουμε ακόμη περισσότερο από τις τυπικές διαδικασίες, περιοδικές διαδικασίες αντιπροσωπικής δημοκρατίας, πρέπει να το ε, διοχετεύσουμε αυτό το αίτημα κάπου. Σίγουρα πρέπει να ξέρουμε ε, και αν υπάρχει στο μεταξύ, μεταξύ δύο διαδικασιών, αν υπάρχει έλεγχος στο μεσοδιάστημα ή όχι. Υπάρχει λοιπόν η συμμετοχή, η επιθυμία για συμμετοχή και αυτό προσκρούει ε, σε κάποια σύγχυση μεταξύ δημοψηφίσματος και συμμετοχής δημοκρατίας. Τι θέλω να πω. Εάν η δημοκρατία, αντιπροσωπευτική δημοκρατία, μάλλον συμμετοχική διορθών, μεγαλύτερη δημοκρατική συμμετοχή, ισοδυναμεί με δημοψήφισμα, υπάρχει πρόβλημα. Γιατί το δημοψήφισμα σε πολλέ περιοχέ, σε πολλέ χώρε έχει ιστορία, έχει παράδοση, ίσω και αρνητική. Ιταλία, για παράδειγμα, για δεκαετίε χρησιμοποίησαν τα δημοψηφίσματα οι εξοκοινοβουλευτικέ δυνάμεις και ουσιαστικά ε, είναι το δημοψήφισμα ένα παιχνίδι μεταξύ του όλα ή τίποτα ουσιαστικά. Και υπάρχουν κάποιες κρίσιμες στιγμές που οι πολίτες δεν ψηφίζουν ακριβώς αυτό που τους ερωτούν στο δημοψήφισμα, αλλά επηρεάζονται από τις καταστάσεις, ε, ε, την πολιτική κατάσταση, τις διαθέσεις τους κτλ. Σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες, να πω επίσης, και να δώσω ένα παράδειγμα την Ισπανία για να μην πάμε πιο μακριά, εάν σε κάποια στιγμή ε, όξυνση τη τρομοκρατία τη ΕΝΤΑ είχαμε ένα δημοσίευμα για την θανατική ποινή, υπάρχει πιθανότητα οι πολίτε να είχαν ψηφίσει υπέρ της θανατική ποινή. Εάν γίνει τώρα αυτό το δημοψήφισμα που αποφάσισε η ΕΤΑ σίγουρα να έχει με την εκεχήρια, σίγουρα δεν θα είχαμε αυτό το, ψήφι, αυτό το αποτέλεσμα στο δημοψήφισμα. Δεν θα ψήφιζαν υπέρ τη θανατική ποινή οι Ισπανοί δηλαδή. Είναι πολύ πλοκά λοιπόν τα πράγματα. και πού πρέπει τελικά, προ τα πού πρέπει να οδεύσει η συμμετοχη δημοκρατία. λοιπον δεν άκουσα όλη σας την παρέμβαση, αλλά από αυτά που άκουσα, πρέπει να σας πω ότι πράγματι αυτό που προτείνεται είναι πολύ σωστό, γιατί μπορούμε να δημιουργήσουμε δομές και διαδικασίες για να είναι η συνήθιση να μην είναι κατά περίπτωση και σε κρίσιμες περιόδους αυτή η συμμετοχή, να είναι κάτι σταθερό που θα διαμορφώνει ε, την κοινή γνώμη και, τις, ε, και θα ε, εμπνέει τις αποφάσεις που θα λαμβάνονται. Και είναι πάρα πολύ χρήσιμη αυτή η περίοδος για να δημιουργήσουμε αυτές τις υποδομές, θα έλεγα. Για τους λόγους που αναφέρετε κι εσείς, γιατί υπάρχει αυτή η νομοθετική πρωτοβουλία των πολιτών, αλλά και γιατί κυρίως είμαστε στο μετέχμιο μιας διαδικασίας συνταγματοποίησης, αν θέλετε, σε ένα ε, ανώτερο επίπεδο, διαφορετικό επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτή τη στιγμή ε, κυοφορείται, είναι στα σπάργανα όλα τα σχετικά με την ε, Τραπεζική Ένωση, το συντονισμό της φορολογικής και δημοσιονομικής πολιτικής, δημοκρατική συμμετοχή, ρόλο κοινοβουλίου κτλ, κτλ. Θα πρέπει να δούμε τι θα προκύψει σε μια δεκαετία θα δώσει αυτό στα 10 χρόνια τα επόμενα. Θα μπορούσαμε να προτείνουμε και εδώ στο κοινοβουλευτικό επίπεδο και στο ακαδημαϊκό επίπεδο κάποιους μηχανισμούς συμμετοχής που θα συνοδεύουν τη συζήτηση αυτή για τη νέα συνταγματοποίηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ώστε τελικά να μην πραγματοποιεί υπόθεση σε 10 χρόνια να αποφασίζονται τα πάντα, όλα αυτά, με ένα δημοψήφισμα σε κάποιες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Που άντε να ξέρουμε τώρα τι ε, διάθεση ε, θα έχουν οι πολίτες. Μπορεί να είναι πάρα πολύ αισιόδοξοι γιατί θα έχουμε υπερβεί την οικονομική κρίση ή μπορεί να είναι πάρα πολύ απεσιόδοξοι γιατί θα έχει εμβαθυνθεί η δημοσιονομική κρίση. Άρα το αποτέλεσμα του υποθετικού αυτού δημοψηφίσματος θα στρέβλωνε ουσιαστικά ε, δεν θα απαντούσε στο ερώτημα που θα έχετε στους πολίτες. Ελπίζω να μην σας μπέρδεψα με αυτά που είπα, να μην ήταν συγκεχημένη η παρέμβασή μου. Θέλω να ε, κλείσω επισημένοντας για μια ακόμη φορά ότι υπάρχει αίτημα και διεκδίκηση των πολιτών για ποιο συμμετοχή δημοκρατία πρώτον. Δεύτερον, πρέπει να βρούμε κάποιους κανονικούς τυπικούς μηχανισμούς δημοκρατικής συμμετοχής και να μην στρεφόμαστε μόνο κατέσκατον στα δημοψηφίσματα. Και τρίτον, πρέπει ε, να ε, καταλάβουμε ότι έχει δρομολογηθεί, τέλο πάντων στα Σπάργανα, μια νέα φάση συνταγματοποίηση, επαναλαμβάνω, τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Σας ευχαριστώ. Να ευχαριστήσω και τους ε, εμπειρογνώμονές μας και θέλω και εγώ να θέσω ένα ερώτημα. Και φαντάζομαι και ο κύριο Χέφνερ δεν θέλει, θα θέλει να παρέμβει. Η ερώτηση μου είναι η εξή. Ήδη πριν από τη συνθήκη της Λισαβόνας, το δικαίωμα υποβολής αναφοράς ήταν το κατεξοχήν περιεχόμενο και η κατεξοχήν έκφραση της Ευρωπαϊκής Ιθαγένειας. Τώρα φαίνεται να υπάρχει διαφορά μεταξύ της πρωτοβουλίας των πολιτών βάσει του άρθρου 11, των αναφορών όπως υπήρχαν προηγουμένως, αλλά δεν μπορούμε να πούμε ότι η διαφορά είναι ποσοτική, ή ο αριθμός των υπογραφών δηλαδή. Αυτό μπορούσε και προηγουμένω να ισχύει. Μια αναφορά θα μπορούσε να υπογραφεί όχι μόνο από έναν ή εκατό πολίτε, αλλά από εκατομμύρια, αν ήθελε κάποιο να το οργανώσει. Η διαφορά αυτή λοιπόν δεν είναι αυτή που κάνει σημαντικότερη την πρωτοβουλία των πολιτών. Η διαφορά είναι ότι τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα οφείλουν να λάβουν υπόψη το αίτημα που προωθεί η πρωτοβουλία. Αποφασίζεται να γίνει αποδεκτή ή να μην γίνει αποδεκτή η πρωτοβουλία μεν, αλλά σε κάθε περίπτωση γίνεται συζήτηση, προξενείται και ε, προκύπτει υποχρέωση να οργανωθεί συζήτηση σε κάποιο επίπεδο. Πρέπει λοιπόν να δούμε ποιο είναι το κατάλληλο επίπεδο για να γίνεται αυτή η συζήτηση της πρωτοβουλία των πολιτών. Διότι το να παραμένουν τα αιτήματα σε ένα σιρτάρι χωρίς να γίνει ποτέ εμβάθυνση σε αυτή την περίπτωση σημαίνει ότι ελαχιστοποιεί τη σημασία του δικαιώματος διοργάνωσης πρωτοβουλίων. Έπειτα, το άρθρο 11 λέει ότι η πρωτοβουλία των πολιτών πρέπει να οδηγήσει σε νομική πράξη υλοποίηση των συνθήκων. Αυτό σημαίνει και ότι υπάρχει ανάγκη μεταρρύθμισης των συνθήκων βέβαια, αλλά ανοίγονται νέες δυνατότητες μέσα από τις συνθήκες. Θα ήθελα τώρα να ακούσουμε τον κύριο Χέφνερ. Ja, das ist ganz wunderbar, weil Sie mir... Ναι, θαυμάσιο αυτό γιατί μου πήρατε από το στόμα το, το ερώτημα και οι δύο έχετε ασχοληθεί εντατικά με τις ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες πολιτών και τις αναφέρατε. Το ερώτημά μου είναι τώρα που έχουμε ένα εξάμεινο εμπειρία, βεβαίως δεν, δεν αρκεί καμία πρωτοβουλία πολιτών, δεν έχει ολοκληρώσει τη συλλογή των υπογραφών, αλλά βλέπουμε ήδη πολλά πράγματα, βλέπουμε ποια θέματα επιτρέπονται, που η Κομισιόν απορρίπτει γιατί λέει πως δεν επιτρέπεται το τάδε πράγμα. Βλέπουμε ποια προβλήματα υπάρχουν με την συλλογή υπογραφών στο διαδίκτυο και το software, αλλά πάνω πολλά να το πω ως εξής. Δεν ε, έχει εκπληρωθεί μέχρι τώρα η προσδοκία πως θα προκύψουν μεγάλες συζητήσεις στην Ευρώπη διασυνοριακές. Το ερώτημα είναι, αυτό οφείλεται στο ότι είναι ακόμα πολύ νωρίς, μήπως το ότι πράγματι είναι πολύ περιοριστικός ο κανονισμός. για το ότι Ε, υπάρχει ερμηνεία πως αποκλείεται πλέον ε, περαιτέρω από αλλαγή της συνθήκης μέσω αυτής της διαδικασίας εκεί οφείλεται, οφείλεται στο περιορισμένο αριθμό χαρακτήρων ε, του κειμένου Δηλαδή θα θέλαμε τις πρώτες δικές σας υποδείξεις για το τι μπορούμε να κάνουμε για να ξεκινήσει η διαδικασία και να επιτύχουμε αυτό το οποίο είπε ο Μπρουνο Κάφμαν. Δηλαδή, περισσότερο κόσμος στην Ευρώπη δεν το έχει αντιληφθεί καν ότι υπάρχει κάτι τέτοιο. Και πρέπει να το αντιληφθεί και να το χρησιμοποιήσουμε το δεύτερο. Αυτό το οποίο είπε ο Ενρίκε Γκερέρο Σαλόμ εμέσως. Μπρούνο Κάφμαν, είπες πως, εάν κοιτάξουμε προς τα πίσω, υπήρχαν ήδη 53, 53 δημοψηφίσματα στην Ευρώπη για ζητήματα Ευρώπης. Εδώ πέρα, ξέρετε, ε, είμαστε πολύ επιφυλακτικοί απέναντι στα δημοψηφίσματα, κατά το οποίο οπωσδήποτε σχετίζεται με τα αρνητικά αποτελέσματα. Στη Γαλλία, Ολλανδία, Δανία, Ιρλανδία για τις διάφορες συνθήκες. Και προβάλλεται το επιχείρημα πως ε, δεν ε, απαντούν οι πολίτες στο ερώτημα το επίμαχο, αλλά σε διάφορα άλλα ζητήματα, ε, ζητήματα προσώπων, ότι στη Γαλλία καταψήφισαν λόγω Ιράκ, ας πούμε, κτλ ή αυτό το οποίο είπε ο Ενρίκε ε, ή εκεί όπου περιορίζεται το δημοψήφισμα στην απάντηση όχι. Ναι ή όχι, αλλά δεν μπορεί να δημιουργήσει νέες ε, πρωτοβουλίες. Γι' αυτό θα ήθελα εγώ να σας ρωτήσω εσάς τους ε, ειδικούς προώτων πώς μπορούμε να κρίνουμε την επίδραση των δημοψηφισμάτων σε ευρωπαϊκό επίπεδο, να το δούμε κάπως μακροπρόθεσμα, και πώς μπορούν να διαμορφωθούν τα δημοψηφίσματα για να απαντάει ο κόσμος στο ερώτημα της ουσίας και όχι σε άλλα πράγματα. Και βεβαίως αυτό τίθεται με το ζήτημα βεβαίω του επιτρεπτού των ερωτημάτων αλλά και τη ίδια τη διαδικασία. σω ε, μπορείτε να μας διαφωτίσετε. Α, και ένα τρίτο ε, ερώτημα που με ενδιαφέρει εμένα. Είναι σε θέση οι άνθρωποι τελικά να αποφασίσουν ich aus meiner eigenen Erfahrung als jemand, der sehr viel είναι ικανή για κάτι τέτοιο. Γιατί έχω και εγώ τέτοια εμπειρία από αμεσοδημοκρατικές ε, διαδικασίε και είχα μια τέτοια εμπειρία και είναι το συναρπαστικό είναι πως ε, τα μέσα αυτά δίνουν την δυνατότητα στον άνθρωπο να αισθανθεί πως και αυτός παράγει Κάτι πήχε στη Βαυαρία, είχαμε ένα δημοψήφισμα για το ζήτημα της διάθεσης των απορρίτων. Ε, πολύ σημαντικό ζήτημα, ε, αλλά εξειδικευμένο. Και το, το προτείναμε τότε στην τοπική βουλή και λέγανε «Μα είναι πολύπλοκο, δεν καταλαβαίνουν οι άνθρωποι από τέτοια πράγματα». Αλλά τελικά έγινε το δημοψήφισμα και είχαμε εννέα μήνες συζητήσεων, κάθε δήμος ε, έκανε εκδηλώσεις και το συναρπαστικό ήταν πως ο πληθυσμός, ο λαός συζητούσε αυτό το ζήτημα και έλαβε τελικά μια λογική απόφαση για την οποία ήταν περήφανη και η κυβέρνηση. Και τελικά καταλήξαμε στην πιο σύγχρονη πολιτική διάθεση απορριμμάτων σε ολόκληρο τον κόσμο. Αλλά μετά από αυτή τη συζήτηση, η οποία ήταν, όπως σας είπα, πάρα πολύ έντονη. Μήπως θα ήταν λοιπόν δυνατόν να γίνει αυτό και σε άλλα επίπεδα. Θα ήταν οι προϋποθέσεις για κάτι τέτοιο. Θέλετε να απαντήσετε. Εσείς ίσως. Κύριος Κάφμαν. Ναι. Βλέπω πως υπάρχει δυνατότητα να μιλήσω σου ειδικά, οπότε θα την εκμεταλλευτώ. Έτεθησαν διάφορα ερωτήματα. Για την δημοκρατία λοιπόν, τη συμμετοχική δημοκρατία και πώς μπορεί αυτό να συνδυαστεί με όλα τα υπόλοιπα. Ιδίως με τα δημοψηφίσματα. Ο Βρετανός βουλευτής επέκρινε την μέχρι τώρα χρήση του όρου δημοκρατία. Πρόσφατα στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λονδίνου χρησιμοποιήθηκε η κορεάτικη σημαία της Βορείου Κορέας. Και κάποιοι αναρωτήθηκαν αν είναι σωστό αυτό, αν είναι δημοκρατικό. είναι δημοκρατία η δυνατότητα να γίνεται συζήτηση, διάλογος πριν τη λήψη αποφάσεων. Υπάρχουν συλλογικά και ατομικά δικαιώματα που προστατεύουν τους πολίτες και τις επίσημες αποφάσεις τις λαμβάνει η πλειοψηφία. Αυτά πρέπει να ισχύουν για να ονομάζεται κάτι δημοκρατία. Η διάσταση του διαλόγου είναι αυτό που εννοούμε όταν λέμε συμμετοχική δημοκρατία. Δεν υπάρχει δημοκρατική απόφαση αν κανείς δεν είχε την δυνατότητα να την συζητήσει προηγουμένω. Το θέμα είναι ποιο μπορεί να συμμετέχει βέβαια σε τέτοια συζήτηση. Εκεί πρέπει να υπάρχει συνέπεια στο σύστημα. Δεν μπορεί να είναι μόνο μια μικρή ομάδα που λαμβάνει αποφάσεις. Πρέπει όλοι να συμμετέχουμε στη διαδικασία αυτή. Πρέπει να βρίσκονται λύσεις που να επιτρέπουν την ε, επίτευξη στόχων και να έχουμε αποτελέσματα. Θα πρέπει δηλαδή να μην υπάρχουν αντιφάσεις και διαφωνίες ή σύγκρουση, αλλά αλληλοσυμπληρωματικότητα. Μας ενδιαφέρει να βλέπουμε και τα αποτελέσματα στα οποία οδηγούν οι αποφάσεις. Πολλές φορές μπορεί να επηρεάζονται οι εκλογές και τα εκλογικά αποτελέσματα ή μπορεί να έχουμε δημοψήφισμα και τα αποτελέσματά τους να έχουν κάποια σημασία, όμως το θέμα δεν είναι να συζητούμε την έννοια της δημοκρατίας μετά από μια εκλογική ή ταϊνίκη, αλλά να είναι σωστά καταρτισμένη η ολόκληρη διαδικασία. Εάν θέλουμε λοιπόν να δούμε τα θεμέλια της δημοκρατίας ή το θέμα του ελλείμματος που συνεχώς τίθεται στην καθημερινότητά μας, εκεί συνειδητοποιούμε ότι πρέπει να υπάρχουν κάποιοι κανόνες του παιχνιδιού, κάποιοι κανόνες που να επιτρέπουν σε αυτή την πραγματικότητα να πάρει σάρκα και οστά. στο κάτω-κάτω της γραφής δεν μπορεί να υπάρχει άμεση δημοκρατία χωρίς να υπάρχουν εκλογές συστηματικά, χωρίς να υπάρχει κάποια συμμετοχή, χωρίς να υπάρχουν εγκαθεντρημένα δικαιώματα, το δικαίωμα πρωτοβουλίας λόγου χάρη, έστω και με την διοργάνωση δημοψηφισμάτων. Το πρόβλημα είναι κυρίως ότι τα δημοψηφίσματα μπορούν να οδηγούν σε πολύ διαφορετικές διαδικασίες. Όμως την απόφαση, την ευθύνη την αναλαμβάνουν οι πολίτες. Είναι υψηλότερο το επίπεδο δημοκρατίας αυτό, παρόλο που μπορεί να υπάρξουν καταχρήσεις από πλειοψηφίες μπορεί να ασκήσουν επιρροή και να περνάνε τις δικές τους ε, επιλογές. Σε κάθε περίπτωση υπάρχουν και δημοψηφίσματα τα οποία είναι διοργανωμένα κατά τρόπο ώστε να δίνουν συγκεκριμένο αποτέλεσμα δεν είναι καθόλου δημοκρατικά βέβαια και είναι μια κατάχρηση αυτή της δημοκρατίας. Στο ευρωπαϊκό όμω επίπεδο έχουμε τη διαδικασία των Ευρωπαίων πολιτών, ε, της πρωτοβουλίας των Ευρωπαίων πολιτών. Αναφέρθηκε πολλά και σε αυτό. Όμως για την ώρα είναι μια αδύναμη διαδικασία δεν είναι αρκετά ελκυστική για να διασφαλίσει ότι θα διοργανωθούν ευρείε συζητήσει, διαβουλεύσει για το όλο θέμα. Ίσως να είναι τόσο μεγάλη η φόβη ότι θα υπάρξει θεσμοθέτηση με όρια ανώτατα και κατώτατα για να προχωρήσει η διαδικασία που αυτό μπορεί να αποθαρρύνει τους πολίτες. Μπορεί ας πούμε να υπάρχει τοποθέτηση για κάποια θέματα που τίθενται ότι δεν είναι θεμητό να συζητηθούν, ότι δεν είναι σκόπιμο. Αυτό μπορεί να αποθαρρύνει τους πολίτες. Εδώ πρέπει να δούμε κατά πόσον είναι και αρκετά ικανοί οι πολίτες στον τρόπο που απευθύνονται και στους εκπροσώπους τους, άλλων όταν ψηφίζουν όπου επιλέγουν απλώς εκπροσώπους, αλλά για να αναλάβουν οι ίδιοι την εξέταση ενός συγκεκριμένου ζητήματος μπορεί να μην έχουν τις απαραίτητες ικανότητες. Αλλά από την άλλη και εμείς δεν μπορούμε να λέμε ότι είναι ανόητοι οι πολίτες ώστε να λάβουν αποφάσεις. Εκλέγουν τους εκπροσώπους του Κοινοβουλίου και αυτό μας φαίνεται λογικό. Πρέπει να βεβαιωθούμε ότι το Ευρωκοινοβούλιο μπορεί να προτείνει και συνταγματικές αλλαγές εφόσον χρειάζονται και οι πολίτες ε, μπορούν να το επιβεβαιώνουν αυτό, να επιβεβαιώνουν τις επιλογές του. Πρέπει να είμαστε συνεπείς. Για την πρωτοβουλία λοιπόν των Ευρωπαίων πολιτών πρέπει να είμαστε κάπως πιο μετριοπαθείς νομίζω. Είναι ένα ξεκίνημα, είναι μια καλή αφετηρία, ένα πρώτο βήμα. Είναι μια ευκαιρία να μάθουμε από την πράξη, να δούμε τι μπορεί να βελτιωθεί και βεβαίω θα υπάρξει και παιχνίδι εξουσία στο πώ θα εφαρμοστεί αυτή η διαδικασία, αλλά ίσω σε ένα-δύο χρόνια να είμαστε πια σε θέση να, το... να διεξάγουμε τα πρώτα συμπεράσματα. Θα έχει δοκιμαστεί. Τώρα απλώ πρέπει να βεβαιωθούμε ότι η πρωτοβουλία των Ευρωπαίων πολιτών μπορεί να είναι καλύτερη. Και δύο λόγια για την πιθανότητα δημοψηφισμάτων σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Δεν σημαίνουν τα δημοψηφίσματα ότι επιλέγουμε ή απορρίπτουμε. Σε μια δημοκρατία πρέπει βεβαίω να μπορεί να, διοργανωθούν δημοψηφίσματα όπω υπάρχει και δυνατότητα εκλογή αντιπροσώπων. Όμω το θέμα είναι πώ θα γίνει αυτό στην Ευρώπη. Ω τώρα είχαμε ε, κρατικά δημοψηφίσματα για την Ευρώπη, όχι ευρωπαϊκά δημοψηφίσματα για άλλα ζητήματα. Σα ευχαριστώ. Πόσο. Ναι, μου ζήτησε να μιλήσω. Λοιπόν, ε, αγαπητοί συνάδελφοι, χαίρομαι πάρα πολύ. Ε, είναι και τιμή μου που είμαι εδώ. Βέβαια, δεν μπορώ να είμαι ε, δύο, σε δύο μέρη ταυτόχρονα παρούσα, γιατί είχαμε και ψηφοφορία στην Επιτροπή Μεταφορών. Να σας καλωσορίσω, να σας ευχαριστήσω για τη δουλειά σας. Και επειδή συζητήσατε και για την ε, πρωτοβουλία των πολιτών, ε, είμαι η μητέρα αυτή τη ε, πρωτοβουλία, θα έλεγα, γιατί συνεισέγραψα τη σχετική έκθεση μαζί με τον Αλέν Λαμασούρ. Πρέπει να σα πω ότι ναι, πράγματι θέλαμε να υπάρχει κάποιο είδου αναθεώρηση και ο Γκέραλτ από την άλλη επιτροπή, γιατί τέλο πάντων τέσσερι είμαστε που είχαμε συμμετοχή σε αυτή την έκθεση. Λοιπόν, είπαμε μετά από τρία χρόνια να έχουμε μια αναθεώρηση ουσιαστικά ε, είναι κάπως ανεξερεύνητα τα ύδατα θα έλεγα και δεν ξέραμε πώς θα ε, εξελιχθεί αυτή η πρωτοβουλία. Θέλουμε πάντως να δώσουμε στους πολίτες ένα εργαλείο για να μπορούν ε, να συμμετέχουν και αυτοί στη δημοκρατία. Να έχουμε λοιπόν συμμετοχική δημοκρατία και θέλουμε και εμείς βέβαια να αξιοποιήσουμε τις δικές σας γνώσεις ως πολιτικοί. Και θα δούμε βέβαια με την αναθεώρηση τι θα γίνει. Στόχος μας πάντως κοινό είναι να λειτουργήσει καλύτερα, όσο το δυνατόν καλύτερα αυτή η πρωτοβουλία. Μιλήσατε για πιλωτικό project. Εγώ λέω, χρειαζόμαστε μια βάση δεδομένων πλήρη. Ε, κάποια πράγματα που έχουμε ζητήσει και από την Κομισιό μας είπε όχι, όχι θα λειτουργήσει. Πρέπει να σας πω ότι εμείς ε, έχουμε κάποιες ιδέες ε, ήδη ε, αποκρισταλώσει για το πώς θα μπορούσε να λειτουργήσει αυτή η πρωτοβουλία και εγώ και ο Γκέραλτ. Καλό είναι λοιπόν που και εσείς μας δίνετε την ε, ε, καθοδήγησή σας, αλλά θα ήθελα να σας ζητήσω να μας στείλετε και περαιτέρω σχόλια, γιατί είναι πολύ καλό να λειτουργήσει καλά αυτή η πρωτοβουλία the left. Ah. It's of course not possible to go through these questions now. It would take much too long also. Δεν μπορώ να απαντήσω όλες αυτές τις ερωτήσεις τώρα. Αλλά είναι μια καλή ευκαιρία να διευκρινίσω αυτά τα οποία έλεγα και να διαφοροποιήσουμε τη δημοκρατία. Θα ξεκινήσω με το σχόλιο από την Ισπανία. Πήγα πέρσι στην Ισπανία όταν ε, ξεκίνησε ε, σε ένα συνέδριο και είδαμε τους νέους στους δρόμους και είδαμε όχι μόνο στην Ισπανία αλλά και αλλού το πώς υπάρχει μια διάθεση σε ένα εθνικό επίπεδο κατά της ευρωπαϊκής διαχείρισης της κρίσης. Γιατί η διαδικασία αυτή λήψη αποφάσεων οδηγεί σε μια πειθαρχία, αν θέλετε, ή διατάζει το εθνικό επίπεδο και για διάφορους κοινωνικο-οικονομικούς λόγους οι κοινότητες αυτές έχουν διαφορετικές απόψεις. Τα, πώς μπορούμε να απαντήσουμε. Να σα πω πώς απάντησε το Γερμανικό Συνταγματικό Δικαστήριο. Λέει το Γερμανικό Συνταγματικό Δικαστήριο. Ναι, πληρώνουμε, αλλά μόνο εάν υπακούτε. Και βεβαίως... Μα, εντάξει, υπερασπιζόμαστε ένα δημοκρατικό δικαίωμα, τη δικαίωμα του Κοινοβουλίου να αποφασίζει για τον προπολογισμό. Αλλά το ίδιο ισχύει για την Ισπανία. Οπότε, τι λέω εγώ, ας αναγνωρίσουμε πως έχουμε αυτά τα δύο πράγματα, αλλά ποια θα ήταν μια δημοκρατική απάντηση και όχι μια υπαγόρευση, μια διαταγή. Αυτό είναι πραγματικά πρόβλημα. Είναι εύκολο να πούμε πως θα βρει κανείς κάτι τέτοιο. Η απάντησή μου είναι Κάπου αλλού λέει η απόφαση του δικαστηρίου πως πρέπει να αποτελέσει μέρος μιας πολιτικής διαδικασίας. Αυτό όμως δεν είναι μια απάντηση για το πώς θα πρέπει να δοθεί στην Ισπανία αυτό το οποίο πρέπει να δοθεί, αλλά η απάντηση είναι να μην δοθεί σε τεχνοκρατικές δομές, αλλά να προσπαθήσουμε να στήσουμε μια δημοκρατική διαδικασία. Και μετά θα συνειδητοποιήσουμε πως οι Γερμανοί, το γερμανικό κοινό, ε, θα δείξει μεγαλύτερη κατανόηση. Αυτή είναι η ελπίδα μας για την δημοκρατία. Εδώ πέρα μπορούμε λοιπόν να δούμε το πώς τα δημοκρατικά δικαιώματα, τη δημοκρατική θεσμή ενός κράτους ε, επιδρούν σε άλλο κράτος. Και αυτό πρέπει να αντιμετωπίσουμε ε, και να δημιουργηθεί μια ε, κοινότητα. Η ελπίδα μου με τις πρωτοβουλίες των πολιτών ε, είναι πως εντάξει θα αποτελέσουν ένα εργαλείο αλλά θεωρώ πράγματι πως η ερμηνεία της Κομισιόν είναι πολύ περιοριστική αλλά ε, γεγονός είναι πως η διαδικασία οργάνωσης ε, κάποιας ευρωπαϊκής συζήτησης θα γίνει όταν μιλήσουμε για πράγματα τα οποία θα ενδιαφέρουν τον κόσμο και δεν πρέπει να απογοητευόμαστε. Τώρα ο κόσμος ασχολείται με, με άλλα ζητήματα. Και δεν πολιτικοποιείται τόσο εύκολα για αυτά τα, τα ζητήματα που θα απασχολήσουν τις ε, πρωτοβουλίε των πολιτών. Άρα η διαδικασία νομίζω θα κινηθεί με το να μαθαίνουμε από τα λάθη μας και μη σας προξενεί εντύπωση το ότι δεν λειτουργεί ακόμα. Ξεκολουθώ να πιστεύω στη δημοκρατία και ότι ο κόσμος έχει ε, συναισθήματα και αυτό το οποίο συμβαίνει αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη, αυτή η κρίση, αυτά μας θυμίζουν πως ο κόσμος δεν αποδέχεται τις τεχνοκρατικέ απαντήσεις. Δεν πείθεται. Και όχι μόνο οι Έλληνες και οι Ισπανοί, οι Πορτογάλοι. Και οι Γερμανοί. Θα σταματήσω εδώ. Σας ευχαριστώ. Νομίζω αυτό την πρώτο κύκλο Τις συναντησίες μας μπορούμε να τον κλείσουμε και να περάσουμε στην επόμενη φάση. Ο κύριος Χέφνερ θα τους παρουσιάσει καλύτερα από μένα βεβαίως και θα διευθύνει τη συζήτηση. Ε, Ευχαριστώ. Μπρούνο Κάφμαν και κύριε Γιώργης. Προτείνω να καθίσετε και να έρθουν εδώ πέρα οι καθηγητές Τέο ε, Σίλερ και Γκέπχαρτ Κίρκεσνα να έρθουν εδώ πέρα. Ο καθηγητής ο κύριος Σιλ ε, διδάσκει στο Πανεπιστήμιο του Μάρμπουργκ και είναι ένας από τους καλύτερους γνώστες και ερευνητές για ζητήματα συμμετοχής των πολιτών και άμεσης δημοκρατίας στην Ευρώπη. Έχει συγγράψει μια βιβλίων ε, πολύ σημαντικών και θα μας δώσει μια εικόνα για τις συνθήκες, για το πώς μπορούμε να διαμορφώσουμε την κατάσταση και τις ευκαιρίες και τους κινδύνους και ο καθηγητής ε, Κίρ στην στο Πανεπιστήμιο του Σενγκάλεν στην Ελβετία και ε, βεβαίως ως οικονομολόγος έχει ασχοληθεί με τη σχέση δημοκρατίας και δημοσίων οικονομικών. Είναι Ελβετός, όπως είπα, και η Ελβετία έχει πολλά τέτοια μέσα. Π.χ. στην Ελβετία υπάρχει συγκεκριμένη μορφή φρένου χρέους. Υπάρχει το λεγόμενο δημοσιονομικό δημοψήφισμα στην Ελβετία και έχουν πολλές ιδιαιτερότητες οι Ελβετοί ψηφίζουν π.χ. για τους φόρους, για τις δημόσιες δαπάνες, αμέσως, αμεσοδημοκρατικά οι πολίτες. Και βεβαίω αυτοί και ακόμα και αυτοί οι οποίοι ε, θέλουν μεγαλύτερη συμμετοχή των, των πολιτών ε, συμφωνούν πως ένα πράγμα δεν πρέπει να αποφασίζουν οι πολίτες. Τους φόρους και τα οικονομικά, αλλιώ θα καταργηθούν οι φόροι και θα χρεοκοπήσει το κράτος. Η εμπειρία όμως στην Ελβετία δείχνει πως δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Γιατί οι πολίτες συχνά είναι πολύ πιο προσεκτικοί και λογικοί στο τι κάνουν τα λεφτά τους, τους φόρους δηλαδή. Ε, πιο λογικοί από τις κυβερνήσεις. Ίσως αυτός είναι ένας λόγος για τον οποίο μπορεί να μας ε, και θα πρέπει να ακούσουμε ιδιαίτερο ενδιαφέρον και προσοχή τον καθηγητή τον κύριο Κίρκεστα. Γιατί η κατάσταση στην Ευρώπη οφείλεται και στο ότι το δημόσιο, το κράτος, ε, κάποια κράτη έζησαν πολύ πάνω από τις δυνάμεις τους και ε, οδηγηθήκαμε σε αυτή την κρίση χρέους. Πρώτο λοιπόν θα ακούσουμε τον καθηγητή Τέο Σίλερ. Έχετε τον λόγο. Yeah. Thank you very much. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Μπορώ να μιλήσω γερμανικά, έτσι, δεν υπάρχει πρόβλημα. And, uh, ich werde mich, uh, recht stark an mein Thema... Και θα μείνω στο θέμα μας άμεση δημοκρατία στην Ευρώπη, συνθήκες, ευκαιρίες, προκλήσεις. Και θα μιλήσω για την κατάσταση στα κράτη-μέλη. Γιατί θεωρώ πως η κατάσταση αυτή και νομίζω αυτοί οι δύο όροι μπορεί να συνεισφέρουν στην άμεση δημοκρατία στο ευρωπαϊκό επίπεδο. Τώρα κάποιες γενικές παρατηρήσεις. Όλοι μιλάνε για τη δημοκρατία, την άμεση δημοκρατία ιδιαίτερα και βεβαίως πρέπει να ξεκινήσουμε την αρχή της λαϊκής κυριαρχίας. Κάθε σύνταγμα βασίζεται σε αυτήν. Όλες οι αποφάσεις πρέπει να νομοποιούνται από τη λαϊκή βούληση και να τηρούν τις αρχές ελευθερίας και της ισότητας. Βεβαίως δεν μπορούν για πρακτικούς λόγους να αποφασιστούν όλα απευθεία από το λαό, γι' αυτό χρειάζεται αντιπροσώπευση, αλλά οι πολίτες πρέπει να μπορούν να εκλέγουν και να ελέγχουν μέσω εκλογών τις διαδικασίες, τους αντιπροσώπους τους και βεβαίω θα πρέπει να μπορούν να τα ανακαλούν αυτά και αυτούς. Αυτό ισχύει για όλα τα επίπεδα, τοπικό, περιφερειακό, εθνικό και ευρωπαϊκό. Δεύτερον, πολιτικές διαδικασίες που ανταποκρίνονται σε αυτή την αρχή ε, υπάρχουν σε δύο μορφές. Αφενός δημοψηφίσματα που ε, γίνονται ad hoc με βάση μία απόφαση της κυβέρνησης του Κοινοβουλίου και αφετέρου θεσμοποιημένες διαδικασίες ε, που ορίζουν γενικώ την μορφή και την διεξαγωγή των δημοψηφισμάτων. Οπότε έχουμε το υποχρεωτικό ε, δημοψήφισμα ε, την πρωτοβουλία των πολιτών και την ε, πρωτοβουλία με βάση κάποιο θέμα με βάση το οποίο υποβάλλεται μια πρόταση τώρα για τα ad hoc δημοψηφίσματα και την θεσμοποίηση είναι πάρα πολύ σημαντικά αυτά γιατί είναι πολύ σημαντικά συγκεκριμένες καταστάσεις αλλά βεβαίως είναι μοναδικές αυτές οι περιστάσεις οι οποίες πιθανώς να προκύψουν μια φορά σε διάστημα δεκαετιών. Τώρα υπό ποιες συνθήκες υπάρχει μια θεσμοποίηση της άμεσης δημοκρατίας. Εδώ πέρα ιστορικά βρίσκουμε κάποιες συνθήκες που ευνοούν μια τέτοια θεσμοποίηση μπορεί να είναι σοβαρές ε, κοινωνικές ε, συγκρούσεις όπως τότε στην Ελβετία ή στο παρελθόν στις ΗΠΑ, δεύτερον ζητήματα ανεξαρτησίας όπως στην Ιρλανδία, τρίτον μια, ένας μετασχηματισμός του συστήματος ε, όπως η Γερμανία το 1919 η Ιταλία πιο πρόσφατα και βεβαίως ε, μεγάλες τιμικές κρίσεις όπως παραδείγματος χάρη στην Ισλανδία. Θα αναφέρω λοιπόν διάφορα βήματα. Θα σας δείξω ε, κάποιες διαφάνειες για τα δημοψηφίσματα ad hoc. Μετά θα κάνουμε μια γρήγορη παρουσίαση των διαφορετικών μορφών της αμεσοδημοκρατικής διαδικασίας. Μετά θα πάμε στο περιφερειακό και στο δημοτικό επίπεδο. Τέταρτον, θα δούμε το τι γίνεται στην πράξη στην άμεση δημοκρατία και κάποια συμπεράσματα, προκλήσεις και ε, εξέλιξη μελλοντική, κάτι το οποίο ονομάζω αναβάθμιση Τη άμεση δημοκρατία. Ελπίζω λοιπόν να λειτουργήσει. Στη διαφάνεια αυτή λοιπόν βλέπετε μία σύντομη έτσι, παρουσίαση των αποφάσεων ad hoc, δημοψηφίσματα. Εδώ πέρα είχαμε διαφορετικές βεβαίως συνθήκες ε, που έπαιξαν ρόλο, δηλαδή αφενός ανεξαρτησία, πολύ σημαντικό βεβαίως, για τα δημοψηφίσματα, η Ιρλανδία, οι Βαλτικές χώρες, η Σλοβενία το 1991, κατόπιν η μετάβαση στη δημοκρατία π.χ. Ελλάδα, η Ιταλία όταν ψήφισε ο κόσμος για τη μοναρχία ή την δημοκρατία, η Ισπανία 76 και 78 και Ανατολική Ευρώπη 1991 και εξή. Μετά βασικά συνταγματικά ζητήματα όπως η μετάβαση στην Πέμπτη Δημοκρατία στη Γαλλία το 1958 τα πάρα πολλές αποφάσεις ένταξης στην ευρωπαϊκή κοινότητα και στο ευρώ. Αναφέρονται οι χώρες που έκαναν δημοψήφισμα και τέλος η περιφερειακή αυτονομία όπως στην Ισπανία αλλά και στο Ηνωμένο Βασίλειο. Και υπάρχουν και κάποιες ε, συγκρούσεις ε, εσωτερικές ε, π.χ. στη Σουηδία κρίθηκε το ζήτημα της πυρηνικής ενέργειας στην Πορτογαλία το ζήτημα της έκτρωσης και στον Ηνωμένο Βασίλειο προσφάτως η εκλογική νομοθεσία Ε, ε. Ja, auf dieser Folie ist äh, in aller Kürze aufgeführt. Εδώ πέρα σε αυτή τη διαφάνεια βλέπουμε εν συντομία τα διάφορα άμεσο δημοκρατικά μέσα που χρησιμοποιούνται στα διάφορα κράτη-μέλη. Έχουμε υποχρεωτικά δημοψηφίσματα στη Δανία, Εσθονία και Ιρλανδία που το χρησιμοποιούν αυτό το μέσο και σε κάποιες άλλες χώρες μετά υπάρχει δημοψήφισμα από τις αρχές του κράτους όπως στην Αυστρία, Δανία, Λουξεμβούργο, Μάλτα, Πορτογαλία. Μετά υπάρχει η πρωτοβουλία των πολιτών. Βουλγαρία, Ουγγαρία, Ιταλία, Λετωνία, Λιθουανία, Σλοβακία, Σλοβενία και υπάρχει και η πρωτοβουλία των πολιτών, όπως λέμε η Ευρωπαϊκή, με βάση ένα θέμα, Αυστρία, Πολωνία, Ισπανία και κάποιες άλλες χώρες που το έχουν ως μια δευτερεύουσα επιλογή. Οπότε τώρα βλέπουμε τα μέσα και τις χώρες ε, στις οποίες ε, χρησιμοποιούνται. Auf der Στο επίπεδο της περιφέρειας και του Δήμου, θέλω να αναφέρω κάποια παραδείγματα, ο Γκέρατ Χέφνερ ανέφερε κάποια, ενώ η Ελβετία έχει σε περιφερειακό επίπεδο, στα καντόνια δημοψηφίσματα και στο επίπεδο του Δήμου, στις ε, χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά κανόνα δεν συμβαίνει κάτι τέτοιο. Εντός της Ευρωπαϊκή Ένωσης ε, κάποιες χώρες έχουν τέτοια διάρθρωση. Στη Γερμανία έχουν πρωτοβουλίες ε, και δημοψηφίσματα κάποιες ε, χώρες, αλλά με περιορισμούς πάρα πολλούς. Είχαμε τέτοια Δημοσφίσματα στο Βερολίνο, το Αμβούργο και αλλού. Σε κάποιες αυτόνομες περιοχές ε, της Ισπανίας επίσης γίνεται κάτι τέτοιο, ειδικά στην προστασία του περιβάλλοντος. Επίσης στην Αυστρία, Ιταλία, Ισπανία και Πολωνία δεν παίζουν ιδιαίτερο ρόλο αυτά τα δημοσφίσματα. Στην πολιτική των Δήμων από το 1990 η Γερμανία έχει μια σημαντική εξέλιξη πρωτοβουλειών και δημοψηφισμάτων και υπάρχει σε όλα τα κρατήδια. Σε κάποια κρατήδια με πιο φιλελεύθερους κανόνες. Χρησιμοποιούνται αυτά για πάρα πολλά θέματα. Στη Βαβαρία, Αμβούργο, Έση, Βόρεια Βεσφαλία. Συνολικά στη Γερμανία ε, είχαμε 6.000 πρωτοβουλίες και 3.000 αποφάσεις των πολιτών. Στην Πολωνία επίσης χρησιμοποιείται το δικαίωμα της πρωτοβουλίας, κυρίως για ανάκληση το του Δημοτικού ε, Συμβουλίου συνήθως ή τοπικού κοινοβουλίου. Επίσης στην Τσεχία παίζει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο αυτό στην προστασία του περιβάλλοντος. Πάρα πολύ περιοριστικοί κανόνες προφανώς οδηγούν σε μικρή χρήση σε Γαλλία, Ιταλία, Βουλγαρία, Ισπανία, σε χώρες όπως Φιλανδία και η Σουηδία μέχρι πρόσφατα υπήρχαν μόνο δημοψηφίσματα με χαρακτήρα συμβουλευτικό και αφορούσαν ζητήματα συγκοινωνιών ή συγχώνευσης δήμων. Σε χώρες ε, με συχνή πρακτική, οι τοπικές ε, πρωτοβουλίες ε, οδήγησαν σε αναζωογόνηση της τοπικής δημοκρατίας. Πολλές αποφάσεις, λόγω της καλής τους ποιότητας, εκτιμώνται ιδιαίτερα και ενεργοποιήθηκαν έτσι και τοπικοί φορείς λήψης αποφάσεων. Τέταρτον, για την πρακτική της άμεσης δημοκρατίας στο εθνικό επίπεδο. Και μάλιστα στο πλαίσιο μιας θεσμοποιημένης διαδικασίας. Το υπόδειγμα της Ελβετίας βεβαίως δεν επιτυχάνεται πουθενά εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συνολικά στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπάρχουν λίγα τέτοια δημοψηφίσματα θεσμοποιημένα και επικεντρώνονται σε λίγες χώρες. Υποχρεωτικά δημοψηφίσματα κυρίως γίνονται στην Δανία και την Ιρλανδία, κυρίως όσον αφορά ζητήματα εκχώρησης κυριαρχίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και εκεί πέρα καμιά φορά γίνονται και διπλά επαναλαμβάνονται. Στην Ιρλανδία επίσης υπάρχουν προβλήματα με τις αξίες της κοινωνίας και τις συγκρούσεις προκύπτουν γιατί υπάρχουν αυτά τα πράγματα στο Σύνταγμα και κάθε αλλαγή του Συντάγματος πρέπει να περάσει από δημοψήφισμα. Πρωτοβουλίες για... λαμβάνονται κυρίως στην Ιταλία με 70 περίπου ψηφοφορίες από το 1974 μέχρι τώρα κυρίως λόγω του κομματικού, του πολυκομματικού συστήματος. Επειδή τώρα απαιτείται μια συμμετοχή των ψηφοφόρων ε, κατά 50% και πάνω για να είναι έγκυρο το δημοψήφισμα. Γύρω στα μισά από αυτά ήταν έγκυρα. Από το 1997 μέχρι το 2010 δεν υπήρχε ούτε ένα έγκυρο. Όμως αποκτά η δημοκρατία. απέκτησε σε τρεις φάσεις ε, μεγάλη σημασία. Στη δεκαετία του 1970 υπήρχαν ζητήματα ηθικής, τα οποία κρίστηκαν προς την κοσμική πλευρά, όπως παραδείγματο, χάρη το διαζύγιο. Δεύτερον, στην κρίση του πολιτικού συστήματος της Ιταλίας αρχές της δεκαετίας του 1990 έγιναν δημοψηφίσματα για τις μεταρρυθμίσεις της εκλογικής νομοθεσίας που οδήγησαν σε μεταμόρφωση του συστήματος. Και τρίτον, τον Ιούλιο του 2011 επιτάχυναν τέσσερα έγκυρα δημοψηφίσματα την πτώση του συστήματος Μπερλουσκόνη, μεταξύ άλλων ε, μέσω απόρριψης της ποινική του ασυλίας και διάφορων άλλων σημαντικών αποφάσεων. Σε αυτές τις καταστάσεις κρίσης ενεργοποιήθηκε η άμεση δημοκρατία και η λαϊκή κυριαρχία θα λέγαμε. σε πολλά κράτη-μέλη της Ανατολικής Ευρώπης, Λιθουανία, Λετωνία, Σλοβενία έγιναν πολλές τέτοιες προσπάθειες, κυρίως όσον αφορά τις κοινωνικές συνέπειες της πτώσης του κομμουνισμού. Με μικρή επιτυχία όμως, κυρίως λόγω των περιοριστικών κανόνων στην Ουγγαρία, ε, θα έλεγα πως ε, δόθηκε νέα δυναμική στη σύγκρουση των κομμάτων και επιδεινώθηκε, θα έλεγα, η ε, κατάσταση καθώς διπλασιάστηκε ο αριθμός των ε, συμμετεχόντων σε ένα δημοσίσμα για να είναι αυτό έγκυρο πήγε από το 25% στο 50%. Ε, Επίση, από ό,τι φαίνεται στις υπόλοιπες χώρες είτε δεν υπάρχουν δημοσίσματα είτε είναι πολύ περιοριστικοί οι κανόνες και δεν εξαντλείται έτσι η συμμετοχική δημοκρατία. και ε, σε λίγες μόνο περιπτώσεις υπήρχε ένα χρήσιμο και ποιοτικό αποτέλεσμα. Χρειάζονται όμως αυτά για να αναπτυχθεί μια πολιτική κουλτούρα άμεσης δημοκρατίας. Και, σύντομα τώρα περνάω στο τελευταίο μου σημείο, για κάποιες προκλήσεις της άμεσης δημοκρατίας και την αναβάθμισή της. Προκύπτει λοιπόν πως η άμεση δημοκρατία έχει μεγάλο δυναμικό, αλλά σε πολλές χώρες δεν χρησιμοποιείται με βέλτιστο τρόπο. Έχουμε λοιπόν την εισαγωγή της διαδικασίας η οποία αποτελεί μια μεγάλη πρόκληση. Μια τέτοια αναβάθμιση θα ήθελα να αναφέρω και εδώ πέρα αναφέρομαι σε όλα τα επίπεδα τοπικό, περιφερειακό και εθνικό. Πρώτον, πολλά κράτη-μέλη δεν έχουν ακόμα την δυνατότητα άμεσης δημοκρατίας σε τοπικό επίπεδο, παρά το ότι είναι εδώ πέρα η σημαντικότερη δημοκρατική εμπειρία των χωρών. Αναφέρω. Ε, Δανία, Πολωνία και Βαλτικές χώρες που θα πρέπει επιγόντως να αποκτήσουν τέτοιους ε, κανονισμούς. Ε, επίσης δύσκολη είναι η σε Βουλγαρία, Ιταλία, Ισπανία, και άλλες χώρες τα θέματα τα οποία επιτρέπονται ε, όπως επίσης το ότι ε, βεβαίως πρέπει να είναι και χαμηλή η απαρτία που θα οριστεί. Όλα αυτά είναι απαραίτητα. Ε, το Συμβούλιο της Ευρώπης έχει κάνει κάποιες συστάσεις για την εισαγωγή της άμεσης δημοκρατίας στο τοπικό επίπεδο. Κατόπιν, σε Ισπανία και Αυστρία τα κρατήδια θα πρέπει να αναπτύξουν την διαδικασία αυτή για να περάσουν στην πλήρη πρωτοβουλία των πολιτών. Στη Γαλλία επίσης θα πρέπει να απομακρυνθούν από την κουλτούρα του δημοσίσματος που προκαλεί η κυβέρνηση. Και σε άλλες χώρες είναι πολύ περιοριστική η Συνολικά θα μπορούσαμε να συστήσουμε πως το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο των Περιφερειών θα πρέπει να ασχοληθεί με αυτό το ζήτημα. Συνολικά, λοιπόν, δεν έχει αναπτυχθεί πλήρως η άμεση δημοκρατία στο τοπικό επίπεδο. Δεν, δεν υπάρχει δε καθόλου στο Βέλγιο, Γερμανία, Φιλανδία, Μάλτα, Ολλανδία, Σουηδία, Τσεχία, Ηνωμένο Βασίλειο και Κύπρο. Το μίνιμουμ εδώ πέρα θα ήταν το επόμενο βήμα. Δηλαδή τουλάχιστον η εισαγωγή μιας πρωτοβουλίας με βάση μια ατζέντα. Δηλαδή στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα μπορούσε να υπάρξει κάτι τέτοιο, αλλά πώς να υπάρχει όταν δεν υπάρχει καν δυνατότητα στα κράτη-μέλη. Κάποιες χώρες έχουν μόνο διαδικασίες ε, δημοψηφίσματος τα οποία μπορεί να ξεκινήσει μόνο η κυβέρνηση, κοινοβούλιο κτλ. Παραδείγματος χάρη Δανία, Εστονία, Γαλλία, Ιρλανδία, Λουξεμβούργο, Πορτογαλία. Και εκεί πέρα δεν υπάρχει χώρος βεβαίως για να εκδηλωθούν οι πολίτες. Ένα πρώτο βήμα εδώ πέρα θα μπορούσε να είναι τουλάχιστον η εισαγωγή της πρωτοβουλίας αυτής με κάποια ατζέντα. Κατόπιν. Κάποιε χώρες έχουν πολύ περιοριστικούς κανόνες, ε, Λιθουανία, Λετωνία, Σλοβακία παραδείγματο χάρη, που ε, επιτρέπουν πολύ περιορισμένη χρήση για την Ιταλία και την Ουγγαρία, τα ανέφερα ήδη. Μία άλλη εξέλιξη, βεβαίως, ε, σημειώνεται σε Αυστρία, Ισπανία, Πολωνία καθώς μπορούμε να οδηγηθούμε από την πρωτοβουλία σε ένα δημοψήφισμα και βεβαίω ξεκινήσει κάτι τέτοιο ως συζήτηση η αστρία. Τέλος, θα πρέπει να ε, συζητηθούν οι διαδικαστικοί κανόνες για να είναι δίκαιοι και να μην υπάρχει δυνατότητα επηρεασμού από τα ΜΜΕ και τα μεγάλα οικονομικά συμφέροντα εδώ πέρα. Απαιτούνται κανόνες διαφάνειας και δήλωση των μεγάλων δωρεών. Οπότε θα έλεγα πως είναι υπαναπτυκτή η τοπική αυτή άμεση δημοκρατία σε αρκετά κρατημέλη, αλλά μπορεί να συνεισφέρει δύο βασικά πράγματα. Με τις πρωτοβουλίες μπορούν οι πολίτες να επαναφέρουν παραμελημένα θέματα και δεύτερον υπάρχει η δυνατότητα του κάθε πολίτη να οδηγήσει σε μια δημόσια συζήτηση με μεγαλύτερη ένταση συχνά να αυξήσει το πολιτικό ενδιαφέρον και να ξεκινήσει έτσι μια διαδικασία πολιτικής ε, εκμάθησης. Και βεβαίως στην Ευρωπαϊκή Ένωση η οποία θέλει να αυξήσει την συμμετοχή των πολιτών θα πρέπει να αυξήσει το ενδιαφέρον για την κουλτούρα της συμμετοχικής δημοκρατίας σε όλα τα κράτη-μέλη. Ευχαριστώ πάρα πολύ ευχαριστώ, κύριε Σούλα. Να παρακαλέσω και τον κύριο Γκέρχατ και να αναμιλήσει. Σας παρουσίασα ήδη. Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Είναι βεβαίως ε, ασυνήθιστο κάποιος να έρχεται εδώ πέρα από μη κράτος μέλος και να μιλάει για τον δημοκρατισμό της Ένωσης. Βεβαίως τίθεται το ζήτημα της σχέσης μεταξύ άμεσης δημοκρατίας και δημοσίων οικονομικών και υπάρχει ο γνωστός φόβος πως εάν αφήνει κάποιος τους ε, πολίτες να αποφασίσουν θα ψηφίσουν υψηλότερα έξοδα και χαμηλότερους φόρους και θα καταστραφούν τα δημόσια οικονομικά. Και για τον λόγο αυτό, παραδείγματο χάρη στη Γερμανία, σε όλα τα συντάγματα των κρατηδίων υπάρχει παραδείγματο χάρη η λεγόμενη οικονομική επιφύλαξη. Δηλαδή, αν υπάρχουν στοιχεία άμεσης δημοκρατίας, είναι διαμορφωμένα έτσι ώστε ζητήματα που έχουν οικονομικές επιπτώσεις δεν μπορούν να τεθούν. Βεβαίως το ζήτημα είναι αν δικαιολογείται αυτή η επιφύλαξη. Δεν υπάρχει κάποια τέτοια περίπτωση, αλλά μπορούμε νομίζω να συγκρίνουμε την Γερμανία με την Ελβετία. Στην Ελβετία οι πολίτες μπορούν σε όλα τα επίπεδα, σε διαφορετικό μέτρο, αλλά μπορούν να ψηφίσουν για οικονομικά ζητήματα. Δεν υπάρχει δηλαδή η γερμανική αυτή διάταξη. Παρ' όλα αυτά, κανένα ελβετικό καντόνι, ούτε και τα χρεωμένα, δεν έχει βρεθεί σε κατάσταση ε, χρεοκοπίας όπως το Ζάρλαντ και η Βρέμη παραδείγματο χάρη στη Γερμανία. Και συχνά είναι σε καλή κατάσταση τα οικονομικά. Ένα δεύτερο παράδειγμα, εάν δείτε την κρίση, η Ελβετία το 2008, στην κρίση δηλαδή, συνολικά είχε αποφασίσει τρία προγράμματα κινητοποίησης ε, της οικονομίας και τηρήθηκαν παρόλα αυτά τα όρια του χρέους το οποίο αποφασίστηκαν το 2001 με, δύο, με πλειοψηφία δύο τρίτων πέρασε μια μεταβατική περίοδος και ισχύουν από το 2007 τα δε γερμανικά όρια για το χρέος που αποτελούν σήμερα πρότυπο για αυτά τα οποία συζητιούνται στην Ευρώπη είναι ε, αντιγραφή του ε, ελβετικού συστήματος. Και διαπιστώνουμε πως το 2009 είχαμε πλεόνασμα στον προϋπολογισμό. Ενώ οι άλλες χώρες είχαν τεράστια ελλείμματα, εμείς χάρη σε αυτό το όριο χρέους, το οποίο υπενθυμίζω το υπερψήφισε ο λαός, είχαμε ε, πλεόνασμα. Βεβαίως, βασική ουσία, βασική αιτία ήταν βεβαίως πως έχουν κυριαρχία όσον αφορά τους φόρους τα καντόνια, κατά οποίο όμως και για τις ε, χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επίσης μπορούμε να συγκρίνουμε με τις Ηνωμένες Πολιτείες όπου έχει αποδειχθεί πως η άμεση δημοκρατία πριν τον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο είχε οδηγήσει σε ε, άνοδο των ε, φόρων ενώ μετά το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο το αντίθετο οπότε συμβαίνουν και τα δύο βεβαίως υπάρχει και η ε, πρόταση 13 που πέρασε στην Καλιφόρνια που αυτή τη στιγμή στραγγαλίζει τα δημόσια οικονομικά της πολιτείας αλλά αυτό οφείλεται και σε κομματικές συγκρούσεις αν δούμε λοιπόν την άμεση δημοκρατία σε οικονομικά ζητήματα Πρέπει να υπάρχει ένα υπόβαθρο, δεν αρκεί απλά να μιλάμε για αυτήν και υπάρχει ε, ένα πρόβλημα που είναι ιδιαίτερο στη γερμανική συζήτηση, πως η άμεση δημοκρατία σε αυτά τα ζητήματα περιορίζεται λίγο πολύ ε, στο επίπεδο της πρωτοβουλίας. Γιατί υπάρχει ο φόβος και όχι στο επίπεδο του δημοψηφίσματος. Οπότε πρέπει να δούμε ποια μέσα υπάρχουν στη διάθεση των πολιτών, ποια επίδραση έχουν στα δημόσια οικονομικά και η πρωτοβουλία βεβαίως εδώ πέρα είναι υποδεέστερη σε σχέση με το δημοψήφισμα. Δεν είναι δημοψήφισμα. Συχνά τα μπερδεύουμε γιατί λέμε πως δημοψήφισμα είναι κάτι το οποίο προκαλεί το κοινοβούλιο ή η κυβέρνηση και ο κόσμος μπορεί να πει μόνο ή όχι μόνο ναι όχι. Αλλά βλέπουμε πως υπάρχει στην Ελβετία το λεγόμενο οικονομικό δημοψήφισμα, δυστυχώς μόνο σε επίπεδο καντονιού και δήμου, όχι σε επίπεδο χώρες. Κυρίως αφορά μεγάλα έργα υποδομών, παραδείγματος χάρη ένα πανεπιστήμιο το οποίο πρέπει να ανακαινιστεί, ε, τότε πρέπει να το αποφασίσει αυτό ο λαός. Εκεί πέρα λοιπόν υπάρχουν διαφορετικές ε, αποφάσεις, ε, δηλαδή συχνά τα όρια είναι χαμηλότερα και εξαρτώνται από το ποσό ή μπορεί να είναι τα ποσά μεγαλύτερα και να δοθούν άπαξ. Εκεί πέρα τότε είναι και τα όρια υψηλότερα του δημοψηφίσματος και μπορεί να είναι το ε, δημοψήφισμα υποχρεωτικό ή προαιρετικό ή και τα δύο. Έχουμε όλα τα συστήματα στα ελβετικά καντόνια. Στο δικό μας καντόνι, το Σενγκάλεν, έχουμε και τα δύο. Δηλαδή όταν είναι επαναλαμβανόμενες οι δαπάνες από 300.000 φράγκα και πάνω είναι προαιρετικό το δημοψήφισμα και από το 1,5 εκατομμύριο φράγκα και πάνω είναι υποχρεωτικό. Αν γνωρίζετε βεβαίως πως ο προπολογισμό είναι 4 δισεκατομμύρια φράγκα το χρόνο. Βλέπετε πως είναι πολύ χαμηλό το όριο και χρειάζονται 4.000 υπογραφές για ένα προαιρετικό δημοψήφισμα. Οπότε είναι πάρα πολύ χαμηλή η απαρτία και δεν ε, χρειάζεται επίσης απαρτία για τη συμμετοχή. Οπότε είναι ένα πάρα πολύ εύκριστο μέσο και βεβαίως μπορούν μόνο να μειωθούν και όχι να αυξηθούν τα έξοδα με το οικονομικό δημοψήφισμα, οπότε είναι ένα μέσο σταθεροποίησης των δημοσίων οικονομικών και όχι το αντίθετο. Το δεύτερο και σημαντικότερο μέσο είναι το νομοθετικό δημοψήφισμα προαιρετικό που υπάρχει και σε ε, ομοσπονδιακό και σε επίπεδο καντονιού, δηλαδή κάθε νόμος μπορεί να ανατραπεί με ένα νομοθετικό δημοψήφισμα και αυτό είναι σημαντικό γιατί το οικονομικό δημοψήφισμα γίνεται μόνο όταν ενεργοποιούνται δαπάνες που δεν αναφέρονται σε κάποιο νόμο δύο όπως είπα μεγάλες υποδομές ε, σε ομοσπονδιακό επίπεδο ή στρατιωτικές δαπάνες ε, που συζητιούνται αυτό τον καιρό στην Ελβετία για την αγορά εννέα, ε, νέων μαχητικών αεροσκοφών. Και βεβαίως είναι σημαντικά θα στο επίπεδο το Ομοσπονδιακό και το νομοθετικό δημοψήφισμα λαμβάνει χώρα όταν εκδίδονται νέοι νόμοι και έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία για τα δημόσια οικονομικά, ε, όπως είπα, όταν αφορά νόμους με δημοσιονομικό αντίκτυπο. Και εδώ πέρα ακριβώς τι συμβαίνει. Μπορεί βεβαίως να απορρίψουν κάποιον νόμο οι πολίτες ο οποίος προβλέπει δαπάνες αλλά μπορεί να απολύψουν και ένα νόμο ο οποίος προβλέπει κάποιες ε, εξοικονομήσεις. Αλλά γενικά οι Ελβετοί πολίτες είναι συντηρητικοί στα οικονομικά. Και το έχουμε δει αυτό σε πάρα πολλές ε, ψηφοφορίες της δεκαετίας του 80 και του 90. Οπότε δεν υπάρχει κίνδυνος εκτροχιασμού από αυτά τα δημοσίσματα. Βέβαια, από την άλλη πρέπει να δούμε πώς σε μια τέτοια κατάσταση λογικό είναι να υπάρχουν επιπλέον μέσα, όπως είπα, το όριο αυτό του χρέους κτλ. Για το υποχρεωτικό συνταγματικό δημοψήφισμα ισχύει το ίδιο. Οπότε ε, έχει και τελείως ε, διαφορετική σημασία βεβαίως. Κάπω διαφορετική τώρα είναι η πρωτοβουλία, γιατί οι διάφορες πρωτοβουλίε είναι κάτι το οποίο ε, μπορούν να κάνουν ε, όλα τα, τα κανόνια. Ε, όχι η Ομοσπονδία. Οι πρωτοβουλίε κατά κανόνα βεβαίως αφορούν κάποιες δαπάνες και υπάρχει ένας κίνδυνος ο οποίος είναι το εξής. Ε, κατά τα 90% απορρίπτονται οι πρωτοβουλίες, οπότε βασικός στόχος τους είναι να τεθεί ένα ζήτημα στην ημερήσια διάταξη. Συνήθως κάνει μια αντιπρόταση το Κοινοβούλιο, οπότε γίνεται κάτι στην πράξη, ακόμα και αν απορρίπτεται η ε, πρωτοβουλία αυτή. Κλασικό παράδειγμα η πρωτοβουλία για την ε, κατάργηση του στρατού που οδήγησε σε ριζική αλλαγή της πολιτικής άμυνας. Και ψήφισαν βεβαίω ε, μόνο το μόνο, όπως λένε, το 1 τρίτο, και 35% υπέρ, παρά το δεν το περίμενε κανείς αυτό από τους Ελβετούς. Οπότε η ένωση αυτή για την ε, κατάργηση του ελβετικού στρατού έφερε άλλη μια πρωτοβουλία για να μην αγοραστούν ε, μαχητικά αεροπλάνα. Και αυτή δεν πέρασε, αλλά όπως είπα και οι πρωτοβουλίες αυτές ε, οδηγούν σε, κάποια, σε κάποιο μετριασμό της στάσης θα έλεγα. Βεβαίως θα πρέπει να πούμε πως σε επίπεδο καντονιού πως χρειάζεται ένα όριο του χρέους και κλασικό παράδειγμα όπως είπα είναι το Σενγκάλεν το οποίο έχει από, την, ε, από το 1989 ένα τέτοιο κανονισμό και λειτουργεί ως εξής. Μπορεί να ξοδέψει και να δανειστεί το κράτος, αλλά αυτό μόνο αν υπάρχουν προσδοκόμενα έσοδα. Αλλιώς επί της αρχής θα πρέπει να γίνονται οικονομίες, εκτός εάν υπάρχει πλεόνασμα. Εάν λοιπόν υπάρχει έλλειμμα, αυτομάτως οδηγούμαστε σε οικονομίες. Ε, αν υπάρξει ξανά πλεόνασμα, υπάρχει, ε, κάποια, υπάρχει ε, περαιτέρω αύξηση των δαπανών. Έχουμε δηλαδή έναν αυτόματο, θα έλεγα, σταθεροποιητή. Το αποτέλεσμα είναι το εξή. Εμεί είμαστε ένα σχετικά φτωχό καντόνι, είμαστε στη 19η ε, θέση από τα 26 καντόνια, αλλά δεν έχουμε χρέος. Ε, Πλέον με ελάχιστους ε, τόκους και κάθε χρόνο έχουμε πλεόνασμα και όχι καινούριο χρέος. Οπότε, ε, επί της αρχής είναι απλή η ρύθμιση αυτή. Με τα δημοψηφίσματα δαπανών ε, ρωτάμε τον κόσμο εάν θέλει κάποια δαπάνη και μετά γνωρίζουν βεβαίως ότι θα πρέπει να τα πληρώσουν και όλα αυτά τα οποία εγκρίνουν. Και νομίζω λειτουργεί καλά αυτό το σύστημα. Εάν το δούμε τώρα σε όλα τα καντόνια, κάναμε μια έρευνα για τις τελευταίες δύο δεκαετίες και είδαμε πώς λειτουργεί το σύστημα. Το όριο αυτό του χρέους οδηγεί συχνά σε αύξηση των ε, εσόδων, μείωση των δαπανών, οπότε τα καντόνια τα οποία έχουν όριο χρέους έχουν πολύ χαμηλότερο χρέος συνολικά με τους Δήμους. Επίσης υπάρχει άμεση δημοκρατία σε οικονομικά ζητήματα. Βεβαίως φαίνεται κάποιοι έχουν υποχρεωτικά οικονομικά ε, δημοψηφίσματα και έχουν κατά κανόνα 25% χαμηλότερο χρέος. Οπότε οδηγεί αυτό σε μια δημοσιονομική σταθερότητα. Βεβαίω διαφέρει η κατάσταση σε ομοσπονδιακό επίπεδο. Εκεί πέρα δεν υπάρχει οικονομικό δημοψήφισμα, δεν υπάρχει επίση αυτόματη προσαρμογή των φόρων. Οι φόροι πρέπει να ψηφιστούν, εάν πρέπει να ανέβουν και οι σημαντικότεροι φόροι π.χ. ο ΦΠΑ ε, αναγράφονται στο Σύνταγμα, οπότε δεν ε, αλλάζουν τόσο απλά, πρέπει να αλλάξει το Σύνταγμα και εκεί πέρα είναι υποχρεωτικό το δημοψήφισμα και βεβαίως ε, εντάξει, είναι διαφορε... λειτουργεί διαφορετικά. Το κράτος εκτιμά τα έσοδά του και αναλόγως κινείται. Βεβαίως, αυτή τη στιγμή από την αρχή της δεκαετίας του 90 μέχρι γύρω στο 2004 το χρέος της Ομοσπονδίας, του Ομοσπονδιακού κράτους ανέβηκε πάρα πολύ Βεβαίω από το 2005 κατέβηκε πάλι πολύ, αλλά δεν έχουμε φτάσει ακόμα στα επίπεδα του 1990. Και Βεβαίω, ο κόσμο δεν είναι διατεθειμένο να δεχτεί εύκολα αυξήσει φόρων, θα έλεγε κανεί. Αλλά στην πραγματικότητα δεν ισχύει αυτό. Το 1993 ο κόσμο υπερψήφισε και την εισαγωγή του ΦΠΑ αλλά και την αύξηση του ποσοστού του τότε κατά 1% κοντά στο 7% για να πάει στο συνταξιοδοτικό σύστημα και ταυτόχρονα ε, υπερψήφισαν την αύξηση του ειδικού φόρου στα πετρελαιοειδή για έργα υποδομής. Πριν από δύο χρόνια υπερψήφισαν μια προσωρινή αύξηση του ΦΠΑ για να πάει στην ασφάλιση αναπήρων. Οπότε, εάν ξεκαθαρίζει κανείς τους πολίτες πως τα έσοδα αυτά χρειάζονται, είναι διατεθειμένοι κατά πλειοψηφία να τα υπερψηφίσουν. Χρειάζεται διάλογος βεβαίως, αλλά γίνεται αυτός ο διάλογος ε, για να ληφθεί μια απόφαση. Αν ε, η απόφαση αυτή απλά λαμβάνεται από το κράτος, δεν υπάρχει καθόλου διάλογος. Και βεβαίως αυτό το οποίο θα σας ε, εκπλήξει είναι πως αυτή τη στιγμή η Ομοσπονδία λειτουργεί με κάποιες προθεσμίες. Δηλαδή, μέχρι ένα χρονικό σημείο μπορεί να επιβάλλει φόρους και μετά ξαναυποβάλλεται αυτός πολίτες που πρέπει να το εγκρίνουν. Βεβαίω μπορεί να μην το εγκρίνουν και να χρειαστεί να επανυποβληθεί, αλλά κατά, κανόνες, ε, κατά κανόνα λειτουργεί. Το 2004 είχαμε τελευταία ψηφοφορία και εκεί χωρί προβλήματα. Η αναγκαιότητα αυτή λοιπόν του να υπερψηφίζονται οι δημόσιες δαπάνες οδηγεί σε εντατικέ συζητήσεις για το εάν και ποιου φόρους πρέπει να επιβάλλουμε και να αλλάξουμε. Οπότε υπάρχει, ε, αν θέλετε, ένας καταναγκασμός να συζητιούνται αυτά τα πράγματα δημόσια. Και τέλος, θα μπορούσε κάποιος να σκεφτεί, να προσπαθήσει με πρωτοβουλίες να μειώσει τον φόρο. Πριν από 20 χρόνια υπήρξε μια προσπάθεια να περάσει μια πρωτοβουλία το ο άμεσος ομοσπονδιακός φόρος εισοδήματος να καταργηθεί και να έχουν το δικαίωμα μόνο τα καντόνια. Όπως ήταν ε, αρχικά στην ε, ιστορία της Ομοσπονδίας μας το, γύρω στο 1850 γιατί ο άμεσος ομοσπονδιακός φόρος είναι εμφανίστηκε από τον 20ο αιώνα μάζεψε ο κόσμος υπογραφές δεν ξέρω αν έφτασαν τις 100.000 αλλά δεν ε, έθεσαν το ερώτημα ενώπιον του λαού γιατί ήταν ξεκάθαρο πως θα απορρίπτονταν δεν είχε δηλαδή καμία προοπτική. Οπότε δεν πρέπει να υποτιμάμε την λογική των πολιτών όσον αφορά και τα δημόσια οικονομικά. Βεβαίως δεν πάει το κάθε δημοψήφισμα όπως θα το ήθελα εγώ, αλλά το ίδιο ισχύει και για την κοινοβουλευτική δημοκρατία. Εάν δείτε την ιστορία μας, νομίζω θα δείτε πως υπάρχει μια εμπειρία οικονομικών αποφάσεων με την άμεση δημοκρατία. Δεν υπάρχει μόνο η Καλιφόρνια. Εάν το διαχειριστεί κανείς λογικά, νομίζω πως και οι αντιδράσεις είναι λογικές και αυτό οδηγεί σε υγιή δημόσια οικονομικά και βιώσιμα δημόσια οικονομικά καλύτερα από αυτά τα οποία γνωρίζουμε συνήθως από την αντιπροσωπευτική δημοκρατία. Ευχαριστώ. ganz herzlichen Dank. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Κύριε Κύρχη Γκέσνα, τηρήσατε το, και το χρόνο. Θέλω να σε επενέσω εδώ πέρα. Τώρα υπάρχει δυνατότητα ερωτήσεων. Okay. Uh, thank you very much. As... Ε, Ευχαριστώ πάρα πολύ. Με τιμή να αναλάβω την Προεδρία. Ο κύριος Μπρόνσα είναι ο πρώτος που έχει το λόγο. Και μετά η Έμιλη. Η Έμιλη Ρέγνερ. Ευχαριστώ πολύ. Ο καθηγητής Σίλερ ανέφερε τα ad hoc δημοψηφίσματα και τα διαφοροποίησε από αυτά τα οποία προβλέπει το Σύνταγμα, η νομοθεσία. Και βέβαια το πρόβλημα με τα ad hoc δημοψηφίσματα είναι ότι είναι ουσιαστικά στα χέρια τη κυβέρνηση αποκλειστικά που μπορεί να αποφασίσει κατά πόσον διεξάγει ή δεν διεξάγει δημοψήφισμα, ανάλογα με το αν είναι πιθανό να τα κερδίσει και πότε είναι πιο πιθανό να τα κερδίσει. Το δημοψήφισμα του, 1975 στο Ηνωμένο Βασίλειο είχε χαρακτηριστεί ως ενταξιακό. Δημοψήφισμα δεν ήταν βέβαια, διότι προσχώρησε το 72, βέβαια με ισχύ το 73 και το δημοψήφισμα διεξήχθη το 1975 για το αν πρέπει να αποχωρήσει ή όχι από την ε, τότε κοινότητα. Βέβαια έγινε αυτό το δημοψήφισμα, αλλά ποιον ε, ε, στόχο είχε να παραμείνει το status quo. Αυτό ήθελαν ε, οι συντηρητικοί. Και υπήρξε και μία ε, έντονη προπαγάνδα 20 πλάσια ναι σε σχέση με το όχι. Αυτό ήταν το αποτέλεσμα. Εκεί δεν υπήρξε κάποια περιστολή δαπανών. Βέβαια το 2000 ε, μας υποσχέθηκαν ότι θα έχουμε δημοψήφισμα και για τη συνταγματική συνθήκη. Όπως όμως σε ερώτημα που έθεσα στη Σουηδική Προεδρία το 2009, όπως παραδέχτηκε λοιπόν η Σουηδική Προεδρία, τα ονόματα άλλαξαν. Τίποτα άλλο όμως, ή ελάχιστα άλλα άλλαξαν. Ουσιαστικά συσκευάστηκε σε άλλο πακέτο ε, μεταρρυθμιστική συνθήκη που μετέπειτα, μετέπειτα έγινε συνθήκη της Λισαβόνας. Βέβαια, Πάντοτε είναι προβληματικά τα επαναλαμβανόμενα ε, δημοψηφίσματα. Είδαμε ότι επαναλήφθη για το Μάστριχτ από τη Δανία το δημοψήφισμα, αλλά η ψήφος, ναι, στο Μάστριχτ ε, η από τη Γαλλία ήταν πολύ μικρή διαφορά. Δεν ζήτησε κανεί όμω να γίνει ξανά το δημοψήφισμα. Διερωτώ με για ποιο λόγο. Στην Ιρλανδία όμω έγινε ε, επαναληπτικό δημοψήφισμα και για το Δημοσιονομικό Σύμφωνο πρόσφατα. Ένα άλλο θέμα είναι μήπω οι πολίτε θα μπορούσαν να έχουν τη δυνατότητα να δρομολογούν οι ίδιοι ένα δημοψήφισμα. Αν δεν υπάρχουν περιορισμοί για το ερώτημα, ναι. Θυμάμαι για τη δεκαετία 50 και 60 όταν τα βασικά βρετανικά κόμματα, φαντάζομαι και στις περισσότερες δυτικές ε, χώρες θεωρούσαν ότι η μαζική μετανάστευση είναι πάρα πολύ καλή ιδέα. Ίσως τότε θα έπρεπε να είχε γίνει ένα δημοψήφισμα, αλλά μάλλον θα είχε κριθεί ακατάλληλο το ερώτημα κωδικός που σημαίνει ότι θα έδινε λάθος απάντηση στο δημοψήφισμα. Τώρα, σε ό,τι αφορά για τις δαπάνες, για το δημοσιονομικό σύμφωνο, δεν ξέρω κατά πόσο θα έπρεπε να υπάρξουν ε, δημοψηφίσματα ή ψηφοφορίες για αυτά τα δύο. Θυμάμαι κάπως ένα δημοσίευμα στην Καλιφόρνια στις ε, αρχές δεκαετίας του 80 ή τέλη ε, της ε, δεκαετίας του 70 όπου οι Καλιφορνέζοι αποφάσισαν ότι ήταν πάρα πολύ ωραία ιδέα να περιορίσουν τις, τους φόρους τους και μετά κατάλαβαν ότι δεν θα είχαν πυροσβεστική ή κάτι άλλο τι θα γίνει για τη γενική οικονομική προσέγγιση. Θα ήταν καλή ιδέα, χωρί να θέλω να παρέμβω βέβαια σε ζητήματα από αυτόν την δηλαδή, Ελλάδα, δεν είναι δική μου διάλογο. Θα ήταν πάρα πολύ καλή ιδέα να γίνει δημοψήφισμα για την πολιτική λιτότητα ε, που επιβάλλεται στην Ελλάδα. Με την υπόθεση ότι αν αυξηθεί η ανεργία και μειωθούν τα εισοδήματα των πάντων, θα μπορέσουν οι Έλληνε να βγουν από τα χρέη του πιο εύκολα. Για ένα τέτοιο δημοψήφισμα εγώ θα έφτανα ε, και στην προσχολική ηλικία για να συμμετάσχουν ακόμη και τα παιδιά προσχολικής ηλικίας στο δημοσίευμα και αυτά ακόμη θα ήξεραν τι απάντηση θα έδιναν σε αυτό. σε ευχαριστώ πολύ. Εύελιν τώρα έχει το λόγο. Ευχαριστούμε κύριε καθηγητά, κύριε Κύρχεσνερ για τις απλές παρουσιάσεις σας. Μη φοβάστε, δεν θα κάνω κι εγώ διάλεξη. Ε, μια ερώτηση έχω. Εμένα με ενδιαφέρουν οι πρακτικές εμπειρίες σας και τα συμπεράσματα με για τα εξή προβλήματα. Και στο καντόνι σας είναι απλούστερο να περάσει κανείς ε, θετικά επιχειρήματα για αύξηση φόρων ε, όταν παραδείγματο χάλη θέλει ένα καινούριο σχολείο ή μια νέα πισίνα, κάτι που θα ωφελήσει άμεσα τους πολίτες εκεί ε, όπου βλέπω εγώ τη δυσκολία, κάτι το οποίο είναι σημαντικό επίσης νομίζω, ε, τι γίνεται παραδείγματο χάρη για ετούντες άσυλο για τη χρηματοδότησή τους ή στο κοινωνικό τομέα. Πράγματα τα οποία δεν είναι πάντα απλά. Ευχαριστώ. Ο κύριος Χέφνερ και μετά εμπειρογνώμονές μας. Θα απαντήσω απλά. Είναι σαφές. Όσο πιο συγκεκριμένη η δαπάνη, τόσο πιο πιθανό είναι οι πολίτες να την υπερψηφίσουν. Είναι ενδιαφέρον παραδείγματο χάρη το ότι η αύξηση του φόρου των πετρελαιοειδών το 1993 θα πήγαινε στις υποδομές των δρόμων. Όσον αφορά τώρα την ε, πολιτική του ασύλου, έχετε δίκιο. Εκεί πέρα πράγματι υπάρχουν προβλήματα. Βεβαίως το πρόβλημα δεν είναι η χρηματοδότηση, η οποία κατά βάση είναι εθνική. Το πρόβλημα είναι πού θα χτιστούν τα κέντρα φιλοξενίας και τέτοια πράγματα. Αυτή είναι αντίσταση, αλλά δεν είναι θέμα δημοψηφισμάτων κτλ. Το ξέρουμε και σε άλλες χώρες αυτό το φαινόμενο, δεν είναι ε, έτσι καμία χώρα Αγίων και η Ελβετία. Αλλά αν δείτε παραδείγματο χάρη το τι έγινε με την αύξηση του ΦΠΑ για τη χρηματοδότηση των συντάξεων, για την αύξηση, την αύξηση του ΦΠΑ για τη χρηματοδότηση των επιδομάτων αναπήρων. Γίνεται ξεκάθαρη η συζήτηση. Αλλά τα καταφέραμε. Πέρασαν δηλαδή αυτά τα πράγματα επίμαχα. Αν γίνει η σωστή ε, εξαρτία, πείθονται οι πολίτες. Δεν πετυχαίνει πάντα δεν περνάνε όλα τα θέματα είπα όπως ε, θα ήθελα εγώ ας πούμε αλλά δεν είναι αδύνατον να ε, πείσουμε τους πολίτες και για τέτοια πράγματα. Πρέπει απλά να προσπαθήσει κανείς και αν δεν προσπαθεί ε, πάνε και τα πράγματα στραβά. Alors, Äh, Ευχαριστώ. Και εγώ θέλω να κάνω μία ερώτηση. Πρώτα απ' όλα ε, μία παρέμβαση στο ερώτημα της κυρίας Ρέντνερ. Ο λόγος για τον οποίο καλέσαμε έναν ειδικό εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα ακούσουμε και άλλους Ελβετούς μετά, ε, είναι γιατί ε, μπορούμε να μάθουμε πάρα πολλά από την Ελβετία, όχι για τη θεωρία της άμεσης δημοκρατίας, αλλά για την πράξη. Γιατί μετά τίθεται το ερώτημα, δεν είναι δύσκολο να χρηματοδοτήσουμε παραδείγματο χάρη τούντες ε, άσυλο, κοινωνικά επιδόματα από ό,τι μία πισίνα. Αλλά πέρα από ε, τα διάφορα πράγματα που είπαμε στην Ελβετία υπάρχει και η αρχαία μορφή της τοπικής ε, συνέλευσης και κοινότητας. Και το έχω δει αυτό. Κάναμε ταξίδια με ένα σύλλογο του οποίου είμαι πρόεδρος και λάβαμε μέρος σε μια τέτοια έτσι, λαϊκή συνελευτή. Γίνεται έρχεται όλος ο πληθυσμός στην πλατεία του χωριού. Αυτό γίνεται στο Απεντσέλ γιατί είναι λίγοι άνθρωποι. Και είχε συμβεί το, το εξή. Αποφάσισαν τότε οι Ελβετοί να πουλήσουν ε, ένα κομμάτι των αποθεμάτων χρυσού ε, που υπήρχαν ε, στην κεντρική τράπεζα και το ρύθμισαν ως εξής. Δεν το αποφάσισε η κυβέρνηση το τι θα κάνει τα λεφτά, αλλά οι πολίτες, οι άνθρωποι. Αποφασίστηκε στα καντόνια το τι θα γίνει και η διοίκηση του καντονιού είπε το συζητήσαμε, έχουμε τις εξής προτάσεις, και μαζεύονταν ο κόσμος στο, στο Δημαρχείο ή όπου αλλού και λέγανε ξέρω εγώ να κάνουμε το τάδε δρόμο, το τάδε κτίριο κτλ. Και έσκαν κάτι νέοι άνθρωποι και λένε ε, αυτά μπορούν να χρηματοδοτηθούν από το γενικό προϋπολογισμό. Αυτά όμως εδώ πέρα είναι η εξοικονόμηση του κόπου του λαού. Οπότε θα πρέπει να πάει σε ένα ταμείο για την στήριξη οικογενειών που έχουν ανάγκη και μονογονεϊκών οικογενειών, ε, σχολεία ξέρω εγώ, αλλά κυρίως κοινωνικές δαπάνες. Το συζήτησαν λοιπόν αυτό στην πλατεία και τελικά ε, κέρδισαν οι νέοι. Αυτοί έπεισαν τους υπόλοιπους. Αλλά έχω ένα ε, ερώτημα. Ένα προς τον κύριο Κύρκη και ένα προς τον Τέο Σίλερ προς τον κύριο Σίλερ πρώτα. Θεόδωρε. Ε, μας έδειξες αναχώρες ε, ποιες είναι οι ανάγκες μεταρρύθμισης ε, που θεωρείς εσύ ότι υπάρχουν, αλλά από ευγένεια δεν είπες τίποτα για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θέλω να θέσω αυτό το ερώτημα. Δηλαδή θεωρείς πως η άμεση δημοκρατία μπορεί να χρησιμοποιηθεί και στο επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αν ναι, τι πρέπει να προσέξουμε. τους χάρη πρέπει να απαιτούνται ειδικέ ε, πλειοψηφίε και άλλα τέτοια πράγματα. Αυτό είναι το ερώτημά μου. Ή προς τον καθηγητή ε, τον κύριο Σίλερ. Ε, ένα έτσι πονηρό ερώτημα. Έχουμε τώρα την εξής κατάσταση. Για να περιοριστούν τα χρέη των κρατών μελών υπάρχει ένα ευρωπαϊκό ταμείο σταθερότητας το οποίο διαχειρίζεται η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα κτλ. Και ταυτόχρονα σε πολλές χώρες Ευρώπης έχουμε τεράστια οργή κατά των μέτρων της πολιτικής λιτότητας που και πάλι υπαγορεύονται από πάνω από τους τεχνοκράτες. Και αυτό το οποίο ζει κανείς αν μιλήσει με τους ανθρώπους είναι πως παντού στην Ευρώπη υπάρχει η διάθεση πως αυτά τα κέρια ζητήματα, σημασία ζητήματα αποφασίζονται χωρίς να ρωτήσουν κανέναν. Ούτε στην μία χώρα, ούτε στην άλλη. Και του λένε κανείς δεν μας ρωτάει, δεν υπάρχει καμία ανοιχτή συζήτηση. λένε δεν υπάρχει εναλλακτική, εφαρμόζονται αυτά και δεν υπάρχει στήριξη των ανθρώπων. Και αν δούμε και το θέμα αυτό, δηλαδή από δημοκρατική σκοπιά, οδηγούμαστε σε κυριαρχία τεχνοκρατών και σε λιγότερη δημοκρατία. Και auf Dauer so funktioniert und ob die Eingriffs... Δεν ξέρω, μπορεί να λειτουργήσει αυτό σε βάθος χρόνου. Το ερώτημα λοιπόν είναι, Πώ μπορούμε να το σκεφτούμε αλλιώ. Στην Ελβετία, παραδείγματο χάρη, υπάρχει αυτό το όριο του χρέου, το οποίο το πέρασαν οι ίδιοι οι πολίτες. Ένα όριο στη χρέωση του κράτους που δεν ορίστηκε από πάνω και δεν το διέταξε κανείς. Οι πολίτες από μόνοι τους και εκπροσωποί τους το έθεσαν. Θα μπορούσαμε λοιπόν στην Ευρώπη να σκεφτούμε κάποιο τρόπο ε, για να λύσουμε δημοκρατικά αυτή τη λύση. Και πόσο μακροπρόθεσμα θα μπορούσε να υπάρχει μια λογική συμπεριφορά των πολιτών στην Ευρώπη για μια εξισορρόπηση ε, των χρεών. Γιατί κάποτε πρέπει να εξορροπηθούν και να μειωθούν αυτά τα χρέη. Σε ποιο μέτρο λοιπόν θα μπορούσε να υπάρξει ένας τέτοιος μηχανισμός στις ευρωπαϊκές χώρες και θα μπορούσαμε να κάνουμε μια τέτοια ανοιχτή συζήτηση γιατί χτες Ρομπέρτο θυμάσαι έθεσα εγώ το ερώτημα για τη συνέλευση και τη δημοκρατία και η απάντηση ήταν ναι αλλά όχι τώρα τώρα είμαστε στην κρίση άμα είμαστε ξανά σε καλύτερη κατάσταση, το ξαναβλέπουμε. Αλλά μήπως ακριβώς στην κρίση πρέπει να γίνει κάτι τέτοιο. Αλλιώς θα χάσουμε τη στήριξη των ανθρώπων και θα βυθιζόμαστε πιο βαθιά στην κρίση. Θέλω λοιπόν να μας πείτε, να μας προσφέρετε την εμπειρία σας που είναι εμπειρία δεκαετιών και στην πράξη. Ευχαριστώ. Uh, ευχαριστώ πολύ και ζητώ συγγνώμη γιατί χρειάστηκε να απουσιάσω από ένα μέρος της συζήτησης διότι πρέπει να είμαι στην Επιτροπή Ασφάλειας και Άμυνας γιατί προετοιμάζουμε την σχετική πολιτική άμυνας και ασφάλειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα σας ρωτήσω το εξής. Ποιος είναι ο αντίκτυπος των πειραμάτων, αν θέλετε, αυτών ή των εμπειριών που έχετε από την άμεση δημοκρατία. Θεωρώ ότι είναι προφανές ότι δεν μπορείτε να προωθήσετε εκστρατεία δημοψηφίσματος αν δεν υπάρχουν και ισχυρά πολιτικά κόμματα με οργάνωση, με χρηματοδότηση, με μήνυμα, με ηγεσία. Επίσης θεωρώ ότι η εμπειρία διδάσκει ότι τα πολιτικά κόμματα τα οποία καταφεύγουν σε δημοψηφίσματα το πράττουν συχνά ε, επειδή βρίσκονται σε θέση μεγάλης αδυναμίας. δηλαδή δεν είναι σε θέση να αντιμετωπίσουν ένα πολύπλοκο επίμαχο θέμα που απαιτεί ε, απόφαση. Και αυτό σημαίνει ότι ουσιαστικά πρέπει να επιβάλλουν την ευθύνη για τη λήψη της πολιτικής απόφασης στους φτωχούς ψηφοφόρους στους κακόμενους ψηφοφόρους. Και πολλές φορές η εμπειρία έχει διδάξει ότι διχάζονται και διαιρούνται τα πολιτικά κόμματα μετά από κάποιο δημοψήφισμα. Δηλαδή διασπάται η συνοχή τους. Μέσα σε αυτή την ε, ατμόσφαιρα ε, των τριβών του λαϊκισμού που πολλές φορές κυριαρχεί στις ε, εκστρατείες ε, διεξαγωγής δημοψηφίσματος. Επίσης, τα κοινοβούλια τα οποία επιτρέπουν τη διεξαγωγή δημοψηφίσματος αποδυναμώνονται και αυτά ως αντιπροσωπευτικοί φορείς μετά από το δημοψήφισμα ή λόγω του δημοψηφίσματος. στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχουμε ομόσπονδα πολιτικά κόμματα και υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη αντίσταση ακόμη και εδώ, ακόμη και εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τη δημιουργία ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μάλιστα μόλις δημοσίευσε ένα πάρα πολύ παράλογο σχέδιο για καταστατικό ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων που ουσιαστικά αποτρέπει, τέλος πάντων επιδιώκει να σταματήσει ε, τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα από το να διεκδικήσουν ένα συντημοψήφισμα συμμετοχή τους εκλογές για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Θα μπορούσατε λοιπόν να μας πείτε ποιος είναι ο ρόλος των πολιτικών κομμάτων σε όλα αυτά μέσα και ποιος είναι ο αντίκτυπος για αυτά, ο αντίκτυπος των δημοψηφισμάτων. Ευχαριστώ. Äh, das waren äh, eigentlich insgesamt drei Fragen. Τρεις ερωτήσεις ακούστηκαν συνολικά. Πρώτη για την οικονομική κρίση. Αν ξεκινήσουμε χρειάζεται κανένα μισάωρο για να απαντήσω σε αυτό. Σύντομα, η άμεση δημοκρατία ε, δεν μπορεί να θεραπεύσει τα όσα έγιναν τα τελευταία χρόνια. Και ξεκινάμε με το ότι η Γαλλία και η Γερμανία ε, παραβίασαν τη συνθήκη του Μάστριχτ, υπήρχε η ρήτρα μη διάσωση στη συνθήκη του Μάστριχτ που παραβιάστηκε και τώρα ε, η Ευρωζώνη ε, έχει μεγάλο πρόβλημα και αυτή τη στιγμή δεν βλέπω πώς μπορούμε να το λύσουμε καλύτερα αμεσοδημοκρατικά. Αυτό δεν σημαίνει πως δεν μπορούμε να σκεφτούμε για το μέλλον ε, ή για άλλες περιπτώσεις την εισαγωγή αμεσοδημοκρατικών στοιχείων που θα μπορούσαν να εμποδίσουν τέτοια πράγματα στο μέλλον. Αλλά δεν βοηθάει αυτό. Το ξέρουμε αυτό. Ε, το ξέρουμε αυτό από την Ελβετία πως χρειάζεται καιρός για να φανούν τα αποτελέσματα των διαδικασίων αυτών. Γιατί όταν ιδρύθηκε και το Ομοσπονδιακό κράτος στην ε, Ελβετία χρειάστηκε χρόνος, δεν υπήρχε τότε τίποτα το δημοκρατικό. Είναι μια εξελικτική διαδικασία. Δεν μπορούμε να ελπίζουμε πως ε, θα κάνουμε κάτι σήμερα π.χ. θα εισαχθεί το δημοψήφισμα και θα λυθούν αυτομάτως τα προβλήματα. Πρέπει να σκεφτούμε τι μπορούμε να κάνουμε καλύτερα στο μέλλον, αλλά η ελπίδα του ότι θα λυθεί η οικονομική κρίση με αυτό είναι φρούδα. Οπότε ε, αυτά τα οποία έχουν ήδη γίνει τα αμαρτήματα του παρελθόντος αν θέλετε δεν μπορούν να ξεγίνουν μέσω της άμεσης δημοκρατίας. Το δεύτερο ερώτημα αφορούσε τη σχέση μεταξύ άμεσης δημοκρατίας και κομμάτων. Και ε, ένα είναι ε, γεγονός πως αν υπάρχει άμεση δημοκρατία και ιδιαίτερα αν υπάρχει στη μορφή την Ελβετική ο ρόλος των κομμάτων είναι πιο περιορισμένος από ό,τι στο αντιπροσωπευτικό σύστημα γιατί υπάρχει δυνατότητα να τεθούν ζητήματα στην πολιτική ατζέντα ανεξαρτήτως από τα κόμματα και αυτό συμβαίνει και επιτυχώς. Τελευταία φορά είχαμε ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα με διάφορες ε, πρωτοβουλίες που παραβίαζαν παραδείγματο χάρη ε, την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Και η οποία όμως παρόλα αυτά ξεκίνησαν δύο γυναίκες και αποδείχθηκε επιτυχής. Είχαμε πει στη συχνή πρωτοβουλία για την κατάργηση του στρατού. Δεν είναι κόμμα και αυτό, παρά το ότι υπάρχουν κάποιες συμπάθειες, αλλά είχε κάποια ε, επιτυχία. Οπότε το γεγονός πως υπάρχουν πρωτοβουλίες ή ε, δημοψηφίσματα κάτι το ε, τα οποία αμφισβητούν πράγματα τα οποία αποφάσισαν όλα τα κόμματα παραδείγματο χάρη στο Κοινοβούλιο. σημαίνει πως το δημοψήφισμα είναι μέσω ελέγχου της κυβέρνησης του Κοινοβουλίου όταν αποφασίζουν κάτι το οποίο προφανώς δεν συμφωνεί με το κοινό αίσθημα με την πλειοψηφία του λαού. Και ακριβώς εδώ πέρα υπάρχει ένα περιθώριο, αν θέλετε, ελιγμών, το οποίο δεν είναι ε, έξω κοινοβουλευτικό. Ξεκινάμε δηλαδή κάποια πράγματα και ελπίζουμε με κάποιο τρόπο να επηρεάσουμε το κοινοβούλιο, αλλά ε, έχουμε ένα σύνταγμα το οποίο θεσμοποιεί αυτή τη διαδικασία και δίνει δυνατότητα επηρεασμού της πολιτικής ατζέντας. Π.χ. στην Ελβετία έχουμε αυτή τη στιγμή ένα μορατόριο για μια απόφαση για την κατάργηση των ε, πυρηνικών σταθμών. Και αυτό, ε, αυτή η απόφαση ελήφθη όταν δεν είχαν σκεφτεί καν στη Γερμανία και σε άλλες χώρες πως είναι κάτι το επικίνδυνο. Αυτό το σκέφτηκαν στη Γερμανία και ετέθη ως ζήτημα με τους πράσινους κτλ. Ήταν πολύ αργότερα αυτό γιατί τότε όλα τα μεγάλα κόμματα της Γερμανίας ήταν υπέρ. Εμείς ε, είχαμε ψηφίσει ήδη επ' αυτού στην Ελβετία. Οπότε εδώ πέρα υπάρχει, υπάρχουν νέες δυνατότητες. Κάτι ακόμα. Βεβαίως μπορεί κάποιος να πει πως στο δημοψήφισμα μπορεί να ψηφίσει κανείς μόνο ναι ή όχι. και όταν μιλάμε βέβαια για κοινοβουλευτική συζήτηση κτλ. Εντάξει, είναι διαφορετική η κατάσταση. Σωστό, αλλά και το κοινοβούλιο στην τελική ψηφοφορία, ναι ή όχι θα πει. Και το δημοψήφισμα δεν διαφέρει. Τι είναι, είναι μια επιπλέον πλειο... Ε, ψηφοφορία μετά από την τελική ψηφοφορία στο ε, Κοινοβούλιο. Και τα σκέφτονται πολύ σοβαρότερα τα πράγματα στο Κοινοβούλιο όταν ξέρουν πώς θα ακολουθήσει δημοψήφισμα. Ενώ το δημοψήφισμα το εκμεταλλεύονται συχνά και τα κόμματα εκείνα τα οποία έχασαν στο Κοινοβούλιο. Δηλαδή λένε ότι χάσαμε στο Κοινοβούλιο αλλά μπορεί ο λαό να μας ε, στηρίξει. Στη Γερμανία παραδείγματο χάρη πάνε στο συνταγματικό δικαστήριο. Νομίζω πως είναι καλύτερο να ρωτάμε το λαό για τέτοια πολιτικά ζητήματα. Ευχαριστούμε κύριο Σίλερ. Σα äh, äh, Σας ευχαριστώ για τις ερωτήσεις και τις παρατηρήσεις σας για το βασικό ζήτημα του Γκέλ Χεφνερ για το ευρωπαϊκό επίπεδο να δώσω δύο πληροφορίες ακόμα πρώτον μόλις μου ανακοίνωσαν πως η Φιλανδία κατά τη διάρκεια του έτους έλαβε μια πρωτοβουλία πολιτών αλλά δεν, δεν είμαι σίγουρος για το αποτέλεσμα. Εν πάση περιπτώσει κάτι κυμα, κινείται σε αυτήν την κατεύθυνση και η Σουηδία κάτι έκανε ανάλογο τα τέλη του προηγούμενου τους και αυτό είναι κάτι το καινούριο. Επίσης, ε, κάτι το οποίο αναφέρθηκε η Καλιφόρνια, Το 1935 η Καλιφόρνια με την τότε κρίση ε, είχε περάσει ένα όριο χρέους αλλά με έναν ιδιαίτερο τρόπο. Δηλαδή, τι γίνεται, για κάθε προϋπολογισμό στην Καλιφόρνια έκτοτε απαιτείται πλειοψηφία δύο τρίτων στο ε, Κογκρέσο της ε, Καλιφόρνιας. Αυτό είναι βασική αιτία. Δηλαδή απαιτείται συνένεση, αλλά ακριβώς εδώ πέρα αποδείχθηκε η αδυναμία λειτουργίας. Και το 76-77 που υπήρξε ε, αυτόματη τεράστια αύξηση των φόρων και δεν μπόρεσαν τα κόμματα να την αντισταθμίσουν, τότε ε, δημιουργήθηκε αυτός ο αρνητικός μύθος πως λόγω της άμεσης δημοκρατίας δεν μπορεί να κουμαντάρει τα οικονομικά της. Όχι. Πρέπει εδώ πέρα να δούμε τη συνολική εικόνα. Και να προσέχουμε τι λέμε. Η Καλιφόρνια δεν είναι στην κατάσταση που έχει φτάσει Ε, για τον λόγο που νομίζουμε, αλλά γιατί δεν μπορεί να καταργήσει τον κανόνα των δύο τρίτων. Αυτό είναι το ζήτημα. Τώρα για το ζήτημα της άμεσης δημοκρατίας στο ευρωπαϊκό επίπεδο. Δεν το παρέλειψα λόγω ευγένειας, αλλά για λόγους ε, χρόνου. Κοιτάξτε. Ε... Εδώ πέρα η Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών μπορεί να αποτελέσει μόνο μία αρχή. Εγώ θεωρώ πως ε, μπορούμε να μάθουμε από την Ελβετία το πως το 1874 ε, εισήχθη τότε το προαιρετικό δημοψήφισμα, δηλαδή η δυνατότητα των πολιτών να καταρρίψουν έναν νόμο ο οποίος είχε ψηφιστεί και να μην ισχύσει αυτός ποτέ. Θεωρώ πως στο ευρωπαϊκό επίπεδο η εισαγωγή ενός τέτοιου δημοψηφίσματος από τους πολίτες δηλαδή απέναντι σε έναν νόμο ο οποίος έχει εγκριθεί αλλά ακόμα δεν έχει τεθεί νομίζω ε, πως θα είναι κάτι το πάρα πολύ σημαντικό. Αφενός για αποφάσεις οι οποίες ε, προκύπτουν από το ευρωπαϊκό σύστημα αποφάσεων, θα έλεγα αυτή της δευτερογενούς δημοκρατίας, για να υπάρχει αν θέλετε μια δοκιμή, ένα τεστ αποδοχής, κάτι το οποίο δεν είναι δυνατόν αυτή τη στιγμή. Μόνο κάποια ισχυρά μήνυε έχουν την δυνατότητα να επηρεάσουν και να επιτεθούν σε μια απόφαση των Βρυξελών για να προξενήσουν μια νέα συζήτηση, αλλά για τους πολίτες είναι αδύνατον. Ή μια μεγάλη ομάδα συμφερόντων, όπως ε, π.χ. Αλλά αυτό γίνεται και για την Ομοθεσία ήδη από πριν. Ξέρουμε πόσες χιλιάδες λομπίστες ε, δραστηριοποιούνται εδώ στις Βρυξέλλες. Και μια τέτοια δυνατότητα να αμφισβητηθεί αυτή η διαδικασία νομίζω θα αποτελούσε μια σημαντική διαδικασία ελέγχου. Αλλά από την άλλη θεωρώ πως η αμφισβήτηση ε, ενός τέτοιου νόμου θα δημιουργούσε μια τεράστια δημόσια συζήτηση στις ευρωπαϊκές χώρες και θα καθιστούσε αναγκαίο για τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα, την Κομισιόν, αλλά και τις κυβερνήσεις, ε, τους υπουργούς του Συμβουλίου, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, να αιτιολογήσουν αυτές τις αποφάσεις σε έναν διάλογο που θα προκύψει μετά σε ένα ευρωπαϊκό κοινό, σε μια ευρωπαϊκή κοινή γνώμη. Και εδώ πέρα μπορεί να υπάρξει μια σύνδεση με αυτό το οποίο αναφέρθηκε για τον ρόλο των, κομμάτων και την επιρροή των κομμάτων. Θεωρώ πως με τη χρήση αυτού του μέσου και τα κόμματα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα είχαν την πρόκληση ενώπιόν τους να τοποθετηθούν και να δικαιολογήσουν την απόφασή τους. Οπότε σε ένα πολιτικό σύστημα στο οποίο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υποφέρει από το ότι δεν υπάρχει κυβέρνηση και αντιπολίτευση ε, στο πλαίσιο των εκλογών και μια τέτοια θεαματική νομοποίηση, αλλά έχουμε κάποιες εκλογές δεύτερης κατηγορίας θα έλεγα με τη μισή συμμετοχή από τις εθνικές εκλογές και έχουμε μια ισχνή νομιμοποίηση ε, τότε και τα κόμματα θα είχαν τελείως διαφορετική λειτουργία και μια ευκαιρία να συζητήσουν για τις πολιτικές αποφάσεις ε, της Ευρώπης. Βεβαίως δεν είμαι καθόλου κατά της χρήσης ε, του μέσου αυτού της ε, πρωτοβουλίας ε, πολιτών και της διεύρυνσης της χρήσης αυτής για να πάμε σε ένα πλήρες δικαίωμα πρωτοβουλίας με ψηφοφορίες αλλά η σειρά ίσως η ακολουθία πιο εφικτή θα είναι μέσω των ε, δημοψήφισμάτων θα έλεγα. για την ε, διαφοροποίηση τώρα ε, που πρέπει να γίνει. Πρέπει να γίνει μια διάκριση όταν μιλάμε για Ευρώπη και δημοψηφίσματα. Μιλάμε για μεγάλα συνταγματικά ζητήματα ή τις συνθήκες, αλλά δεν μιλάμε για ζητήματα πολιτικής. Για τις απλές, τα, τα φυσιολογικά θα έλεγα ζητήματα πολιτικής. Και ε, τι γίνεται. Όταν ακριβώς συζητιούνται τα μεγάλα συνταγματικά ζητήματα και σκέφτεται ο κόσμος ένα δημοψήφισμα, τι γίνεται. Τίθεται το ζήτημα του εάν για πρώτη φορά οι πολίτες ε, θα πρέπει να βρεθούν ενώπιον μία τέτοιας συνθήκης, όπως έγινε στην Ολλανδία. Αυτό ήταν το πρώτο δημοψήφισμα που έγινε στην Ολλανδία γενικώ. Και όταν η κυβέρνηση δεν είναι και υπέρ, δεν απορεί κανείς ε, για το ότι χάθηκε η ψηφοφορία, αλλά η σημασία της άμεσης δημοκρατίας στο ευρωπαϊκό επίπεδο δεν ε, θα εξελιχθεί κυρίως με τα συνταγματικά ζητήματα, αλλά με τις φυσιολογικές εντό εισαγωγικών πολιτικές αποφάσεις. Γι' αυτό αναφέρθηκα στην κατάσταση στα κράτη-μέλη, γιατί το ζήτημα εκεί πέρα δεν αφορά μόνο συνταγματικά ζητήματα, τα οποία εντάξει είναι οπωσδήποτε σημαντικά, τα σημαντικότερα, αλλά μόνο σε μια τακτική και θεσμοποιημένη πράξη και πρακτική ε, που θα οδηγήσει σε μια δημοκρατική κουλτούρα μπορούμε να ε, θεωρήσουμε πως έχουμε μια βάση δημοκρατικής κουλτούρας και ε, πολιτική συμμετοχή στο ευρωπαϊκό επίπεδο. Τελευταία σύντομη παρατήρηση για αυτά τα οποία είπε ο κύριος Ντάφ. Επιρροή στα κόμματα. Εδώ πέρα υπάρχει μία συζήτηση μεταξύ των επιστημόνων για το μήπως τα κόμματα κυριαρχούν στα ζητήματα δημοψηφίσματος και είναι άρα άλλη μία μορφή διαμάχης που μεταφέρεται σε άλλο επίπεδο. Δεν το βλέπω εγώ έτσι. Έχουμε αναφερθεί στο εάν τα δημοψίσματα μπορούν να οδηγήσουν σε διχασμό και διάσπαση κομμάτων. Υπάρχει και η αντίστοιχη εμπειρία. Είναι διχασμένα τα κόμματα και τι κάνουν. Ξεκινάνε ένα δημοψήφισμα για να ε, απαντηθεί το ερώτημα. Οπότε πάει και προς δύο κατευθύνσεις αυτό. Και νομίζω πως μπορούμε να δούμε και την εμπειρία πως τα κόμματα σε ένα περιβάλλον άμεσο δημοκρατικών διαδικασιών ενισχύονται γιατί υπάρχει η πρόκληση του να διατυπώσουν καλύτερα την πολιτική τους, να είναι πιο κατανοητοί, να την υπερασπιστούν, να ζυγίσουν τα επιχειρήματα και έτσι αναπτύσσονται τα κόμματα. Τα κόμματα συχνά είναι ασθενή γιατί χάνουν την επαφή με τους πολίτες και τέλος μια παρατήρηση για την τρέχουσα οικονομική κρίση. Αυτό το οποίο ζούμε δεν είναι μόνο γενικά μια απώλεια εμπιστοσύνης των πολιτών στην ε, ικανότητα λήψη αποφάσεων των αντιπροσωπευτικών θεσμικών οργάνων της Ευρώπης και των κρατών μελών, αλλά είναι απώλεια εμπιστοσύνης στην ικανότητα των θεσμικών οργάνων. που ακριβώς ζητάνε και απαιτούν αυτή την εξουσία για λόγους τεχνοκρατικούς, αλλά δεν αποδείχθηκαν ικανοί να αποτρέψουν την κρίση. Οπότε αναρωτιέμαι πού ήταν αυτή η ικανότητα των Ισπανικών τραπεζών για να αποφύγουν τη φούσκα των ακινήτων. Εντάξει, υπάρχει το κίνητρο του κέρδους για όλες τις τράπεζες, αλλά αυτό ισχύει γενικώ για ολόκληρη την, ε, για ολόκληρη την νομιμοποίηση των τεχνοκρατών που βασίζεται όπως είπαμε στο αποτέλεσμα το οποίο όμως προφανώς δεν ε, υφίσταται και δεν ε, καλύπτεται από την νομοποίηση τη αντιπροσωπευτική δημοκρατία. Σε αυτό το πλαίσιο μιλάμε για την άμεση δημοκρατία ω αναζωογόνηση τη δημοκρατία. Έχουμε μόνο πέντε λεπτά ακόμη, αλλά έχει ζητήσει το λόγο ο κύριος Γιέργεν. Θα του δώσω το λόγο. Σα ευχαριστώ για την ευκαιρία. Το ερώτημά μου απευθύνει στον κύριο Κύρκιασνα και αφορά το εξής. Ε, αναφερθήκατε στο εάν υπάρχει ευρωπαϊκή αλληλεγγύη, αν υπάρχει δυνατότητα να... Ε, δεν το είπατε εσείς έτσι, αλλά αυτό είναι το υπόβαθρο. Ότι οι Γερμανοί πρέπει να πληρώσουν ε, κάτι, αλλά να δουν τι βγάζουν από αυτό. Δηλαδή και οι Έλληνες πρέπει να ανταποκριθούν στις, στους όρους. Οπότε το ερώτημα είναι... Εκεί πέρα ο Πέτερ Σνάιντερ έγραψε μια πολύ ωραία επιφυλίδα που λέει πως η Ευρώπη θα πρέπει είτε να ελβετοποιηθεί είτε θα διαλυθεί. Σε αυτό λοιπόν το θαυμάσιο ελβετικό αμεσοδημοκρατικό παράδειγμα υπάρχει κάποιο παράδειγμα για τους για την βοήθεια ας πούμε στους γείτονες και στα συμφέροντα των γειτόνων Δηλαδή υπάρχει κάποιο παράδειγμα στο οποίο οι Ελβετοί είπαν πρέπει να λάβουμε υπόψη τα συμφέροντα και των διπλανών μας. Ε, κάτι τέτοιο θα μας ενθάρρυνε. Ε, απάντηση. Οπωσδήποτε, κοιτάξτε, δεν θα παραβιάσουμε τους, τους νόμους μας ε, γι' αυτό. Δύο πράγματα. Κοιτάξτε. Υπάρχει βεβαίως πολύ μεγαλύτερη οικονομική αλληλεγγύη, αλλά αμφιβάλλω για το εάν η Ευρώπη έχει φτάσει στο σημείο για μια ευρωπαϊκή οικονομική αλληλεγγύη. Υπάρχει το περιφερειακό ταμείο, δεν ξέρω αν μπορεί να επεκταθεί σε τέτοιο βαθμό. Η Ελβετία έφτιαξε ομοσπονδιακό κράτος το 1848, οπότε η αλληλεγγύη μεταξύ των καντονίων ήρθε πολύ αργά. Το εάν μπορούν τέτοια πράγματα δηλαδή έτσι απλά να μεταφερθούν σε τελείως διαφορετικές άλλες μορφές και δομές είναι ένα ερώτημα. Ε, τώρα στις μεθοριακές περιοχές είτε στο Μπόντεντζε είτε στη Βασιλεία Μιλούς και τα λοιπά έχουμε πολύ καλές σχέσεις με τα διπλανά γειτονικά κράτη και κρατήδια αν θέλετε και Φόραλμπεργκ εκεί πέρα και ε, στη γειτονιά μας δηλαδή το κάνουμε αυτό οπωσδήποτε. Στο πλαίσιο του συντάγματος πάντα. Επιπλέον, η Ελβετία σε πολλούς τομείς δραστηριοποιείται ε, διεθνώς ε, σε τομείς όπου δεν δραστηριοποιούνται άλλα κράτη. Οπότε Είμαι επιφυλακτικός για το εάν θα μπορούσε η Ευρώπη σύντομα να κάνει κάτι τέτοιο ανάλογο με αυτό το οποίο σημαίνει στο ελβετικό κράτος γιατί η Ευρώπη ακόμα πρέπει να αναπτυχθεί σε ψυχολογικό επίπεδο από κοινού. Δηλαδή δεν μπορούμε να μιλάμε για Ευρωπαϊκό Δήμο ακόμα. Πρέπει να υπάρχουν κάποια πράγματα, κάποιε υποθέσεις πριν προχωρήσουμε σε αυτό το, το βήμα. Τώρα για τα γερμανικά ερωτήματα του εάν πρέπει να υποστηριχθεί η Ελλάδα, η συντριπτική πλειοψηφία είναι κατά και νομίζω και στι υπόλοιπε χώρες έτσι είναι η κατάσταση. Οπότε, δεν, κατά την άποψή μου πάντα, δεν νομίζω πως έχει φτάσει στο σημείο να κάνει αυτό το βήμα. Ο συμπρόεδρος θέλει να παρέμβει. Ήταν πολύ ενδιαφέρουσα η συζήτηση, δεν ήταν το τέλος, αλλά η αρχή ε, μιας ενδιαφέρουσας συζήτησης. Η Γερμανία τώρα και η Ελβετία είναι γείτονε και το συναρπαστικό βεβαίω στην Ευρώπη είναι η πάρα πολύ μεγάλη ποικιλία. Δεν είμαστε όλοι οι ίδιοι. Διαφέρουμε. Παραδείγματο χάρη, η Ελβετή είναι πολύ πιο σεμνή, σεμνή από τους ε, Γερμανούς. Ε, εσείς λέτε πράγματι πως ε, δεν μπορείτε να θεωρήσετε πρότυπο αυτό το οποίο συμβαίνει στην Ελβετία. Εντάξει, ναι, γιατί πράγματι είναι ένα εθνικό κράτος η Ελβετία, αλλά το να απαντήσουμε ένα απλό όχι θα ήταν λάθος. Εμείς θα μπορούσαμε να μάθουμε κάποια πράγματα από σας. από τις ε, εμπειρικές σας έρευνες ε, ε, στη δεκαετία του 80 και του 90 μπορούμε να μάθουμε και διδασκόμαστε πως έχει τεράστια διαφορά το να συμμετέχει κανείς σε μία απόφαση ή όχι και αυτό το ξέρουμε και από τη ζωή μας. Αν μου λένε πως αυτό πρέπει να κάνεις και αυτό απαγορεύεται και εγώ οργίζομαι. Αν όμως συμμετέχω και εγώ στην απόφαση, είναι αλλιώς τα πράγματα. Εάν το κράτος απλά ζητάει λεφτά και φόρους από τους πολίτες και οι πολίτες δεν συμμετέχουν στη λήψη αποφάσεων, η λογική είναι πώς, πώς δεν θα μου πάρουν τα λεφτά. Δεν θα τους τα δώσω. Αν γίνει όμως μια συζήτηση όπως στην Ελβετία πρέπει να χρηματοδοτήσουμε την κοινή μας ύπαρξη είναι μια κοινή απόφαση και βεβαίως έχετε δίκιο όταν στατικά βλέποντας τη σημερινή κατάσταση λέτε πως δεν είναι διατεθειμένοι οι Γερμανοί να δώσουν κάτι στην Ελλάδα αυτό ακριβώς είναι το, το μοιραίο, αυτό το οποίο πρέπει να μας απασχολήσει. Υπάρχει οργή στη Γερμανία γιατί λένε δεν μας ρωτάνε, μας παίρνουν τα λεφτά και τα δίνουν Και στην Ελλάδα λένε Αντιστρόφως δεν υπάρχει και καμία ευγνωμοσύνη, αλλά οργή για τις ε, οικονομίες οι οποίες γίνονται. Και λένε αυτοί εκεί πάνω τι αποφασίζουν, όλα αυτά είναι λάθος. Οπότε δεν είναι τόσο απλό να λυθούν αυτοί οι κόμποι και να λέμε εσείς εκεί πάνω λάβετε καλύτερες αποφάσεις. Όχι, οι άνθρωποι οι ίδιοι πρέπει να εμπλακούν στο πρόβλημα, να δούμε ποιοι τρόποι υπάρχουν και τότε νομίζω μεσοπρόθεσμα θα υπάρξει κάτι τέτοιο, ένα είδος ευρωπαϊκής οικονομικής ε, αλληλεγγύης αν θέλετε. Τελείως διαφορετικό από αυτό το οποίο υπάρχει στην Ελβετία και στη Γερμανία σήμερα. Και εδώ πέρα είναι το ζήτημα του εάν μπορεί να υπάρξει μια συζήτηση, μια διαδικασία στην οποία ο κόσμος θα θεωρήσει ότι συμμετείχε ή απλά ότι λαμβάνει διαταγές. Αυτό νομίζω προσπαθήσαμε να δούμε σήμερα. Δηλαδή, τι μπορούμε να έχουμε ως νέα μέσα α, ως οικονομική διακυβέρνηση. Πώς μπορεί να γίνει αυτό ε, δημοκρατικά και όχι τεχνοκρατικά. Αυτό νομίζω θα μπορούσε να μας βοηθήσει και να πω ακόμα, ε, δεν το θεωρώ συμπτωματικό πως η Ελβετία κατάφερε να δημιουργήσει αυτή την ιδιαίτερη ταυτότητά της, ενώ είναι τόσοι, τόσοι διαφορετικοί άνθρωποι με τέσσερις διαφορετικές γλώσσες. Στην Ευρώπη βεβαίω έχουμε 23 ε, διαφορετικές γλώσσες. Το ζήτημα λοιπόν είναι η ταυτότητα. Οι Ελβετοί συζητάνε συνεχώς μεταξύ τους μέσω δημοψηφισμάτων, μέσω πρωτοβουλειών, τι θέμε να κάνουμε έτσι και αυτό δημιουργεί ταυτότητα. Μας μένουν λίγα δευτερόλεπτα, αλλά πρέπει να δώσω και πάλι το λόγο στους καθηγητές μας, ε, ιδίως τον κύριο από την Ελβετία. Ένα πράγμα να πω. Ε, τώρα μου ήρθε, ακούγοντα τον κύριο Γιώργες. Ψηφίσαμε στην Ελβετία για να δώσουμε ένα δισεκατομμύριο, να πληρώσουμε ένα δισεκατομμύριο στο Ταμείο Συνοχής της Ένωσης για τη διεύρυνση. Δηλαδή υπάρχουν παραδείγματα τα οποία σκεφτόμαστε όχι μόνο την άμεση γειτονιά μας αλλά και παραπέρα και δίνουμε λεφτά. Ευχαριστούμε την Ελβετία. Θα χρειαστούμε και άλλες ενισφορές και δωρεάν αν γίνεται. Κλείνουμε τώρα την πρωινή φάση της ακρόαση. Ευχαριστώ όλους τους συμμετέχοντες, ιδίω του συζήτητε. Το απόγευμα θα με αντικαταστήσει η κυρία Γκουρμάη στην Προεδρία, διότι δυστυχώς έχω ηλυμένε υποχρεώσει. Και ευχαριστώ όλους τους εμπειρογνώμονε που μας μίλησαν και αυτούς που θα μας μιλήσουν το απόγευμα.